Okay. Where are colleagues? Πού είναι οι συνάδελφοι? Ναι, πάντα εμείς οι δυο θα είμαστε, μου φαίνεται εδώ. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει κατά δύο λεπτά την έναρξη της συνεδρίασης. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά τις αποφάσεις σας. Ελπίσουμε ότι μεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση αφού οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ έγκαιρα. Η υιοθέτηση του ημερήσια διαταξή για τον Ιούνιο και οι ανησυχίε ε, των ομάδων για τι μεταγενέστερε ατζέντε ε, τα εξετάσαμε. Τα δύο αιτήματα του ΕΛΚ θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη Καθώ και η αναφορά 0720 για τι ε, γυναίκε Αραμπή που κρατούνται στην Νιγηρία. Για τι εκθέσει και τι γνωμοδοτήσεις αποφασίσαμε να μην υιοθετήσουμε νέε γνωμοδοτήσει για τις προσβαλλόμενες συστάσεις 0004 θα διατηρηθεί ανοιχτά, ανοιχτή η 0017 και η 0022 φετινές θα τις εξετάσουμε από κοινού θα διατηρηθούν ανοιχτές και οι υπόλοιπε από τις προσβαλλόμενες ε, αναφορές ε, υιοθετήθηκαν με την μορφή που πρότεινε η Πρόεδρος όσον αφορά τα σημεία η 706 του 2016 θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά 1562 επίσης θα παραμείνει ανοιχτή και θα δοθεί στον αναφερόμενο ε, διάστημα δύο μηνών επιπλέον για να απαντήσει στην απάντηση της Επιτροπής. Για τις διερευνητικές επισκέψεις ε, όρισαν τις ημερομηνίες οι συντονιστές ως εξής 19 με 21 Σεπτεμβρίου για το Ντονάνα στην Ισπανία και 29 με 31 Οκτωβρίου για το Βαλεντόρα στην Ιταλία ονόματα μελών που ενδιαφέρονται θα πρέπει να σταλούν στη γραμματεία μέχρι την 5η Ιουνίου. Αυτό δίνει αρκετό χρόνο στις ομάδες ε, για να τα εξετάσουν. Ο διαρθρωμένος διάλογος που έλαβε χώρα πρόσφατα ε, ψηφίστηκαν τα βασικά μηνύματα, εστάλησαν στην CCC. Είναι λίγο περίεργο που το λέω αυτό γιατί στέλνονται ουσιαστικά σε μένα ως πρόεδρο της CCC. Ε, Οπότε τώρα ξέρω τι θα βρω μπροστά μου. Πιθανές προφορικές ερωτήσεις για τα δικαιώματα ψήφου. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα προφορικό ερώτημα για τα ζητήματα της πύλης της ΠΕΤΗ. Οι εργασίες ε, προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο και οι συντονιστές θα διατηρηθούν ενήμεροι σε όλη τη διαδικασία. Αποφασίσαμε επιπλέον να διοργανώσουμε μια κοινή διακοινοβουλευτική συνάντηση με τη Γιούρη, με την υποστήριξη των νομικών υπηρεσιών και σε συνεργασία με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Η συνεδρίαση, η Επιτροπή αυτή θα προτιμούσε να διεξαχθεί τον Νοέμβριο, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, και εγώ θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ με την Γιούρη και τις νομικές υπηρεσίες, ώστε πράγματι να γίνει τον Νοέμβριο φέτος. Διότι οι συντονιστέ θεώρησαν το ότι το να την κάνουμε το Φεβρουάριο με επικείμενε τι εκλογέ δεν ήταν και η καλύτερη λύση. Η επιστολή της ΕΜΠΛ όσον αφορά το προφορικό μας ερώτημα και ψήφισμα για την ε, αναφορά για την καταπολέμηση ε, των αβέβαιων συμβάσεων εργασίας και της καταχρηστικής χρήσης των συμβάσεων εργασίας ε, ορισμένου χρόνου. Εγώ ήθελα να απαντήσω ε, στην επιστολή λέγοντας ότι η Επιτροπή μας και ε, οι διαδικασίες μας ε, έχουν με κάποιο τρόπο που αυτό δεν γίνεται, όπως θα το εξηγήσω επίσημα σε μια επιστολή. Περαιτέρω κάποια ενημερωτικά σημεία ακούσαμε, τα σημείωσαν οι συντονιστές, αυτά ήταν όλα. Τώρα ας πάμε πίσω για να δούμε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο, ένα πανέμορφο μέρος της Ευρώπης, πρέπει να πω. Εκεί είχαμε εμεί την διερευνητική επίσκεψη, επίσκεψη μελέτη στην Αμόχωστο και θα ήθελα να αναφέρω πολύ σύντομα ότι η αντιπροσωπεία είχε εμένα, τον Αλμπέρτο Τσίριο, ε, Φεραγκούτη, τη Σοφία Σακοράφα, Άντζελα Βαλίνα και η Γκορ Σόλτες ως ε, τακτικά μέλη και τρεις, τρία μέλη, εξοφίτσιο ε, Δημήτρης Παπαδάκης, ε, Τερέσα και Χτάκης Χατζηγεωργίου. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η αποστόλη, η αντιπροσωπεία μας αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι Πράγματι συμμεριζόμασταν όλα τα συναισθήματα και όλες τις απόψεις ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού. Τη Δευτέρα συναντήσαμε τους αναφερόμενους δικαινοτικές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τον ε, Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώστου στους χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Το βράδυ είχαμε ένα δείπνο από τον πρόεδρο της Βουλής, ε, τον κ. Δημήτρη Ξυλούρη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, και με τον Αλέξη Γαλανό τον δήμαρχο της Αμοχώστου. του. Επίσης συναντηθήκαμε με τον ειδικό εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της αποστολής των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και μετά πήγαμε στην Αμόχωστο για να δούμε το αποκομμένο κομμάτι της Βαρόσα και τις προσπελάσιμες περιοχές, προσπελάσιμες παρότι είναι δύσκολο να τις προσπελάσει κανείς, συμπερέλαβε και μία επίσκεψη στην παραλία που ονομάζεται Γλώσσα. Εκεί είχαμε μια ε, συνέντευξη τύπου με τον δήμαρχο της Αμοχώστου αργότερα στο πολιτιστικό κέντρο της ε, Αμοχώστου η κυρία που είναι επίσης κοντά και έτσι ολοκληρώθηκε το επίσημο κομμάτι της επίσκεψης. Λοιπόν, παρά την υψηλή συναισθηματική φόρτιση ε, του αναφερομένου και με τη συνάντηση μπροστά στο σπίτι όπου μεγάλωσε και από το οποίο, το οποίο χρειάστηκε να εγκαταλείψει με τη βία και με δύο γενιές πρώην ε, κατοίκων που έκλεγαν ε, εκλυπαρώντας να τους βοηθήσουμε να γυρίσουν στα σπίτια τους ε, δεν μπορεί να κάνει και πολλά το κοινοβούλιο αυτό πέραν του τελευταίου ψηφίσματος του Ιουλίου του 2017 και εγώ προσπάθησα να το επαναλαμβάνω σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε οποιαδήποτε πρόοδο στη διαδικασία αφού η διεθνή κοινότητα έχει αποτύχει εδώ και 44 χρόνια όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και όλοι οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Αλλά αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι να διατηρήσουμε ζωντανό το ζήτημα. Αυτό το δήλωσα εγώ επανειλημμένος. Αποφασίσαμε να μην επιδιώξουμε οποιαδήποτε επαφή με την ε, τουρκοκυπριακή πλευρά. Εστιαστήκαμε αποκλειστικά στο ζήτημα της αμοχώστου βάσει της αναφοράς που είχαμε λάβει. Δεν ασχοληθήκαμε με το κυπριακό ζήτημα γενικότερα. Μια συνολική διευθέτηση θα ήταν αυτό βέβαια που θα επιθυμούσαν όλοι. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις για τέτοια διευθέτηση έχουν καταλήξει σε απόλυτο αδιέξοδο μετά από το κλείσιμο χωρίς καμία συμφωνία της ε, διασκέψης στο Κραν Μοντανά το 2017 στην Ελβετία που είχε οργανωθεί από τα Ηνωμένα Εθνή. Ωστόσο, οι γενιές εξελίσσονται, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Έχουν πέρασει 44 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή και έτσι αποφασίσαμε εμείς ως αντιπροσωπεία να παρακολουθούμε στενά τα τεκτενόμενα. Θεωρούμε ότι ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία αυτή ε, να πάμε σε αυτή την επίσκεψη μελέτη. Ε, η κάλυψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση ήταν καταπληκτική. Ακόμη και στι Ηνωμένε Πολιτείε μα μετέδωσαν και ο κόσμο το εκτίμησε ιδιαίτερα το ότι προσπαθήσαμε να ρίξουμε φως σε αυτό το θέμα ότι υπάρχει μια πόλη σφραγισμένη εν μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι υπάρχει μια πόλη χωρισμένη στα δύο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ε, κάτοικοι με νόμιμο δικαίωμα διαμονής απαγορεύεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πρέπει λοιπόν να το διατηρήσουμε αυτό στο νου μας, να πούμε ότι η κατοχή που πλέον έχει διαρκέσει 44 χρόνια πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρεθεί μια πολιτισμένη λύση εποφελής ε, για τους ε, ντόπιου ανθρώπους, για τις χώρες, για τις ενδιαφέρομενες χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσω εδώ. Απλά έκανα μια αναφορά των όσων συνέβησαν. Ε, θα μιλήσω λίγο προσωπικά τώρα. Σπάνια αισθάνομαι ότι η Επιτροπή μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Αφήνει τέτοιο ίχνος στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Το πετύχαμε αυτό και είμαι ιδιαίτερα περήφανη ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής που αναλάβαμε αυτή την αποστολή και που καταφέραμε να δώσουμε έστω και λίγη ελπίδα και συμπόνια στους ανθρώπους της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Τάκη, θέλατε να μιλήσετε. Ναι, ήθελα να πω, ε, θα συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Ε, απλά ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τις προσπάθειές σας και για όλα όσα κάναμε στην Κύπρο. Ε, προσβλέπω στη συζήτηση. Ελπίζω να γίνει κάποια συζήτηση το συντομότερο δυνατόν. Βεβαίω θα γίνει. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και όλους όσοι ήταν παρόντες ήταν μια καλή στιγμή όπου δείξαμε ότι στεκόμαστε ενωμένοι και ενωμένοι πέφτουμε. Ευχαριστώ πολύ για το εκπληκτικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας. 718 on harm Πάμε στην ε, αναφορά 718. ο αναφέρον ο κ. Γκαρθία Παλαθιός Αλβάρες αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας. Σας δίνω πέντε λεπτά. Μπορείτε να τα μοιραστείτε ή ο ένας από εσά μπορεί να μιλήσει για ολόκληρο το λεπτό Όχι παραπάνω όμως. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα σχέδιο υδατοκαλλιέργειας, το οποίο προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε το 2004. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην καλλιέργεια μαλακόστρακων γλυκού νερού. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ είχε πάρει όλες τις απαραίτητες άδειε προκειμένου να καταρτιστεί η εταιρεία, προκειμένου να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί. Ζητήσαμε μάλιστα και επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίθηκε και στα πλαίσια αυτού προβλεπόταν ότι μαλακόστρακα από την Αυστραλία, καθώς επίσης και άλλα είδη καρκινοειδών, θα καλλιεργούνταν στην Ισπανία, ότι τα μαλακόστρακα αυτά θα προέρχονταν από την Αυστραλία. Αυτή ήταν η βασική χώρα, αν θέλετε, προέλευση των ειδών που εμείς θα καλλιεργούσαμε εν συνεχεία στην Ισπανία. Πήραμε λοιπόν την άδεια προκειμένου να κάνουμε αυτή την υδατοκαλλιέργεια, δημιουργήσαμε και την απαραίτητη υποδομή και έπειτα το 2005 και αργότερα το 2008 υποβάλαμε εκθέσεις προς αρμόδιες αρχές, δείχνοντας ότι ουσιαστικά ακολουθούσαμε το αρχικό σχέδιο, ότι είχαμε αναλάβει τις αρχικές μας ευθύνες. 867.000 ευρώ μας δόθηκαν ως επιδότηση και οι πληρωμές έλαβαν χώρα το 2008 και το 2010 αφού βέβαια προσκομίσαμε τα δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, τον Ιούλιο του 2009, αρχίσαμε να λειτουργούμε 100%. Και ξαφνικά, εκείνη την εποχή, μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαμε να εισάγουμε τα ίδια, αυτή, τα ίδια αυτά καρκινοειδών από την Αυστραλία, διότι είχαν αλλάξει οι κανόνες. Δυστυχώς όμως η δική μου εταιρεία, η εταιρεία που εκπροσωπώ, η Aqua Farm, μέχρι τότε είχε λάβει απολύτως καμία ενημέρωση από καμία αρμόδια ισπανική αρχή. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ως αθέμητη πρακτική απέναντι σε μια εμπορική επιχείρηση σαν αυτή την οποία εκπροσωπώ. Ξέρετε ότι στο αρχικό προφίλ της εταιρεία, αλλά ακόμα και στις επιδοτήσεις που μας δόθηκαν προβλεπόταν ότι μια εταιρεία σαν αυτή που εκπροσωπώ, που εισάγει ουσιαστικά ήδη από την Αυστραλία, μπορούσε να λάβει κοινοτική χρηματοδότηση και ξαφνικά μας είπαν ότι δεν ήμασταν επιλέξιμοι ούτε καν γι' αυτό. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι όλες οι αρχικές μας επενδύσεις, όλες οι επενδύσεις στις υποδομές, 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ήταν ε, δαπάνες τις οποίες αναλάβαμε για να στήσουμε την επιχείρηση, γίναν περαιτέρω επενδύσεις εν συνεχεία για τη βελτίωση αυτής της υποδομής και ξαφνικά είδαμε ότι δεν μπορούσαμε καν να εφαρμόσουμε το αρχικό μας επιχειρηματικό σχέδιο. Ζητήσαμε, όπως σας είπα, και μία υποστήριξη της τάξης των 270.000 ευρώ. Και αφού στήσαμε λοιπόν την επιχείρηση και αφού δόθηκε και απαραίτητη κοινοτική και εθνική υποστήριξη, μας ενημέρωσαν πολύ απλά ότι δεν μπορούσαμε πλέον να συνεχίσουμε με την εν λόγω επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα. Ξέρετε ότι ε, προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε σε εθνικούς και σε διεθνείς φορείς, αλλά δεν καταφέραμε να πετύχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ότι η απόφαση αυτή η οποία λήφθη σε εθνικό επίπεδο, που υποτίθεται ότι απορρέει από κάποια κοινοτική απόφαση, ουσιαστικά έχει βάλει κατά τις ίδιες της εικόνας επιχείρησης, κατά της οικονομικής βιωσιμότητας επιχείρησης αυτής, και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να καταφέρουμε να συνεχίσουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα τη στιγμή που δεν έχουμε καν έσοδα πλέον από αυτή τη δραστηριότητα. Νομίζω ότι κάθε φορά που λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις από τα κράτη-μέλη όταν μεταφέρουν κοινοτικέ οδηγίες ή γενικότερα όταν εφαρμόζουν το νοσιακό δίκαιο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, ότι εν μία νυχτή ουσιαστικά μια επιχείρηση μπορεί να πτωχεύσει, ακριβώς επειδή λαμβάνονται τόσο δραστικές αποφάσεις, οι οποίες στην αρχή ε, δεν, είχαν, δεν υπήρχαν καν α, α, ε, ε, πιθανό ενδεχόμενο. Δεν είχαν δοθεί ε, πληροφορίες Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να ποσοτικοποιηθεί ε, η ζημιά μας, το ότι έπρεπε να επανέλθουν τα εδάφη, το ότι υπήρξε μεγάλη, μεγάλο πλήγμα στη φήμη μας. Και ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πρώτον η αποζημίωσή μας ότι θέλουμε να είναι τουλάχιστον 5 εκατομμύρια. Ζητούμε να λάβετε υπόψη ότι εμείς τηρήσαμε και επί χρόνια καταβάλαμε προσπάθειες, κάναμε έρευνα, θυσία χρόνου, προσωπικού ε, χρόνου, οικογενειακού χρόνου και θέλουμε μια δίκαιη αποζημίωση για όλες αυτές τις προσπάθειε ε, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω το θέμα αυτό να μην το δείτε απλά ένα θέμα ε, νομικό, αλλά ε, πρέπει με τον ίδιο δίκαιο και νόμιμο τρόπο, όπως και εμείς με νόμιμο και δίκαιο τρόπο φέραμε σε πέρα τις υποχρεώσεις μας, να διευκαιριώσετε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ελπίζουμε μάλλον να υπάρξει ιδέουσα ευαισθησία για να μας δοθεί καλή τυπή στη ζητούμενη αποζημίωση ως απόδειξη το ότι εμείς φέραμε σε πέρα στις υποχρεώσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Thank you very much. The Commission Ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ποιος είναι σήμερα, ο κ. Λέινεμαν, η Γκουτ. Yes. Yes, thank you. Um, <clears throat> what I see the issue is... Από ό,τι κατάλαβα, είναι το εξή. Η Επιτροπή είναι δημόσια υπηρεσία. Και από την Αυστραλινή πλευρά πάλι με δημόσια υπηρεσία ε, έχουμε να κάνουμε. Δεν δίνουμε εγκρίσει σε εμπορικού φορεί, αλλά σε χώρε. Η Αυστραλία λοιπόν δεν έχει αυτή την έγκριση ακόμη. Δεν μπορεί να εξάγει τα προϊόντα αυτά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό είναι η αρμόδια αρχή, η Αυστραλιανή κυβέρνηση δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, να καταθέσει έτοιμα εξοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ξεκινήσουμε εμείς τότε τη διαδικασία μας, θα αξιολογήσουμε τις εγγυήσεις, ενδεχομένως θα κάνουμε ελέγχους και θα εγκρίνουμε ενδεχομένως τελικά την Αυστραλία. Ω χώρα η έπειτα θα πρέπει να παράσχει τα χέγγια πιστοποίηση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για αυτέ τι εγγυήσει που πρέπει να δοθούν. Και μόνο μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να παράσχει αυτέ τι εγγυήσει. Δεν βασιζόμαστε σε εμπορικού φορεί να δώσουν τι εγγύσει αυτέ. Και πρέπει να υπογραφεί πιστοποιητικό. Και μόνο ένα κτηνίας μπορεί να το υπογράψει το πιστοποιητικό αυτό. Πρέπει λοιπόν η Αυστραλία να ε, τύχει αξιολόγηση, να δοθεί έγκριση και έπειτα να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, ότι η Κομισιόν δεν έλαβε ποτέ μέχρι τώρα τουλάχιστον σχετικό αίτημα από την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς από μόνοι μα να αναλάβουμε δράση, δεν μπορούμε να ενεργήσουμε αν δεν υπάρχει αίτημα. Επομένως, Το θέμα είναι αν η εταιρεία έκανε τα δέοντα, εάν προσέγγισε την Αυστραλινή κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί απευθείας ένας φορέας εμπορικός από την Αυστραλία να απευθυνθεί στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you for Ευχαριστώ που μας ξεκαθαρίσατε με πολύ ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο το θέμα. Εδώ μιλάμε για την εσωτερική αγορά. Και το αίτημα είναι αυτό. Να μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά κάποια προϊόντα. Τώρα, όποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ, η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά την εταιρεία και ε, τους ε, επιχειρηματίες. Ήμουν και μέλος ε, της Αντολουσιανής Κυβέρνησης ε, πριν γίνω Ευρωβουλευτής ε, και γνωρίζω το θέμα. Γιατί είχαν ζητηθεί σχετικέ άδειε από την περιφερειακή κυβέρνηση τη Ανταλουσία από την επιχείρηση αυτή. Και πρέπει να σα πω ότι αυτό που γίνεται εδώ τώρα δεν θα έπρεπε να είχε γίνει. Πέραν των όσων είπε η Κομισιόν, πέραν των όσων είπε η Κομισιόν, λέγω, για την αναγνώριση των ειδών και τα αιτήματα που λέω ότι πρέπει να κατατεθούν από τη χώρα για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να έχουμε για μια σειρά ετών μια τέτοια επιχείρηση η οποία ζητά βοήθειες. Τις δίνονται οι ενισχύσεις αυτές, ε, η βοήθεια αυτή. και έφερε σε πέρα όλη αυτή τη διαδικασία περιφερειακή κυβέρνηση, εθνική κυβέρνηση τέλειξε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για χρόνια ολόκληρα. Και ποια είναι η τελευταία ε, φάση, το τελευταίο στάδιο, να μην μπορεί τελικά να ε, εισαχθεί από την επιχείρηση αυτή το συγκεκριμένο είδος. Και είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί το πρόβλημα δεν προέκυψε σε έξι μέρες, σε έξι μήνες, αλλά χρόνια ολόκληρα που επενδύει αυτή η επιχείρηση και έχει κάνει τα πάντα που έπρεπε να κάνει πήρε δημόσιες βοήθειες, ε, δημόσια ε, ενίσχυση και με αναγνώρισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα για αυτό το project, μεγάλη εμβέλεια έργο. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Εδώ πραγματικά ε, έχουμε πάρα πολλά ε, πράγματα πρέπει να υπόψη Ζημία προσωπική, επαγγελματική, επιχειρηματική. Και αυτό που λέει ο άνθρωπο αυτό ουσιαστικά είναι να μην επαναληφθεί στο μέλλον τουλάχιστον. Λέει υπάρχει τρομερό πρόβλημα έλλειψη συντονισμού. Και αυτά που λέει τώρα ο, ο αρμόδιο εκπρόσωπο Επιτροπή το λαμβάνω υπόψη για τα αιτήματα. Είμαι μέλο Επιτροπή Αλία επίση, θέλω να σα πω, και ο κύριο Βαλέ. Ε, και έχουμε την έκθεση για την υδατοκαλλιέργεια. Με βάση ακριβώ είναι πώ μπορούμε να προωθήσουμε την υδατοκαλλιέργεια. Αλλά αν έχουμε τέτοια φαινόμενα, πώ ε, να προωθηθεί τελικά η υδατοκαλλιέργεια ως εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό. Είναι ένα χείριστο παράδειγμα διαχείρισης. Αν θέλουμε να δώσουμε εναλλακτική ε, στην υδατοκαλλιέργεια, ε, γιατί έχουμε υπεραλίευση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σοβαρά διοικητικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Και σε μέρη, εν, οφείλονται και στην Κομισιόν. Αυτό το λέω για την υδατοκαλλιέργεια. Και ελπίζω να ε, δικαιωθεί η επιχείρηση αυτή και αυτό να είναι και ένα παράδειγμα για το μέλλον, να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε. Θα χρειαστεί να βάλω το ρολόι τώρα. Να είστε σύντομοι. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση απόψε. Γιάρεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να εργαζόμαστε μαζί στην Επιτροπή Αλίας, οπότε μπορούμε να μιλάμε για τα θέματα αυτά για ώρες για την υδατοκαλλιέργεια. Ξέρετε, είναι μία από, ένας από τους κλάδους με την ταχύτερη ανάπτυξη στον κόσμο. Αν δείτε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, έχουμε μείνει πίσω. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα ε, για τους ε, παραγωγούς. Αυτό το κομμάτι της οικονομίας δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Καλό είναι που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια όρια για την εμπορική αλία στα ανοιχτή θάλασσα. Οι υδατοκαλλιέργειες λοιπόν είναι το μέλλον. Για να έχουμε ψάρια και προϊόντα αλίας στο τραπέζι μας πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα. Να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν η παραγωγή όλη την υποστήριξη που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν όσο πιο ανταγωνιστικός ε, είναι ο τομέας ε, και όσο πιο αποτελεσματικός ε, τόσο το καλύτερο. Αυτός πρέπει να είναι ο μεγάλος μας στόχος και ο στόχος του σχετικού ταμείου. Σίγουρα δεν είναι δικό τους λάθος των ανθρώπων αυτών, είναι πρόβλημα της νομοθεσίας, είναι θέμα καλής συνεργασίας, οπότε σίγουρα έχουν δίκιο αναφερόμενοι και πρέπει να διατηρήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ρώσα. Eh. Ευχαριστώ. Όπως είπε και η Κλάρα Αγγιλέρα ε, και όπως είπε και ο δικός μου σύντροφος ε, Βαλέσα, δεν ε, είναι λογικό να κατατίθεται ένα έργο επιχειρηματικό να λαμβάνει την ενίσχυση και την ευρωπαϊκή και έπειτα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί, να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ποιος φταίει, τι γίνεται, εάν δίνεται μια βοήθεια δυνάμει της νομοθεσίας και ο ετών αυτή την ενίσχυση ξεκινά το έργο, φταίει. Πότε δεν φταίει ο επιχείρηση που έχει κάνει σωστά τη δουλειά τη. Αυτό που δημιούργησε τι προσδοκίε ε, φταίει. Δεν έπρεπε να τι και δημιουργήσει τι προσδοκίε. Και αν τι δημιούργησε, θα πρέπει να ε, προβεί σε αποζημίωση. Εγώ είμαι δικηγόρο και στο δίκαιο έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, αυτά λέει η νομική όταν σπουδάζει κανεί. Απλά η Κομισιόν αποστασιοποιείται εδώ ε, και λέει ότι δεν ε, φταίει σε τίποτα. Αλλά ας μην έδινε τις ενισχύσεις από τη στιγμή που τις έδωσε και το έργο αυτό όμως δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Ε, έχουμε το έτος που χάθηκε γιατί δεν μπόρεσε να ξεκινήσει το έργο και υπάρχει και το επόμενο έτος που επίσης έχει διαφυγόντα κέρδη ο επιχειρηματίας. Πρέπει να αποζημιωθεί. Και εντάξει, για το μέλλον λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει επιδότηση ή χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου. Αλλά αυτό αφορά το μέλλον. Εδώ μιλάμε για ένα έργο του παρελθόντος. Δεν είναι σωστό από πολιτικής πλευράς. Ε, ε και αυτό που γίνεται τώρα ε, δεν, ε, δεν είναι σωστό και νομίζω ότι ήρθατε πολύ ε, σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή εδώ εσείς οι αναφέροντες ε, γιατί πρέπει να δείξουμε λίγο μεγαλύτερο σθένος ε, και γενναιότητα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος πρέπει να αναλάβει ευθύνε και κάποιος υπεύθυνος πρέπει κάπως να λογοδοτήσει. Ευχαριστώ. I'm happy also Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξανδώσω τώρα το λόγο στους αναφέροντες για δύο ακόμα λεπτά. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απαντώντας στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φυσικά και ζητήσαμε από την Αυστραλία ε, τη διαχείριση. Ήταν δύο οι πολύπλοκες πτυχές. Πρώτον, στην Αυστραλία υπήρχε ένας μόνο παραγωγός που εξήγησε στο Βόρειο Μισφαίριο. Σε εμάς. Ήταν η πρώτη και μόνη άδεια για την ε, ε, εκτροφή και την εξαγωγή του είδους αυτού. Άρα ήταν πάρα πολύ λίγο για μια ελάχιστη εισαγωγή-εξαγωγή να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Και το δεύτερο που θέλω να πω. Σκεφτείτε το εξής. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση. Οι πολίτε μα, οι επιχειρήσει μα ε, θα πρέπει να μπορούν να καταθέσουν την ε, θεμητή αυτή εμπιστοσύνη. Ε, Ιδίω όταν μιλάμε για μια τέτοια σύμβαση δημοσιοδικού τομέα. Και φυσικά και πρέπει να υπάρχει και απαραίτητο έλεγχο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι κατάλαβα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε για το project αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ε, το ταμείο αυτό, το οποίο έδωσε την χρηματοδότηση, βρίσκεται σε καθεστώς έμεσης διαχείρισης, δηλαδή είναι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία το, κράτη, το κράτος μέλος αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για την χρηματοδότηση από το Ταμείο αυτό. Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα δεν εμπλέκεται τουλάχιστον στο πρώτο αυτό στάδιο. Σίγουρα είναι λυπηρό αυτό το οποίο συνέβη, αλλά δεν πρόκειται για άμεση πράξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε που διευκρινίσατε το ζήτημα αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και να ενημερώσουμε επίσης δεόντως την κατάλληλη στιγμή και τον αναφέροντα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Συμφωνούν οι συνάδελφοι. Πολύ ωραία, έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και ευχαριστώ και τους ε, αναφέροντες όλους ιδιαιτέρως. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη αναφορά. Την 0578 για την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Δανία για την επέκταση της υδατοκαλλιέργειας. Η αναφέρουσα είναι η Κριστίνε Μπίλε και μπορεί να Μπορείτε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Για πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σύμβαρο. Προφανώς διαβάσαμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου της Δανίας Γνωρίζουμε επίσης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλίας. Η Επιτροπή Γεωργίας αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γνωμοδότησή της μας λέει ότι τα όσα καταγγέλουμε δεν συνιστούν παραβίαση της κοινωτική νομοθεσίας. Μας λένε όμως ότι η Δανέζικη αυτή νομοθεσία δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή ούτε έχουν δοθεί περαιτέρω άδειες για επέκταση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Η κυβέρνηση της Δανίας από την άλλη λέει ότι η εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας δεν θα λάβει χώρα μέχρι το 2019. Επομένως, εμείς ζητούμε από την Επιτροπή σας να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά μέχρι τη στιγμή εκείνη που η Δανέζικη κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι έχει τεθεί πλέον επισήμως σε ισχύ ο κανονισμός αυτός. και θα θέλαμε έστω και αναδρομικά να γίνει μια επιτήρηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Και έχουμε και μια νέα εξέλιξη που καταδεικνύει ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με την ρήπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος που έχει προκύψει από την δέσμευτη μέτρων που εγκρίθηκαν το 2015. Έχουμε όλο και περισσότερη συγκέντρωση αζότου στο θαλάσσιο περιβάλλον και αυτό έχει συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια Ήδη από το 2010 έχει αρχίσει η συγκέντρωση αζότου στο θαλάσσιο περιβάλλον της Δανίας. Η ημερομηνία η οποία λήφθη υπόψη αρχικά ήταν εντελώς λανθασμένη. Στην πραγματικότητα η ρήπανση ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή άρχισε να εφαρμόζεται η νέα αυτή δέσμη μέτρων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είδαμε ότι είχε αυξηθεί η ρήπανση του θαλασσιού περιβάλλοντος. Νομίζω ότι ακριβώς αντίστοιχες εμπειρίες είχαμε και στα πλαίσια των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της γεωργίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε όλο και περισσότερο με τις επεκτάσεις αυτές μονάδων υδατοκαλλιέργειας που χρησιμοποιούν ε, ανοιχτού κλωβούς. Ο πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος μας είχε υποσχεθεί μία ανάλυση περιβαλλοντικού αντικτύπου, η οποία όμως δεν πρόκειται να γίνει από ό,τι φαίνεται μέχρι το 2019. Επομένως, όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν τη λειτουργία του ανενόχλητες εντελώς στη Δανία και βλέπουμε τώρα ότι το 2018 εγκρίθηκε τροποποίηση της ισχύουσας δανέζικης νομοθεσίας όσον αφορά την νομοθετική πράξη προστασίας του περιβάλλοντος. Με τις νέες εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις προβλέπονται τώρα θα αυξηθεί σίγουρα η ρήπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και όπως είχα πει και σε προηγούμενη καταγγελία, θεωρούμε ότι η δική σας η Επιτροπή, η Επιτροπή Αναφορών, θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά αυτή και ζητούμε από την Επιτροπή σας να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να ελέγχει αποτελεσματικά την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση της Δανίας προκειμένου να μην μολυνθούν περισσότερο τα νερά της χώρας. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εκπρόσωπος μάλλον, έχετε το λόγο. Η Λίντα Νίλουντ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Είναι περίπλοκο το πλαίσιο αυτού του ζητήματος όπως ανέφερε η λιντα νιλουντα απο την επιτροπη ευχαριστω κυρια προεδρε ειναι περιπλοκο το μέτρα για την γεωργία είναι κομμάτι ε, της ε, δεσμής μέτρων ε, τροφίμων και γεωργίας που συμφωνήθηκε στο Δανέζικο Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2015. Η δέσμη μέτρων βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τροφίμων στη Δανία και περιλαμβάνει 15 διαφορετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων την αύξηση της παραγωγής των ιδιωτικών καλλιεργειών. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η πρόσφατα υιοθετημένη τροπολογία στη σχετική πράξη για τα, τα αντισταθμιστικά ε, θαλάσσια μέτρα για τα υδάτινα ε, έργα έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική οδηγία. Αντιληθεύει ότι την 1η Ιουνίου πέρυσι, το 2017, το Δανέζικο Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια τροπολογία στην ε, πράξη προστασίας του περιβάλλοντος που δημιουργεί μια νομική βάση ώστε ο Υπουργός να θεσπίσει κανόνες όπου η έγκριση για νέες ιδεοκαλλιέργειες, για επέκταση υπαρχουσών εγκαταστάσεων μπορούν να λάβουν άδειες που να μπορούν να περιλαμβάνουν ε, συνθήκες συγκεκριμένες για συγκεκριμένα μέσα που να είναι αντισταθμιστικά στην ε, αποβολή ε, θρεπτικών ουσιών από αυτέ τι θεατοκαλλιέργειες. Δίνεται δηλαδή άδεια στον Υπουργό να υιοθετεί τέτοιου κανόνε. Αυτό ο παράγων μόνο του, όπω έχει ξαναπεί η Κομισιόν, δεν αποτελεί ωστόσο παραβίαση τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό το συμπέρασμα όμω δεν εμποδίζει την Επιτροπή από το να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δανία ώστε να διασφαλίσει ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παραβιάζεται. Ευχαριστώ. The floor is open to members. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχουν τα μέλη. Γιάρεκ, θα είμαι απλός. Το αίτημα της αναφέρουσας πιστεύω είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να παρακολουθούμε. Νομίζω ότι το αίτημα της αναφέρουσας είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να παρακολουθούμε την κατάσταση, να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, να προσέχει την όλη κατάσταση και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Έχουμε ακόμα ένα έτος και παραπάνω. Οπότε α μην το χάσουμε από τα μάτια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μάργκρετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα και να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ένα ακόμα παράδειγμα πολιτών που έρχονται σε μια κατάσταση post-mortem ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή έχει συμβεί το κακό, καλείστε εσείς να, να έρθετε να διορθώσετε τα κακό σκήμενα. Ενώ έρχονται πολίτες και σας προειδοποιούν εδώ πέρα ότι μια εθνική νομοθεσία ουσιαστικά θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στο περιβάλλον, εσείς μας λέτε ας περιμένουμε και θα δούμε. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε όμως ότι στη Δανία έχουν γίνει συγκεκριμένοι υπολογισμοί για το ανώτατο ύψος ε, αζότου που μπορεί ποτέ να υπάρχει στο περιβαλλοντικό λεγόμενο χώρο. Είναι 800 τόνοι αζότου και 96 τόνοι φωσφόρου. Ξέρετε όμως ότι παλιότερα, το 1980, στο Δανέζικο Κοινοβούλιο, λέγαμε ότι τα ύδατα της Δανίας θα μπορούσαν να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες τέτοιων ουσιών. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι ακτές της Δανίας αλλά και της Σουηδίας από την προβλεπόμενη αυτή αύξηση της μόλυνσης. Και δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα μόνο σε θρεπτικές ουσίες, σε μόλυνση από θρεπτικές ουσίες, αναφερόμαστε και σε μόλυνση από φαρμακευτικά προϊόντα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αναφερόμαστε σε ύδατα τα οποία είναι ήδη πολύ μολυσμένα και ξαφνικά φαίνεται εδώ πέρα να προωθούμε όλο και περισσότερο μια εντατική καλλιέργεια μειώντα ουσιαστικά τους κανόνες ελέγχου της και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Πρέπει λοιπόν να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να λαμβάνει δράση προτού συμβεί το κακό, όταν ακόμα τώρα μπορούμε να προλάβουμε την κατάσταση. Πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης, πάση θυσία, αυτή τη στιγμή υπάρχει αρχή αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να την εφαρμόσει, οφείλει να την προασπίσει. Και κάτι ακόμα. Έχουμε και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος προς την Επιτροπή Αλίας, στην οποία λέγεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται και οι οποίες δεν πληρούνται προκειμένου. Και κάτι τελευταίο και ολοκληρώνω. Υπάρχουν ε, ήδη πολλοί πολίτες που έχουν ζητήσει να πάρουν άδεια για μονάδες καλλιέργειας, αλλά ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν σε μια πολύ επισφαλή κατάσταση, γιατί δεν γνωρίζουν αν στο μέλλον θα τους δοθεί τελικά η άδεια αυτή, εφόσον δηλαδή γίνει μια εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτό που θα έλεγα στην δανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σταματήστε εδώ πέρα, έχουμε ήδη αρκετές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ας μην τις πολλαπλασιάσουμε, ας μην μολύνουμε ακόμα περισσότερο τα ύδατα της χώρας αυτής. Ας μην ξεχνάμε ότι ε, έχουμε και άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, χώρες οι οποίες κινδυνεύουν από την απόφαση αυτή. Όχι μόνο η Δανία λοιπόν. Ελπίζω θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους θα αναλάβει έγκαιρη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή που έχει προκύψει και ιδιαίτερα χαλαρή στάση που κρατάει η Δανία για το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο συνάδελφο θέλει να πάρει το λόγο για αυτή την υπόθεση. Να ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην αναφέρουσα για άλλα δύο λεπτά αν το επιθυμείτε. Γιατί όχι. Δύο πολύ σύντομα σχόλια από πλευρά μου. Ασπάζομαι απόλυτα τα όσα είπε η Μαγκρέτε Άγκαρν. Δεν υπάρχει απαρκή φιλοδοξία. Επειδή δεν έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο της μόλυνσης, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να μολύνουμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτό, ούτε φιλόδοξα. Σε αυτό πρέπει να παραμείνουμε πιστοί, να μην το ξεχνάμε. Να πω κάτι άλλο για τα αντισταθμιστικά μέτρα. Ε, το να χρησιμοποιούνται καλλιέργειε με γι' αυτό. Δεν είναι κανεί σίγουρος για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Αλλά ακούμε τώρα ότι δεν πρέπει να βρίσκονται καν κοντά στι ηχθειοκαλλιέργειε. Πρέπει να βρίσκονται κάπου αλλού ε, για, και μπορούν να αντισταθμίσουν ούτω ή άλλως ε, Δηλαδή τι σημαίνει ότι μπορούμε να ρηπαίνουμε όσο θέλουμε με διοξίδιο του άνθρακα οπουδήποτε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ούτε επαρκώ φιλόδοξα. Ελπίζω να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά έω ότου ολοκληρωθεί η ανάλυση του σημείου αυτού και έω ότου υλοποιηθεί η νομοθεσία στη Δανία. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Σειρά μου είναι τώρα για να κλείσω. Ήθελα να το πω σε μια σκανδιναβική γλώσσα γιατί ένιωσα ξαφνικά στο σπίτι μου. Αλλά Ας ε, πράξουμε όπως λέμε, ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή των συναδέλφων, διατηρούμε ανοιχτή την ε, αναφορά και θα εντείνουμε τις επαφές μας με την Κομισιόν, η οποία υποσχέθηκε να παρακολουθεί την κατάσταση. Ε, σας ενθαρρύνω να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας τα πορίσματά σας. Αν μπορείτε να μας στέλνετε γραπτός ό,τι παρατηρείτε και εμείς από πλευράς μας θα στείλουμε μια επιστολή στη δανική κυβέρνηση όπου θα επισημαίνουμε ότι παρότι δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική παραβίαση της νομοθεσίας, ε, το θέμα είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οπότε πρέπει να το προσέχουμε. Ας επιστήσουμε την προσοχή τους λοιπόν στην κατάσταση και θα το παρακολουθούμε και εμείς ως θεσμικά οργάνα μαζί με την Κομισιόν. Μπορούμε να... Fine. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία. Καλό ταξίδι. Καλή επιστροφή στη Δανία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η παρουσίαση μελέτης για τον νόμο περιφορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών οργανών ΦΑΤΚΑ. Με τα χαράς καλώ τον καθηγητή Κάρλο Γκαρμπαρίνο από το Πανεπιστήμιο Μποκόνη του Μιλάνου να πάρει το λόγο. Είμαστε πολύ περήφανοι και ευτυχείς σας έχουμε μαζί μας και περιμένουμε τη ομιλία που θα κάνετε και να ακούσουμε τα βέβαια ενδεχομένω και συστάσεις που έχετε να διατυπώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χρόνο έχω, 15 λεπτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμά και εμένα πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να απευθυνθώ στην Επιτροπή Αναφορών. Το θέμα που μας απασχολεί μπορεί να φαίνεται ένα ε, καθόλου ενδιαφέρον τεχνικό ζήτημα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την πολυπλοκότητα, το πολύπλοκο αυτό ζήτημα και τις πτυχές του. Θα ξεκινήσω με μια ιστορική αναδρομή. Οι χώρες φορολογούν τους υπηκόους τους φορολογούν το εισόδημά τους και πρέπει να δηλώνουν τη... στους λογαριασμούς που έχουν στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται με ανταλλαγή πληροφοριών. Ζητάει μια χώρα από την άλλη πληροφορίες για τους υπηκόους της και τους νομίμως διαμένοντες εκεί. Υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα, περιλαμβάνονται οι διαταξίες και οι συνθήκες και υπάρχουν και οι συμφωνίες ε, ανταλήσεις φορολογικών πληροφόρων. Τα τελευταία 10-15 χρόνια υπήρξε μια εκστρατεία για την ε, παροχή αυτών των πληροφοριών. Το 2010 ε, και στο μέσο της χρηματοπιστωτικής κρίσης οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δρομολόγησαν ε, αυτό το νέο σύστημα, ΦΑΤΚΑ, και τότε υπήρξαν πολλές εξελίξεις, τώρα πλέον είναι αυτόματη σχεδόν αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών Δηλαδή είναι ρουτίνα η ανταλλαγή πληροφοριών από τις φορολογικές διοικήσεις για τις ε, ε, των βουλικών δηλώσεων. Ε, ο νόμος αυτός ε, περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών ε, ΦΑΤΚΑ έχει την εξής διαφορά από άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Οι τράπεζες υποχρεούνται από τις ΥΠΟ που και αν αυτές έχουν την έδρα τους, να δίνουν πληροφορίες για τους ε, επικόσαμε πολιτείων και αν δεν συμμορφούνται ε, υπόκεινται σε κυρώσεις. Και είναι πολύ αποτελεσματικό το αποτρεπτικό αυτοκίνητο γιατί όλες οι τράπεζες δραστηριοποιούνται στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν δικυβερνητικέ ε, συμφωνίες με διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά διεθνείς συμφωνίες που πολλές φορές προβλέπουν υποχρέωση της κυβέρνησης ε, να επιβάλλει αυτές τις ε, υποχρεώσεις. Μου ζητήθηκε λοιπόν να αναφερθώ στον αντίκτυπο ε, αυτού του νόμου και πρακτικά τι στοιχεία κρίσιμα τον χαρακτηρίζουν αυτόν τον νόμο. Πρώτα απ' όλα αυτός ο νόμος εφαρμόζεται ακόμη και αν οι τράπεζες δεν είναι κατεστημένες, ε, δεν έχουν την έδρα τους στη ΣΥΠΑ. Εξοεδαφική δηλαδή η φύση του νόμου αυτού. Επίσης μιλάμε για αμοιβή ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό τουλάχιστον προβλεπόταν στην αρχή. Αλλά στην ουσία εξελίχθηκε σε μονοδρομή, μονομερή ε, ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή μόνο οι υπόλοιπε χώρε στέλνουν στη ΣΥΠΑ πληροφορίε και όχι οι ΥΠΑ στι άλλε χώρε. Mm, has created uh, Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, συστημικές ε, και ποια είναι τα συστημικά εξωτερικά στοιχεία της, ε, του νόμου αυτού. Είναι από τα βασικά σημεία νομίζω της αναφοράς είναι ακριβώς ένα, μια διάταξη της σχετικής νομοθεσίας, τον είπα. Αρκεί να είναι ε, υπήκοοι ε, και δεν χρειάζεται να είναι ε, διαμένοντες, δηλαδή να είναι citizens και όχι residents. Αυτό είναι ένα στοιχείο αυτής της ε, νομοθεσίας. Υπάρχουν κάποιοι που γεννήθηκαν στη ΣΥΠΑ, χωρίς να έχουν όμως κανένα άλλο δεσμό. Λόγω όμως ε, όλου αυτού του μηχανισμού που επιβάλλει στις τράπεζες ε, να δίνουν στοιχεία για όλους, υπάρχουν και Ευρωπαίοι πολίτες που από σπόντα ε, γίνονται Αμερικανοί πολίτες. Αυτοί λεγόμενοι accidental Americans. Και πρέπει να παρέχουν αυτές τις προφορές. Και αυτό δείξα στην εξή κατάσταση. Πολλές τράπεζες εμπορικώς αρνήθηκαν να παρέχουν ε, υπηρεσίες στους ε, υπηκόους αυτούς, στους πολίτες αυτούς. Ή ακόμη και αν δέχονταν να τους παρέχουν υπηρεσίες, ε, θα έπρεπε να δίνουν αυτοί οι άνθρωποι του κόσμου της πληροφορίας. Πάρα πολύ πολύπλοκο αυτό. Θέλω να πω ότι απέχουμε 10 μέρες από τη θέση ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ένας ευρύτατος κανονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργείται πλέον ένα θεμελιώδη δικαίωμα το δικαίωμα της προστασίας δεδομένων, το οποίο είναι διαφορετικό από το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, privacy. γιατί ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα και τους φορολογουμένους για να μπορούν να του φορολογούν. Αλλά το δικαίωμα της προστασίας ε, ε, δεδομένων είναι πρόσθετο δικαίωμα, πολύ σημαντικό. Και αυτό θα καλύψει όλους τους τομείς, φορολογικά στοιχεία αλλά και big data και όλα τα άλλα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να υποθεί εδώ είναι πως όταν οι ευρωπαϊκές τράπεζες δίνουν σε μια τρίτη χώρα, τη ΣΥΠΑ, πληροφορίες για υπηκός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε υπάρχει απέτηση συμμόρφωσης προς αυτό τον νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων, το GDPR. και πολλές φορές υπάρχουν κάποια, κάποια αντικρώμενα συμφέροντα. Δεν ξέρω αν διαβάζετε πολύ καλά τι λέει το άρθρο 23 του GDPR, του κανονισμού για την προστασία δεδομένων λέει ότι οποιοδήποτε περιορισμό και στο φορολογικό τομέα θα πρέπει να σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και πρέπει να είναι ένα μέτρο απαραίτητο και αναλογικό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι ότι τώρα οι ΙΠΑ απαιτούν να λαμβάνουν φορολογικέ πληροφορίε για να προστατεύσουν τα δικά του εθνικά συμφέροντα, όχι τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ κρατών μελών και αυτό είναι προφανές, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την έλλειψη αμοιβαιότητα. Αν λοιπόν θέλαμε να προστατεύσουμε τα κοινά συμφέροντα για να μειωθεί η φοροαποφυγή και η φοροδίφυγη, αλλά και από τις δύο πλευρές, θα έπρεπε να υπάρχει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. και θα ήταν πιο δικαιολογημένη η, η λιγότερα αστήρη ε, περιορισμή στην ανταλλαγή πληροφοριών με τη ΣΥΠΑ. Από τη στιγμή που δεν είναι παρά μονόδρομη μονόπλευρη παροχή αυτών των στοιχείων, είναι λιγότερο κατανοητό αυτό. Επίσης, θέλω να τονίσω το εξή. Υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον κανονισμό το γενικό για την προστασία δεδομένων, το οποίο αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, όπως είπα. Και αυτό αφορά όλα τα δεδομένα, όχι μόνο τα φορολογικά. Η συλλογιστική είναι προφανής. Ποιο είναι το σκεπτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται διαφάνεια, λογοδοσία και άλλα χέγγια. Όταν όμως ο παγκοσμιοποιημένο κόσμο έχουμε μεταφορά μέσα σε μια τρίτη χώρα ως Ευρωπαίοι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα χέγγια αυτά διατηρούνται, παραμένουν σε ισχύ. Περάσουμε στο τμήμα αυτό που αφορά βασικά τα συμπεράσματα τα δικά μου ή κάποιες προτάσεις που κάνω για θέσπιση πολιτικής, συμπεράσματα που θα μπορούσε να εξετάσει η δική σας η Επιτροπή και που ενδεχομένω να εφαρμόσουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ προφανώς ασχολούμεθα με την νομοθεσία και των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως από πολιτικής πλευράς είναι κάπως πολιτικά ευαίσθητο το ζήτημα. Καταρχάς, προφανώς υπάρχουν διμερεί μέτρα. Έπειτα μπορούμε να έχουμε μονομερή μέτρα από την αμερικανική, την ευρωπαϊκή πλευρά και τέλος, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, εδώ στην Ευρώπη προωθούμε σαφώς τις πολυμερείς σχέσεις. Και ακριβώς αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να προωθήσουμε και εν προκειμένου. Κανείς δεν αρνείται ουσιαστικά ότι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Εφόσον λοιπόν η ανάγκη αυτή έχει διεθνείς διαστάσεις, διεθνή και πολυμερή θα πρέπει να είναι και τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν. Κάνω λοιπόν κάποιες πρακτικές προτάσεις εδώ πέρα. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναδιαπραγματευτεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες τις διεθνείς αυτές συμφωνίες προκειμένου αυτές να ευθυγραμμιστούν καταρχάς με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων και να τις επανεπραγματευτεί προκειμένου να είναι πραγματικά αμφίδρομες και αμοιβαίε. Νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση αυτή και οι Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα και με την κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει τουλάχιστον να ακούσει το αίτημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τις διαπραγματεύσεις θα ήταν η λήψη μονομερών μέτρων. Αν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν τιμήσουν το καθήκον αμοιβαιότητος το οποίο έχουν, τότε νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει μονομερή δράση και να ανακοινώσει μια νομοθεσία η οποία θα μπλοκάρει ουσιαστικά κάποια δεδομένα από το να μεταφερθούν αυτά στι Ηνωμένε Πολιτείες και θα τα απελευθερώσει εντό αγωγικών πάλι αυτή τη στιγμή επιστρέψει ένα καθεστώς αμοιβαιότητος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την παρεμπόδιση αυτή της Αμερικανικής νομοθεσίας, να μην μεταφέρουμε δηλαδή δεδομένα όταν η μεταφορά αυτή δεν συνάδει, δεν συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αποσύρουμε κάποιες πληροφορίες να μην διαβιβαστούν στι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας δούμε ένα ακόμα στοιχείο τώρα. Η δυνατότητα ανάληψης μονομερούς κοινοτική δράσης, μιας εγκάρσιας δηλαδή πολιτικής, ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε το άρθρο 8 κατά της διακριτικής μεταχείρισης και το άρθρο 14 για την προστασία της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Είναι λοιπόν δυνατό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει συγκεκριμένες υποθέσεις και να αποφασίσει τελικά ότι εξαιτίας αμερικανικής αυτής νομοθεσίας υπάρχει παραβίαση της οικογενειακής και ιδιωτική ζωής των ε, λεγόμενων ε, Αμερικανών λόγω συγκυριών, των Accidental Americans. Ξέρετε ότι ε, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να είναι δυνατή. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσε να λάβει η Αμερική και στα οποία θα μπορούσε να αντιδράσει έπειτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την απόφαση αυτή μόνο ο Αμερικανός νομοθέτης μπορεί να πάρει. Και εδώ αναφέρομαι στο σύστημα αυτό της φορολόγησης βάση ηθαγένειας. Στα πλαίσια του στήματο αυτού γίνεται ένα έλεγχο τώρα στι ΗΠΑ γιατί θεωρείται ότι αυτή η φορολόγηση είναι ιδιαίτερα ευρεία. Ακριβώς λοιπόν επειδή Υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες οι οποίες πρέπει να υποβάλουν πάρα πολλά στοιχεία στα πλαίσια του νέου αυτό φορολογικού νόμου. Συντοποιούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικάνοι λόγω συγκυριών οι οποίοι καλούνται να διαβιβάσουν στοιχεία στις ε, Αμερικανικές φορολογικές αρχές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αυξήσουμε το κατόφλι το οποίο είναι 50.000 δολάρια αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσό αυτό ή θα μπορούσε να εξαλειφθεί εντελώς η υποχρέωση υποβολή στοιχείων από τους Αμερικανούς λόγους συγκυριών ή θα μπορούσαν αυτοί οι Αμερικάνοι λόγους συγκυριών ή ακόμα και οι Αμερικάνοι πολίτες να αποχωρήσουν από την Αμερικανική ηθαγένεια χωρίς όμως αυτό να επιφέρει κάποιο κόστος. Και τέλος, και ολοκληρώνω κύρια Πρόεδρε, Πρέπει να τονίσω και κάτι ακόμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολυμερή προσέγγιση στη ρύθμιση της ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Ήδη από το 2010 υπάρχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχουν προσχωρήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε όμως. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, θα ήταν πάρα πολύ θετικό να είχαμε ένα πολυμερές παγκόσμιο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών, στο οποίο να συμμετέχουν και οι Πολιτείε. Θα μπορούσαμε να είχαμε όχι απλώς ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε καν διαβίβαση πληροφοριών, αλλά πραγματικό επιμερισμό δεδομένων και πληροφοριών με έναν τρόπο αμοιβαίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή και που μας αφήσατε και αυτό το έγγραφο. Είναι πολύ καλό, θα μας βοηθήσει ειδικό, ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Θα επανέλθω στον Φραντς Κάφκα και στον Τζόσεφ Κέι. Θυμάστε τον Τζόσεφ Κέι να κατηγορείται κάτι για κάτι το οποίο έμοιαζε με αυτούς τους Accidental Americans για κανέναν απολύτως λόγο και να μπλέξει άσχημα. Μιλάτε για αμοιβαιότητα, μιλάτε για διμερείς συμφωνίες. Εδώ και χρόνια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε αυτό το κοινοβουλίο, όπου οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να παίξουν μαζί μας. Ενώ το παιχνίδι παίζεται με δύο. Διαρκώς πρέπει να τους ασκούμε πίεση. Ξανά και ξανά. Το θεωρώ τελείως παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Και αυτή η οι Αμερικανοί από συγκυρία έχουν έρθει, έχουν στραφεί στην Επιτροπή μας. Πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Αυτό είναι βέβαιο. Όχι σήμερα, αλλά θα ήθελα να ενθαρρύνω τώρα την Κομισιόν να πάρει το λόγο και να μας πει τη δική της άποψη. Ε, πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό Ευρωπαίοι πολίτες να αποτελούν το αντικείμενο δυτικής μεταχείρισης. Ε, δίνω το λόγο στον κύριο Τζερμάνο Μιράμπλε. Or did you prefer not to speak? Ή μήπως δεν θέλετε να μιλήσετε. I was not supposed to speak, but... Δεν ήταν να μιλήσω νομίζω, δεν είχε προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή είναι η επόμενη αναφορά για το ίδιο θέμα, μια παρουσίαση που είχε προβλεφθεί να μιλήσω εκεί Κοιτάξτε, ναι, όντω, απλά εγώ σα ζητάω αν έχετε την ευγένεια έτσι να πείτε κάτι για τον καθηγητή. Ναι, για τα όσα είπε μόλι. Ε, αν θέλετε να εκφράσετε την εκτιμήσή σα, κάποια ερώτηση, οτιδήποτε. Μπορείτε και να μην πάρετε το λόγο. Κοιτάξτε, ε, ένα διαδικαστικό. Η ανάλυση του κυρίου καθηγητή βασίζεται στο γενικότερο σύστημα διακυβερνητικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων. Εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών διακυβερνητικών συμφωνιών, δύο IJ, αλλά αυτές προσαρμόζονται στην επιμέρους σχέση μεταξύ του ε, κάθε κράτους μέλους και των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές από αυτές τις συμφωνίες υπάρχει τέτοια αμοιβαιότητα. Δεν αποκλείεται, αλλά ακόμη και χωρί απόλυτη συμμετρία υπάρχει κάποια αμοιβαιότητα. Αυτό το αναφέρω εγώ διαδικαστικά, διότι εάν οι επιμέρου συμφωνίες κάποιων κρατών μελών με τι ΗΠΑ, ε, αν τι αναλύσουμε αυτέ τι συμφωνίε μπορούμε να αλλάξουμε κάποια, ε, μπορεί να αλλάζουν κάποια εχέγγυα διότι υπο, υποβλήθηκαν στου εθνικού επόπτε προστασία δεδομένων πριν υιοθετηθούν και υπογραφούν και εκεί υπάρχει κάποια διαφορά σε θέματα αμοιβαιότητα. Οπότε θα πρέπει να γίνει πολύ ευρεία και βαθιά ανάλυση για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα κατά την άποψή μου, αλλά είναι προσωπική άποψή μου από τα όσα γνωρίζω εγώ. Πρόεδρο ε, ωραία, έχουμε τώρα και τι δικέ σα προσωπικέ απόψει για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την γενοδορία με την οποία μα προσφέρατε ε, τι πληροφορίε που ξέρετε. Αν τα μέλη έχουν κάποια ερώτηση προ ε, τον κύριο καθηγητή που μα έκανε την παρουσίαση. Αν όχι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του Αμερικανικού νόμου περιφορολογική Συμμορφώσης αλλοδοπών λαγοργασμών για του πολίτε Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως για τους λεγόμενους Accidental Americans. Λοιπόν, Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους της Κομισιόν που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Σας καλώ λοιπόν να πάρετε πράγματι το λόγο. Πριν σας διαβάσω την ενημέρωσή μου, θα ήθελα να σας πω ότι ο ΦΑΤΚΑ ε, απλά αναδεικνύει μια προϋπάρχουσα κατάσταση. Διότι όταν κάποιο είναι Αμερικανό πολίτη, υπόκειται στο Αμερικανικό φορολογικό σύστημα. Το θέμα είναι ότι και πριν το ΦΑΤΚΑ δεν υπήρχε υποχρέωση αναφοράς ε, ε, για τα δικά μας ε, τραπεζικά ιδρύματα να παρέχουν πληροφορίες στις Αμερικανικές Αρχές. Ένα σωρό ο κόσμος λοιπόν με διπλή υπηκότητα ζούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν Αμερικανοί πολίτες και έπρεπε να πληρώνουν φόρους στην Αμερική. Ένας πολύ συνάδελφός μου στην Κομισιόν είχε τέτοια διπλή υπηκότητα. Δεν είχε απλά γεννηθεί όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ζήσει εκεί, είχε σπουδάσει εκεί γνώριζε δηλαδή τις φορολογικές υποχρεώσεις στην οποία ήταν υποκειμένη στις ΗΠΑ. Σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση ε, έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι γεννήθηκαν μεν στις ΗΠΑ και το είδαμε στη γαλλική τηλεόραση τις προάλλες πριν δύο εβδομάδες περίπου στις, στο κύριο Δελτίο Ειδήσεων ο Πέργιο Κόσμος ξέρετε γεννήθηκα στο Σικάγο έζησα εκεί δύο εβδομάδες και μετά η οικογένεια μου έφυγε από τι ΗΠΑ. αλλά τώρα ξαφνικά ανακαλύπτω ότι ε, πρέπει να πληρώσω ε, φόρο στην Αμερική διότι το βρήκε η τραπεζά μου ότι γεννήθηκα στην Αμερική και με υποβάλλει ε, στο φορολογικό σύστημα των Αμερικανών. Υποτίθεται στη Γαλλία, λέμε βέβαια έχουμε την αρχή ότι κανείς δεν υποτίθεται αγνοεί τον νόμο, αλλά αυτό ήταν πραγματικά γιατί καινούριο. Είναι τόσο χαλαρός αυτός ο δεσμός αυτών των ανθρώπων με τη ΣΥΠΑ που πραγματικά του εξέπληξε. Είναι Γάλλοι πολίτε, πολίτε οποιασδήποτε χώρα, αλλά ο νόμο είναι αυτό που είναι. Δεν ε, του αφήνουν άλλη επιλογή, δυστυχώ. Υποχρεούνται να αναφέρουν στην Αμερική τα έσοδά τους και να υπόκεινται στην Αμερικανική φορολογία. Το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών ότι υπήρχε δυνατότητα να εγκαταλείψει κανείς την Αμερικανική υπηκότητα. Αυτό όμως έχει ένα κόστος. Το είδαμε και στην γαλλική τηλεόραση. Κάποιοι άνθρωποι ε, χρειάζονται νομικούς συμβούλους, κυρώσεις, διότι δεν είχαν αναφέρει έγκαιρα. Δεν είχαν στείλει ε, τις δηλώσεις τους έγκαιρα στην Αμερική και έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμο και μετά έπρεπε να πληρώσουν και πρόστιμο για να εγκαταλείψουν την Αμερικανική του υπηκότητα. Όπω ε, συνέβη με τον Μπόρι Τζόνσον ε, πριν από μερικού μήνε πέρυσι. Αυτό συνεπάγεται δαπάνε, αλλά υπάρχουν ε, οδοί διαφυγή. Τώρα, όσον αφορά εμένα, το θέμα είναι τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την Οδηγία για τους Λογαριασμούς Πληρωμών. Εμείς έχουμε ερευνήσει τα κράτη-μέλη, έχουμε αναλάβει διάφορες δράσεις όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα τραπεζικά ιδρύματα. Έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και τις ενώσεις του κλάδου για να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, να μάθουμε πόσοι ε, κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται να ε, γίνουν δεκτοί σε τραπεζικές υπηρεσίες γιατί υπόκειται στο φάτια και επειδή πρέπει να δώσουν κάποιο αριθμό ε, αφημίου, ουσιαστικά αμερικανικό στις τράπεζές τους. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, αλλά υπάρχουν ε, λόγοι γι' αυτό. Διότι όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε διοικητική και συνεργασία και το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτούμε μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι διαφορετικό από αυτό που ζητούν οι ΙΠΑ. Το ζήτημα που έχουμε με την Αμερική, με τους Accidental Americans, είναι ότι έχουν αυτή την απόσταση με τις ΗΠΑ εκ των πραγμάτων. Κατά τα άλλα όμως, αν ένα 40χρονο ζού είχε ζήσει 30 χρόνια στη ΣΥΠΑ, θα γνώριζε την υποχρέωση αυτή. Το θέμα αφορά περισσότερο αυτού που ονομάζουμε Accidental Americans, του ε, Αμερικανού κατά συγκυρία, από συγκυρία. Ζητήσαμε λοιπόν να μάθουμε πόσε τέτοιε περιπτώσει υπάρχουν και δεν λάβαμε ιδιαίτερα στοιχεία. Επίση, ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, αρχή να συμβουλευτεί τα κράτη, του εθνικού επόπτε επί του ζητήματο για να μάθουν πόσοι οι καταναλωτέ δεν μπόρεσαν να ανοίξουν λογαριασμό ή να διατηρήσουν ε, τραπεζικό λογαριασμό λόγω του ΦΑΤΚΑ, διότι αυτό είναι που μα αφορά ουσιαστικά στη γενική μα διεύθυνση. Όπω προκύπτει από την έρευνα αυτή, μόνο μία εθνική αρχή έλαβε καταγγελία σε σχέση με τον ΦΑΤΚΑ. Μικρός αριθμός δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για το εν λόγω άτομο, αλλά προς το παρόν ε, δεν έχουμε στοιχεία ε, συστημικού προβλήματος. Επίσης θέσαμε το ζήτημα ε, και με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μας για τις υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Λιανικής τον περασμένο Απρίλιο. Γιατί δεν έχουμε συμπεράσματα. Ε, μετά από αυτή την έρευνα ο λόγος είναι ότι ο κόσμος δεν το γνώριζε. Οι δημόσιες αρχές δεν γνώριζαν, οι εμπειρογνώμονες τέλος πάντων που βρίσκονταν στην αίθουσα δεν γνώριζαν για το πρόβλημα. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ναι, ίσως να είναι κακόμπιστο, αλλά όπως φαίνεται ε, σε πολλές δικαιοδοσίες ο κόσμος, οι δημόσιες αρχές δεν γνωρίζουν το θέμα. Και αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της δικής μας έρευνας στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ε, και κλεισμένο των θύρων μπορεί να μιλούσαν πιο ανοιχτά, αν το γνώριζαν. Ε, και μα είπαν ότι είχαμε μόνο ένα περιστατικό. Τι δέσμευση μπορούμε να λάβουμε εμεί ω Κομισιόν, λοιπόν, όσον αφορά εμά. Όσον αφορά την οδηγία λογαριασμών πληρωμών, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε διαδικασία επιπαραβάση εφόσον προκύψει ότι το δικαίωμα πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό, όπω προβλέπεται από την οδηγία, απορρίπτεται σε οποιονδήποτε Αμερικανό πολίτη ε, εντό εισαγωγικών ή σε κάποιον accidental American αν δεν είναι σε θέση να δω... ακόμη και αν είναι σε θέση να παρουσιάσει τον αμερικανικό του αφημί ε, και λέει ότι δεν έχω πρόβλημα να ότι ο φόρους μου μέχρι ότου εγκαταλείψω την αμερικανική μου υπηκότητα. Αν μιλήσει δηλαδή καλόπιστα. Αλλά βλέπουμε ότι οι τράπεζες υφίστανται έναν διοικητικό φόρτο απορρίπτουν την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ένα βασικό λογαριασμό για αυτούς του accidental Americans. Οπότε παρακολουθούμε την κατάσταση. Πολλά βήματα θα ληφθούν, του χρόνου βέβαια, αλλά δεν θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου για να προσαρμόσουμε τις δράσεις μας. Μόλι λάβουμε πληροφορίε ε, για τι καταγγελίε, ε, οι καταγγελίε πρέπει να εξετάζονται αρχικά σε εθνικό επίπεδο από τι εθνικέ αρχέ. Εφόσον εμεί αντιληφθούμε ότι οι εθνικέ αρχέ ε, ε, αποτυγχάνουν στην επιβολή της οδηγίας λογαριασμών πληρωμών, τότε θα δράσουμε. Αυτά όσον αφορά τη δική μας Γενική Διεύθυνση. Τώρα να πάρω το λόγο και για τα θέματα προστασίας δεδομένων, εκτός αν θέλουν οι συνάδελφοι, για την προστασία δεδομένων, λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στην Επιτροπή και στην Γραμματεία ε, που μοιράστηκε μαζί μας την εκθέση του κ. Γκαμπαρίνα. Εμείς λάβαμε την έκθεση χθε μόλι. Χρειάζεται να διαβάσουμε και να δούμε, αφού θα την έχουμε διαβάσει ε, επιμελώς, ποια είναι τα πορίσματα και κατά πόσο απαιτείται επακόλουθη δράση από πλευρά μα. Ήδη όμω αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων θέλουν να επιληφθούν του ζητήματος και μάλιστα πρόσφατα το Φεβρουάριο έστειλαν μία επιστολή στην ομάδα στον Ευρωπαϊκό Αυτοσύλλογο των Αμερικανών Λόγω Συγκυριών λέγοντας το εξής, ότι στα πλαίσια του καθεστώτος ΦΑΤΚΑ θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ ακριβώς ποια δεδομένα απαγορεύεται να διαβιβαστούν Φαίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολλές εθνικές αρχές φορολογικές και αρχές προστασίας των δεδομένων οι οποίες λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις βασικές αρχές, εθνικό τουλάχιστον επίπεδο. Και όπως είπε και ο Τζερμάνο πριν από λίγο, απαντώντας στον καθηγητή Καμπαρίνο, οι βασικές αρχές που διέπουν τον ΦΑΤΚΑ είναι βασικά διακρατικές συμφωνίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα είχε προτείνει τις δικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπραγματευτούμε μία πολυμερή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη-μέλη πολύ ευγενικά πέριψαν αυτή την πρότασή μας. Εμείς εξακολουθούμε να προσκαλούμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε μαζί μας για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο πολυμερές εργαλείο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι υπάρχουν τελικά πάρα πολλά κράτη-μέλη που θα ήθελαν μια τέτοια πολυμερή ευρωπαϊκή συμφωνία με, τα, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, στα πλαίσια του γαλλικού αυτού ντοκιμαντέρ είδαμε και τον Γαλλικό Σύλλογο Αμερικανών Λόγω Συγκυριών, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας της Γαλλίας προκειμένου να στραφούν κατά του ΦΑΤΚΑ. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένω να πρέπει όντω να περάσουμε από τέτοιε εθνικέ προσφυγέ πρωτού καταλήξουμε τελικά σε ένα αποτέλεσμα. Πάντω, ε, εμεί είμαστε σε θέση, εφόσον έχουμε στοιχεία μη συμμόρφωση, να αναλάβουμε δράση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι ε, και για μας το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και μέσω των αναφορών αλλά και μέσω των μεμονωμένων Αμερικανών λόγω συγκυριών οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με εμά τους Ευρωβουλευτές λέγοντά μα ότι θα πρέπει να επιληφθούμε του ζητήματο επιγόντω. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που οι συντονιστέ αποφάσισαν να υποβάλουν προφορική ερώτηση όχι μόνο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και προ το Συμβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και έρθε την κατάλληλη στιγμή και ελπίζω ότι τι επόμενε μέρε θα δούμε μία διοργανική πλέον προσέγγιση για το ζήτημα. Πρέπει από κοινού να εργαστούμε άλλωστε, προκειμένου να έχουμε ένα σύστημα πιο ανθεκτικό, το οποίο θα δημιουργεί παρέκκληση, εξαίρεση για τους ανθρώπους αυτούς που, ας μην το ξεχνάμε, είναι Ευρωπαίοι πολίτες ουσιαστικά και απλώς έτυχε να γεννηθούν μια Τετάρτη Ιουλίου. Φαντάζομαι βέβαια ότι ε, υπάρχουν και κάποιοι Ευρωπαίοι που θα ήθελαν να είχαν γεννηθεί μια Τετάρτη Ιουλίου στι ΗΠΑ για άλλου πάλι λόγους, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία, στην αφήσουμε τώρα. Επανερχόμενοι στη σημερινή αναφορά, Κύριε καθηγητά, θεωρώ ότι μας δώσατε πολλές πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό που πρέπει εμείς τώρα να κάνουμε είναι ως μέλη της Επιτροπής αυτής να εγκρίνουμε το σχέδιο ψηφίσματος και το προφορικό ερώτημα. Μπορείτε να πάρετε λοιπόν τώρα το λόγο ή διαφορετικά μπορούμε να ψηφίσουμε ευθύ αμέσω. Να σας πω ότι η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο ψηφίσματος είναι 23η Μαΐου, 3 το μεσημέρι. Είδατε να βάλαμε τη ημερομηνία, σας δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να εξετάσετε το ζήτημα. Δεν βλέπω να θέλει κανείς όμως το λόγο, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε για το προφορικό ερώτημα, αν γκρίνετε το κείμενο. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ, Ποιο είναι υπέρ του προτινόμενου κειμένου, πολύ ωραία. Όλοι, ομόφωνα υπέρ, ομόφωνα υπέρ, καταπληκτικά, άψογα. Λοιπόν, θα προωθήσουμε το προφορικό αυτό ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στην όλη συζήτηση και κύριε Γκαρμπαρίνο, κύριε καθηγητά, εσάς όλους ιδιαίτερος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη αυτή παρέμβασή σας. Μη σας προξενήσει έκπληξη αν σας καλέσουμε πάλι σύντομα στο μέλλον για να μας βοηθήσετε με το ζήτημα αυτό. Ναι βέβαια, μπορείτε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν θέλω να αντιδράσω, γιατί είπε πολύ λογικά πράγματα η Κομισιόν. Ή μάλλον γρήγορα, γρήγορα να πω δύο πράγματα, ότι είναι φυσικά και θα πρέπει κατά περίπτωση να ερευνούμε και να δούμε σε κάθε συμφωνία κατά πόσον ε, τηρείται η αρχή της αμοιβαιότητας ή όχι. Χρειάζεται δηλαδή εμπειρική ανάλυση. Υπάρχει ωστόσο η εξή στάση. Η εξη ταση η αμοιβαιοτητα ε, έχει γίνει ουσιαστικά μονομέρεια από τη ΣΥΠΑ. Και το άλλο είναι ότι φυσικά αυτή η accidental Americans, οι αποσπόντα Αμερικάνοι είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο. Είπα είναι η μόνη χώρα που φορολογεί το παγκόσμιο εισόδημα και πραγματικά αυτό προκαλεί κατακραυγή και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς φορολογικές πρακτικές. Σίγουρα, αν ένας κάτοικος, είπα, ε, φοροδιαφεύγει, φυσικά και θα πρέπει να ζητούνται πληροφορίες από τις τράπεζες. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησα να μελετώ το θέμα των Accidental Americans, αλλά είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων σε ό,τι αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Εγώ έχω ανησυχίες με αυτή την ανταλλαγή, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμη και αν είναι φορολογικά τα στοιχεία. Είναι πολύ καινούριο αυτό ο κανονισμό, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα τα ξανασυζητήσουμε. Αυτά είχα να πω. very few days to come θα έχουμε τη νέα πραγματικότητα σε λίγε ημέρε με τη θέση σε ισχύ του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Πράγματι. Ωραία, λοιπόν, αφήνουμε προ το παρόν το θέμα και θα το ξαναπιάσουμε την επόμενη φορά. Πότε θα είναι? 19 Ιουλίου. Οπότε και θα ψηφίσουμε. Το ψήφισμα και τις τροπολογίε. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά και Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το παρθμόν 16, προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και την αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέταση και έγκριση σχεδίου προφορικής ερώτησης. Το ιστορικό το γνωρίζετε, μας απασχολεί εδώ και καιρό το ζήτημα. Έχουμε μαζί μας όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κριστίνα Κάνιγχαμ συγκεκριμένα, όχι. Πού είστε? Α, πάρα πολύ ωραία. Τώρα σας βλέπω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό της μερικής διάταξης, νομίζω ότι είναι σαφές πως η παρέμβαση μου σήμερα είναι αμυγός διαδικαστικού χαρακτήρα. Σήμερα το μόνο που μπορώ να κάνω ουσιαστικά είναι να επαναλάβω αυτό που είπα και την τελευταία φορά που είχα τη χαρά να βρίσκομαι εδώ, στην Επιτροπή Αναφορών. Δηλαδή, πρώτον, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία την επίκαιρη για την αναφορά αυτή που ουσιαστικά είναι η βάση, το θεμέλιο της προφορικής ερώτησης που υποβάλλεται στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και σε ό,τι αφορά τις συστάσεις που συνδέονται με έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρεται στην προφορική ερώτηση η Επιτροπή Αναφορών, αυτό θα εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα. Αναβλήθηκε για μια εβδομάδα η έγκριση. Θα εγκριθεί λοιπόν στις 22 Μαΐου. Εν συνεχεία, θα είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για μια ανταλλαγή απόψεων και μια συζήτηση για τα ζητήματα που συμπεριλάβατε σε αυτή την προφορική ερώτηση. Και που φαντάζομαι ότι θα εγκρίνετε και όλα σας στην σημερινή σας ψηφοφορία. σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιο συνάδελφο το λόγο, κύριε Μαλίνοφ, ίσω, όχι. Κύριε Μαλίνοφ. Πρέπει να πω ένα ευχαριστώ για όλους τους συναδέλφους, γιατί νομίζω ήταν μια από τις πιο καλές συζητήσεις αυτή που είχαμε για το θέμα αυτό. Και εν συντομία θα μπορούσα ίσως να επαναλάβω κάποια επιχείρηματα. Το γεγονός ότι προχωρούμε μαζί με την Επιτροπή Καλτ δείχνει ότι υπάρχει αλληλεγγύη και υπάρχει βαθιά κατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των επιτροπών. Για ένα πρόβλημα αναγνωρισμένο ως ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Θα έχουμε συζήτηση στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι μικρότερες γλώσσες αξίζουν να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια, σε αυτό το, ευρύτερο φόρουμ συζήτησης. Δεν έχω να προσθέσω κάτι νέο. Απλά κάποιες φορές όταν λέμε ότι κάτι είναι επίκαιρο, εδώ ισχύει ε, κυριολεκτικά όρος. Γιατί έχουμε αυτές τις νέες προτάσεις και νέες ιδέες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω από την ε, Βουλγαρική Προεδρία. Περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τι προτάσεις. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρο. άρα ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε και μπορούμε να προχωρήσουμε στην έγκριση του σχεδίου προφορικής ερώτηση. Ε, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όλοι ήσασταν υπέρ. Ωραία. επομένω. έγινε δεκτή το σχέδιο προ αλλά δεν τελείωσε το θέμα. Θα πρέπει τώρα να συνεχίσετε εσεί να ασκείτε πιέσει στι πολιτικέ σα πολιτικές να ενημερώσετε του επικεφαλεί των πολιτικών σα ομάδων, διότι τώρα το θέμα αυτό θα πάει στη διάσκεψη των Προέδρων που θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια. Και εγώ νύπτω τα σχήρα μου από το σημείο αυτό και μετά. Λοιπόν, για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Πάντως ομοφόνος εγκρίθηκε αυτή η προφορική ερώτηση και αυτό πάντοτε είναι ένα καλό επιχείρημα το οποίο μπορείτε και εσείς να χρησιμοποιήσετε στις συζητήσεις που θα έχετε με τους επικεφαλής των πολιτικών σας ομάδων εξαιρετικά. Να παρακαλέσω να καθίσετε όσοι δεν είστε στις θέσεις σας και να μιλάτε και λίγο χαμηλόφωνα παρακαλώ και το προσωπικό να μιλάει πιο σιγά Αναφορά αριθμός 1086. Το σημείο 17. Είναι η αναφορά εξ του Δήμου Δωρίδα σχετικά με τι επιπτώσει λειτουργία του φράγματο και τη τεχνητή λίμνη του Μόρνου στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Μόρνο, αλλά φαντάζομαι ότι ε, θα μα ε, διαφωτίσουν ε, οι παριστάμενοι. Δεν είναι εδώ όμω οι Να ηρεμήσουν ε, ε, όσοι είναι όρθιοι και μιλάνε. Για 30 λεπτά, ε, συγγνώμη, δευτερόλεπτα διακόπτω. 30 δευτερόλεπτα. We are a little bit ahead. Είμαστε μπροστά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, σε ό,τι αφορά τη μεσιά διάταξη. Εκμεταλλεύτηκα με το χρόνο τα πάρα πολύ επιτυχημένα. Δεν ξέρω αν ήρθαν αναφέροντες και που είναι. Α, εκεί, μάλιστα. Είστε εδώ κύριε Καπεντζόνη. Ωραία, πολύ καλά. Καλώς ορίσατε θερμά Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά για να μας εξηγήσετε την κατάσταση και να μας δείξετε και πού στο χάρτη βρίσκεται ο Μόρνος ή δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του, της Επιτροπής Αναφορών και γιατί έγινε δεκτό, παραδεκτό το αίτημά μας να συζητηθεί και γιατί ε, μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να αναπτύξουμε τις θέσεις μας από κοντά. Είμαστε ο Δήμος Δωρίδος, είμαστε στην κεντρική Ελλάδα, έχουμε έδρα το Λιδωρίκι, το οποίο απέχει από την Αθήνα 245 χιλιόμετρα. Στην περιοχή μας, στην κεντρική Ελλάδα, τέλος της δεκαετίας του 60, φτιάχτηκε ένα μεγάλο φράγμα στον ποταμό Μόρνο, δημιουργώντας την τεχνητή λίμνη του ποταμού Μόρνου, το οποίο λειτουργεί ως ταμιευτήρας πόσιμου νερού για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα και την περιοχή της στην ευρύτερη. Ένα φράγμα χωρητικότητας πάνω από 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και με ένα δίκτυο αγωγών μεταφέρεται νερό από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι την Αθήνα για την ίδρυυση της ευρύτερης περιοχής. Αργότερα χρειάστηκε να γίνει ακόμα ένα φράγμα στο γειτονικό ποταμό, στον ποταμό Εύινο, στη Δυτική Ελλάδα, για τον ίδιο λόγο και έτσι έχουν καλυφθεί πλήρω οι ανάγκε τη ε, περιοχής τη αθηνα Αθήνας, πάνω από 5-6 εκατομμύρια πληθυσμό ε, οι κάτοικοι ε, και έχει λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Αυτό το δίκτυο αγωγών μεταφέρει πάνω από 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίω στην Αθήνα. Ένα έργο πνοή λοιπόν για την ε, χώρα μας έχει καταστεί γάγκρενα, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη δικιά μας περιοχή και το πρώτο πρόβλημα που είναι είναι γιατί κατασκευάστηκε το έργο την δεκαετία του, τέλος της δεκαετίας του 1960 όπου στην Ελλάδα είχαμε δικτατορικό καθεστώς και ακόμα δεν υπήρχε περιβαλλοντική νομοθεσία και δεν έχει εφαρμοστεί καμία περιβαλλοντική νομοθεσία και για, την, ε, για το έδος εκτέλεσης αλλά και στη συνέχεια. Μια σειρά οδηγιών που έχουν εκδοθεί και από την ε, Ευρώπη στα επόμενα χρόνια δεν έχουν εφαρμοστεί. Αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο. Το μεγαλύτερο ζητούμενο για μας είναι ότι πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή και έχουν να κάνουν, με συντομία θα σας τα περιγράψω, τα έχετε δει στην αναφορά σας, με την αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των οικισμών του Δήμου μας και της έδρας του, Λιδωρίκη, τα οποία οι αποστάσει αυτέ έχουν μεγαλώσει δραματικά, αυξάνοντα το κόστο ζωή. Από έναν οικισμό, λοιπόν, παράδειγμα το Κάλιο, που η απόσταση είναι περίπου στα ήταν στα 7 χιλιόμετρα, η απόσταση έγινε 17 και ο χρόνος μετακίνηση πολλαπλασιάστηκε. Τέτοια προβλήματα έχουμε σε πάρα πολλού οικισμού και έτσι το κόστο ζωή έχει αυξηθεί δραματικά. Άλλο πρόβλημα μεγάλο που έχει δημιουργηθεί, τα λέω επιγραμματικά, είναι ένα καθεστώ προστασία, απόλυτη προστασία γύρω από τη λίμνη, η γκρι ζώνη που βλέπετε, 1500 μέτρα σε οριζόντια απόσταση που καθιστά αδύνατη την οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή. Ούτε τουρισμός, ούτε κολύμπι, ούτε ε, γεωργικέ καλλιέργειες, ούτε κτηνοτροφία, οτιδήποτε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί. Ένα άλλο πρόβλημα πολύ μεγάλο είναι η... το ότι οι κτηνοτροφικέ μονάδε όσε ήταν ανοιχτέ και αυτέ οδηγούνται σε μαρασμό. Επίση, από τον ε, ταμιευτήρα γύρω στη... μέσα στη ζώνη αυτή των 1500 ε, μέτρων δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να κατασκευάσουμε έναν βιολογικό καθαρισμό που έπρεπε να υπάρχει από τι αρχέ των, ε, της κατασκευής του φράγματος και ένα βιολογικό που θα πήγαινε τα λίματα από το λιδωρίκι στον ποταμό, τα επεξεργασμένα, ένα χιλιόμετρο απόσταση, χρειάζεται πλέον να κάνει 30 χιλιόμετρα απόσταση διάνυση τα επεξεργασμένα λίματα και αυτό καθιστά το έργο ανέφικτο, πολυδάπανο και δεν έχει κατασκευαστεί από τότε μέχρι σήμερα. Και δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε ως αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν και αυτή μια δραματική συνέπεια για την περιοχή μας, όπως επίσης δραματική συνέπεια για την περιοχή μας είναι και προκαλεί το, το γεγονός ότι δεν έχει κατασκευαστεί ποτέ οικολογική παροχή. Η οικολογική παροχή είναι ποσοστό ύδατος που πρέπει στις περιπτώσεις που φράζονται τα ποτάμια ένα ποσοστό ύδατος να κατεβαίνει κάτω από το φράγμα, κατάντι του φράγματος για την συνέχιση της ζωής, για την συνέχιση για την χλωρίδα και την πανίδα και το ανθρωπογενές περιβάλλον κάτω από το φράγμα. Γίνεται, συμβαίνει σε όλα τα φράγματα στον κόσμο εκτός από τη δικιά μας περιοχή. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλες συνέπειες για το ποτάμι από το φράγμα και μέχρι τη θάλασσα και για τη γεωργία και για την κτηνοτροφία και τα, τα αλλιεύματα έχουν μηδενιστεί και όλες αυτές οι δραστηριότητες πλέον έχουν μηδενιστεί. Ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια δημιουργεί, πρόβλημα μας δημιουργεί το ότι αφού είναι το ποτάμι 5, 6, 7 μήνες το χρόνο χωρίς νερό δεν κατεβαίνουν φερτά υλικά, δεν έρχεται υλικό από το βουνό όπως κάνουν όλα τα ποτάμια, με αποτέλεσμα να υπερισχύει η διάβρωση της θάλασσας στην εκβολή και το μέτωπο, το παραλιακό μας μέτωπο υποχωρεί κατά ένα μέτρο σύμφωνα με μελέτη που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε χρόνο. Χάνουμε τις παραλίες μας και υπάρχουν χαρακτηριστικές εικόνες που θα δείτε. Εδώ 40 μέτρα παραλία υπήρχε σε αυτό το σημείο και τώρα έχουν μείνει ούτε 10 μέτρα. Και αυτό θα το πάθουμε πολύ πιο έντονα στην μεγαλύτερη παραλία του Δήμου μα που είναι ακριβώ δίπλα, στα 2 χιλιόμετρα, που είναι η παραλία τη Χιλιαδού, το πιο τουριστικό μα κομμάτι. Θα το πάθει αυτό που είδατε στην προηγούμενη εικόνα και η Χιλιαδού που βλέπετε εκεί. Είναι λοιπόν μια σειρά προβλημάτων και δεν θα αναφερθώ ε, κλείνοντα από μια κουβέντα για τον αρχαιολογικό χώρο τη αρχαία Καλύπολη, μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη, που έχουμε και μια ευαισθησία εκεί. Όταν έγινε το φράγμα δεν λήφθηκε καμία μέρημνα ούτε για την προστασία του χώρου, ούτε για την ανάδειξη και το σχετικό μουσείο, αρχαιολογικό μουσείο που έχουμε στο Λιδωρίκι δεν έχει κανένα από τα ευρήματα. Α, όλα αυτά γιατί τα λέω, τα λέω γιατί είναι ξεκάθαρο η χώρα μας έλυσε το πρόβλημα ίδρυυσης της πρωτεύουσας και καλά έκανε. Δεν λήφθηκε καμία μέρημνα και καμία υποδομή δεν έγινε και ένα μέτρο δεν λήφθηκε για το ανθρωπογενές περιβάλλον, για το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μας όλα αυτά τα χρόνια. Και θα μπορούσε να έχουν ληφθεί μέτρα, να έχουν γίνει έργα αποκατάστασης αυτών των προβλημάτων, θα μπορούσε να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα μέσω της αυτοδιοίκησης να μπορούν χρόνο με το χρόνο να λύνονται αυτά τα προβλήματα και αυτό είναι που ζητάμε συν το ότι θέλουμε από την ελληνική κυβέρνηση να υπάρξει ένας διάλογος και να καταφέρουμε στο τέλος να, κάνουμε, να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι χρονίζοντα και πάρα πολύ μεγάλα. Κύριε Ευρωβουλευτές, ένα έργο ζωής για τη χώρα μου κατέστη καταστροφή, υποβάθμιση και μαρασμός και υπανάπτυξη για τον τόπο μας, για το Δήμο μας με παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς καμία συνένεση, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς κανένα κίνητρο και κανένα αντιστάθμισμα, δεν λύθηκε ποτέ καμία μέρημνα. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, ιδιαίτερο καθεστώς Τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερο καθεστώ, ιδιαίτερε συνθήκε από ό,τι είδατε στην περιοχή μα, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Θέλουμε ένα θετικό σήμα από εσά και από την Επιτροπή σα και τη διαβίβαση και σε άλλα ενδεχομένω αρμόδια όργανα που εξειδικεύονται περισσότερο για αυτά τα ζητήματα, αν μπορεί να γίνει, και ένα θετικό σήμα προ την ελληνική κυβέρνηση μαζί με την αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα. Δεν θεωρούμε σωστό σε καμία περίπτωση ο Δήμος, η περιοχή της χώρας που δίνει το πολυτιμότερο αγαθό που χρειάζεται το 60% περίπου του πληθυσμού της χώρας μας να έχει καταστεί ο πιο φτωχός, ο πιο ταλαιπωρημένος Δήμος στη χώρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και ζητούμε την αρρωγή σας. Thank you very much. And... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για όλες τις εξηγήσεις. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Είμαι σίγουρη ότι θα θελήσουν οι συναδελφοί να κάνουν ερωτήσει Να ακούσουμε και του εκπροσώπους τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, προχωρήσουμε στην ανταλλαγή απόψεων με του συναδέλφου. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω αρχικά ότι πολύ σύντομα θα στείλουμε στην Επιτροπή σας μια γραπτή απάντηση με όλες τις αξιολογήσει αυτού του φακέλου. Αλλά αφού είμαι μαζί σας σήμερα, με μεγάλη μου χαρά, να σας παρουσιάσω προφορικά τη θέση μας. Για αυτή την αναφορά πρέπει να διακρίνουμε δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο αφορά την άδεια λειτουργίας του έργου και το δεύτερο τη λειτουργία του. Και οποιασδήποτε πιθανές τροποποίησεις μπορεί να γίνουν στο μέλλον. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, όπως υπογράμισε ο αναφερόμενος, το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε πριν ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, δυστυχώς, όσον αφορά την αδειοδότηση αυτού του έργου, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για οποιαδήποτε παραβίαση. Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, και εκεί είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της αναφοράς, ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το ίδιο το έργο, αν είχε μόλις τροποποιηθεί τώρα ή αν τροποποιηθεί μέσα σε λίγα χρόνια και αν αυτή η τροποποίηση είναι σημαντική, αν δημιουργηθεί ένας δεύτερος αμοιβήρα ή ένα μικρό πράγμα σε περίπτωση σίγουρα ε, ισχύει η ευρωπαϊκή σιγουρα ισχυει η ευρωπαικη νομοθεσια και σε τέτοια περίπτωση πράγματι θα πρέπει να γίνει μία μελέτη ε, αντικτύπου περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι η αξιολόγηση αυτή δεν θα αφορά μόνο το νέο έργο, τη νέα προσθήκη ή το νέο στοιχείο, αλλά το σύνολο του έργου. Το πώ δηλαδή ολόκληρο το έργο, ε, τι επιπτώσει έχει στο περιβάλλον, στη χλωρίδα, στην πανίδα, στην ανθρωπινή υγεία κτλ. κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να το θυμόμαστε σε περίπτωση τροποποίηση του έργου. Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται αν δεν υπάρξει τροποποίηση, αν δεν επέλθει τροποποίηση θα συνεχίσουν οι ντόπιοι να υφίστανται τις συνέπειες του έργου αυτού και για πόσο καιρό. Ένα κομμάτι της απάντησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε πίεση από, ως Κομισιόν αφού δεν έχουμε παραβίαση της νομοθεσίας. Η πίεση αυτή θα μπορούσε να βασιστεί στην οδηγία 2060 για τα ύδατα. Να σας επιβεβαιώσω ότι το σχέδιο διαχείρισης υδρογραφικών ε, περιοχών. Μιλάμε για το σχέδιο ε, για την κεντρική δυτική και δυτική Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2014. Το εν λόγω σχέδιο περιλάμβανε αυτό το φράγμα. Το σχέδιο αυτό μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής θεωρήθηκε ότι δεν ε, τηρούσε τι υποχρεώσει τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μετά από αυτό το πρώτο σχέδιο, λοιπόν, η Ελλάδα, και αυτό πάλι αποτελεί μια υποχρέωση που απορρέει από την οδηγία για, πλαίσιο για τα ύδατα, άλλαξε όλα τα σχέδια περιοχών και τα σχέδια διαχείριση η Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου τη Κεντρική Ελλάδα. Το νέο σχέδιο λοιπόν εγκρίθηκε από τις ελληνικές αρχές και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 29 Δεκεμβρίου του 2017. Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την υιοθέτηση αυτού του νέου σχεδίου και τώρα ε, συγκεντρώνει όλα τα τεχνικά στοιχεία, δηλαδή όλα τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, τις αλληλεπιδράσεις κτλ. Δεν έχουμε ακόμα λάβει όλα τα στοιχεία. Μόλις πραγματοποιηθεί αυτό, ε, μιλάμε για μερικές εβδομάδες, το πολύ ελπίζω, μόλις ολοκληρωθεί η παραλαβή θα αναλύσει η Κομισιόν όλα τα σχέδια των υδρογραφικών περιοχών που σχετίζονται με αυτή την αναφορά προφανώς, ώστε να δούμε αν η Ελλάδα έχει λάβει υπόψη τις συστάσεις της Κομισιόν που είχαν υποβληθεί μετά από την αξιολόγηση του πρώτου σχεδίου. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας παρέχει μια δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στην Ελλάδα και φυσικά θα ήθελα να αναφέρω και το σχέδιο του κύριου Αναφερομένου. Θα το αναφέρω ώστε οι συνάδελφοι που θα ασχοληθούν με την Δυτική και Κεντρική Ελλάδα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το έργο. Ελπίζω λοιπόν ότι τα σημεία του αναφερόμενου θα μπορέσουν να εξεταστούν πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι αφού δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε άμεση παραβίαση της ε, Ευρωπαϊκής Δομοθεσίας, αυτό το έργο χρονολογείται πριν από την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε όλες τις οδούς προσφυγής που έχουμε σε εσωτερικό επίπεδο και με μια εκτίμηση αντικτύπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που διευκρινίσατε κάποια πράγματα και κάποια τουλάχιστον δικά μου ερωτηματικά έχουν απαντηθεί. Τώρα έχουμε τη συζήτηση και πρώτο κύριο Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω την ομιλία μου φορώντας τα γυαλιά γιατί έχω ένα πρόβλημα από το πρωί οφθαλμολογικό γι' αυτό και δεν μπόρεσα να ε, συμμετάσχω στην Επιτροπή, δεν έφυγα ξαφνικά και θα με συγχωρέσετε αν τελειώντας την ομιλία μου φύγω πάλι γιατί πρέπει να ε, συνεχιστεί η ιατρική παρακολούθηση. Ε, είναι μια σοβαρή υπόθεση και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι πραγματικά συζητείται σήμερα η αναφορά. Με τους αναφέροντες και κυρίως τον Δήμαρχο Δωρίδος συζητήσαμε από την αρχή την περίπτωση να έρθει αυτή η υπόθεση εδώ ως αναφορά κουβεντιάσαμε πραγματικά τους βοήθησα και στην διαμόρφωση της ίδιας της ε, πετησιών. Ε, ήρθαν εδώ, την κατέθεσαν και όπως γνωρίζετε μετά από πρόταση δική μου εκπροσωπώντας το ECR ζητήσαμε εκτάκτως να συζητηθεί σήμερα κατά την ε, διαδικασία που έχει δικαίωμα κάθε πολιτική ομάδα να ζητήσει κάποιες υποθέσεις, κάποιες αναφορές να προηγηθούν. Θεωρώ λοιπόν σημαντική την συζήτηση. Νομίζω ότι με τον τρόπο που παρουσίασαν οι αναφέροντες ε, τα αιτήματά τους ήταν ξεκάθαρα τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Ε, νομίζω ότι και η Επιτροπή Κομισιών ε, έθεσε πραγματικά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του νέου τρόπου διαχείρισης των υδάτων και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η περίπτωση της ε, αναφοράς. Επομένως ε, θεωρώ ότι τα ζητήματα έχουν τεθεί με σαφή τρόπο, έχουμε παραβίαση της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οτιδήποτε νέο έργο γίνει και πρέπει να γίνει νέο έργο στην περιοχή πρέπει μετά να συνδυάσει τον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του συνολικού έργου και έτσι όπως λειτουργεί. υπάρχουν οι παράπλευρες προβληματικές περιπτώσεις, δηλαδή το ότι χτυπιέται η ίδια ανάπτυξη της οικονομίας στην περιοχή, απομονώνονται ολόκληρες περιοχές, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μας απαιτείται η προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως δε ότι χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα απορροής των υδάτων, δηλαδή να συνεχίσει το ποτάμι να τρέχει, ούτως ώστε να μπορεί να έχουμε ε, τα αποτελέσματα που φέρνει η ίδια η φύση, δηλαδή να μην, να μην εξαφανιστούν οι ίδιες οι ακτές, να συνεχιστεί η ζωή από το φράγμα μέχρι ε, εκεί που εκβάλλουν τα, τα ύδατα. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει, είναι βάσιμη αναφορά, έχουμε πλήρη παραβίαση των δικαιωμάτων και του Δήμου και των πολιτών, χρειάζεται προστασία της περιοχής, χρειάζεται εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η Κομισιόν έχει ήδη ανοίξει το φάκελο και στη βάση αυτή νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την έρευνα και τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σοφία, κυρία Σακοράφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ε, θέλω να πω ότι το θέμα όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Δήμαρχο και παρουσιάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ αναλυτικά για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι αλλά και όλοι εμείς και που βρίσκεται το έργο και τη σημαντικότητα του έργου αλλά και την καταστροφή που δημιουργεί στη ζωή των ε, κατοίκων της ε, περιοχής είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιβεβαιώνει θα έλεγα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, την ορθή κατεύθυνση που κινήθηκε θα έλεγα όλο το περιβαλλοντικό κίνημα όσον αφορά τις οδηγίες, να πετύχει οδηγίες, τις συγκεκριμένες που επικαλείται ο κύριος Δήμαρχος σήμερα εδώ, στην αναγκαιότητα να πιέσει για να τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης το γεγονός ότι αυτό το έργο παρότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη την Αττική γιατί όπως είπαμε ιδρεύει ένα τεράστιο μέρος ε, την ίδια στιγμή δημιουργεί και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Το ερώτημα για μένα που μπαίνει είναι ποιες θεραπείες, γιατί περί αυτών πρόκειται και για, αυτά θα πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, ποιες θεραπείες μπορούν να ληφθούν και να δρομολογηθούν για ένα έργο που έχει γίνει προθύστερα. Υπόθηκε και από τον κύριο Δήμαρχο ότι έγινε το 1960. 68-69. Εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ πίσω, πολύ πριν ε, ε, ξεκινήσει η διαδικασία αυτή με τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Ε, θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι το έργο έγινε τόσο παλιά, δεν μπορούμε σήμερα να επικαλυστούμε ακριβώ επειδή έγινε το έργο τότε ότι ό,τι έγινε έγινε, ό,τι κακό έγινε στην περιοχή να το αφήσουμε έτσι. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε και τον Δήμο να ορθοποδήσει και οικονομικά αλλά και του πολίτε να μην αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί, ότι έχουν καταστραφεί περιουσίε του ε, και όλα αυτά. Ε, θέλω να, να παρακαλέσω τον κύριο Δήμα. Καταρχήν θα ήθελα να παρακαλέσω κυρία Πρόεδρε να μείνει ανοιχτή η υπόθεση, ε, το θέμα, ε, και έτσι όπως το ανέφερε και η Επιτροπή, διότι η Επιτροπή έχει ένα φάκελο αυτή τη στιγμή τον οποίο δεν τον έχει ελέγξει. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή να ελέγξει το φάκελο και να μας τον φέρει ολοκληρωμένο να το συζητήσουμε εδώ. Να μείνει λοιπόν ανοιχτή η επιστολή. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα στον κύριο ότι θα ήθελα και θα παρακαλούσε αν είναι δυνατόν, επειδή ακριβώς μίλησε για αντισταθμιστικά ωφέλη, εάν μπορεί να περιγράψει με κάποιον τρόπο αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη και πώς, τα, πώς τα βλέπει εκείνος, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Λέω ένα παράδειγμα κύριε Δήμαρχε, επειδή όντως εκεί πέρα είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ έφορη, πολίτες έχουν χάσει τα χωράφια τους ας πούμε είχατε ποτέ βοήθεια ή θα θέλατε βοήθεια που θα μπορούσε η Επιτροπή να πιέσει και την κυβέρνηση στην ελληνική ε, να κατευθύνει τους πολίτες προ καλλιέργειες οι οποίες δεν μολύνουν το περιβάλλον, λέω ένα παράδειγμα. Ή πώς βλέπετε εσεί το γεγονό ότι ε, ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή οι πολίτες ε, μεταφέροντα τα, τα και οι ίδιοι μεταφερόμενοι δηλαδή και τα, την περιουσία τους τόσα χιλιόμετρα κάνοντα αποστάσει οι οποίε έχουν δημιουργηθεί. Αυτό θα μπορούσατε να μα το περιγράψετε, γιατί για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κύριε ε, Πρόεδρε, επίση, ε, ξαναεπαναλαμβάνω ότι θα πρέπει η, υπόθεση να παραμείνει ανοιχτή. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτερ Γιάρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες ε, που ήρθαν ε, στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα σχεδόν ε, θα ασκούσα κριτική στην Κομισιόν γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια απάντηση. Βέβαια η προφορική απάντηση μου άρεσε, ήταν καλά δομημένη και επομένως ε, αποσύρω την κριτική που θα ασκούσα εφόσον υπάρχει η καλή αυτή προφορική απάντηση. Φοβόμουν να πω α, ε, ότι θα άκουγα από την Κομισιόν τι να σας κάνω, κακοτυχία είχατε, ατυχήσατε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει και τα σχετικά στοιχεία και θα παρακολουθήσουμε σίγουρα και εμείς ε, το θέμα και πράγματι δεν υπήρχε περιβαλλοντική διαχείριση ή περιβαλλοντική αξιολόγηση τότε ανεγέρθη το έργο και αυτό ήταν. Ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές κατά πόσον υπάρχει ε, μια τέτοια μελέτη ή θα μπορούσε να γίνει ε, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το ότι το πόσιμο νερό φτάνει στην πρωτεύουσα στην προκειμένη περίπτωση αλλά είναι πολύ κακά τα ε, όσα υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής. Και αυτό πρέπει επίσης να το λάβουμε υπόψη. Και το τρίτο σημείο, από ό,τι φαίνεται, ε, δεν φαίνεται να ε, υπάρχει διάλογος με τις ελληνικές αρχές και την ελληνική κυβέρνηση γιατί τα προβλήματα που μας μετέφερε ο Δήμαρχος φαίνεται πλέον ότι είναι γνωστά, άρα δεν υπάρχει ίσως ε, λόγος ε, ε, η αφορμή να γίνει μια νέα συζήτηση με την κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθούν και οι περιβαλλοντικές πτυχές, διαχείριση υδάτων, αλλά να συμπληθούν επαναλαμβάνω και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και αν ε, είμαι σωστά ενημερωμένο, ε, θα επιληφθεί και η Επιτροπή Περιβάλλοντο ε, για τη συγκεκριμένη αναφορά. Εγώ λοιπόν θα ζητήσω επίση να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και ελπίζω να υπάρξει και ένα επικοδομητικός διάλογος στην Ελλάδα για το θέμα αυτό πλέον. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, ενώ ωφελούνται κάποιοι άλλοι που παίρνουν το πόσιμο νερό. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει τώρα να ξαναδώσουμε πάλι το λόγο στον Δήμαρχο, τον κύριο Καπετζόνη. Θα θέλετε να ξαναπάρτε το λόγο κύριε Δήμαρχε και ενδεχομένω να απαντήσετε γρήγορα στα όσα μόλι υπόθηκαν. Ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, στο πρώτο θέμα της ε, Κομισιόν να απαντήσει η τεχνική μας σύμβουλος η κυρία συνεργάτη μας, η κυρία Μορελάτου. Σε σχέση με την απάντηση της ε, Κομισιόν θα θέλαμε να σημειώσουμε δύο σημεία. Το πρώτο που ανέφερε είναι ότι λόγω παλαιότητα του έργου δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όμω το ελληνικό κράτο επιχείρησε να βγάλει περιβαλλοντική αδειοδότηση για το έργο το 1993, όταν στην Ελλάδα με την πολύ μεγάλη ξηρασία χρειάστηκε να προσθεθεί ακόμη ένα φράγμα για να μπορέσει να δοθεί περισσότερο νερό στο φράγμα για το οποίο συζητάμε. Στην αδειοδότηση αυτή όμω αδειοδότησε περιβαλλοντικά μόνο το πολύ πολύ μικρό έργο ενώ και η ίδια η Επιτροπή μας είπε ότι θα έπρεπε να ειδωθεί συνολικά τόσο σύμφωνα με την Οδηγία 85337 όσο και με την Οδηγία 2001 κάθετο 42. Μιλάμε για έργο με απόσταση 200 χιλιόμετρα και δύο με τους μεγαλύτερους ταμιευτήρες της Ευρώπης. Σε σχέση με τη δεύτερη, το δεύτερο τεχνικό σκέλος που απάντησε η Επιτροπή πράγματι, τα σχέδια λεκανών απορροής στην Ελλάδα εγκρίθηκαν το 2014 και το συγκεκριμένο απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναδιορθώθηκε και υποβλήθηκε το 2017. Το εξετάσαμε τεχνικά ιδιαίτερα προσεκτικά και θα θέλαμε να σας πούμε και να καταθέσουμε ότι το σχέδιο αυτό είναι όμοιο με αυτό του 2014 και καμία από τις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν το έκανε δεκτό δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε για δύο λεπτά να δώσω απαντήσεις στην κυρία Σακοράφα και στον κύριο Γιάρης, αν είναι εύκολο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Σακοράφα για την παρέμβασή σας και την στήριξή σας. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι διαφορετικά τα ζητήματα όπως αντιληφθήκατε νομίζουμε και οικονομικά και νομικά και κυρίως περιβαλλοντικά θα πρέπει να λυθούν με διαφορετικό τρόπο και από διαφορετικούς φορείς της ελληνική της πολιτείας. Το πρώτο που χρειάζεται και που θέλουμε να γίνει να υπάρχει συνεργασία του κράτους με την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλουμε είναι για παράδειγμα αν έχουν μεγαλώσει πολύ οι αποστάσει, πρέπει να γίνουν κάποιε γέφυρε πάνω στη λίμνη για να μπορούν να μικρούν οι αποστάσει. Εάν έχει νεκρώσει μια περιοχή, να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν να φύγουν οι κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν εκεί να αδειοδοτηθούν, να μεταφερθούν σε κάποια άλλη περιοχή και κάνοντα κάποιε υποδομέ και δίνοντα κάποια κίνητρα θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντο για να μπορέσουμε να, επιτέλου να φτιάξουμε ένα βιολογικό καθαρισμό, άσχετα αν είναι πάρα πολύ δαπανηρό το έργο αυτό, που δεν μπορεί μόνο του ο Δήμο να σηκώσει αυτό το βάρο, γιατί ξαναλέω, τέτοιο βιολογικό με αυτέ τι απαιτήσει δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη ανάγκη να γίνει, μόνο σε εμά υπάρχει, χωριστά δε, που θα έχει και επιπλέον κόστο μεγάλο κόστο στη λειτουργία του. Μετά, άλλο να μεταφέρει στα λίμματα ένα χιλιόμετρο, άλλο 30 χιλιόμετρα μακριά για τα οποία θα χρειάζεται ενέργεια και την οποία θα επιβαρυνόμαστε εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής. Άρα είναι διαφορετικά ζητήματα που θα πρέπει να τα δουν διαφορετικά υπουργεία ενδεχομένω και υπάρχουν λύσεις. Τι θέλω που θέλω να καταλήξω όμως. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν έργα στην, ε, για την διάβρωση στο, ε, στο παραλιακό μέτωπο, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι αδιανόητο, κυρία Πρόεδρε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, τώρα που μιλάμε, άσχετα ποια νομοθεσία ήταν τότε, να υπάρχει φράγμα χωρί οικολογική παροχή. Χωρί ποσότητα νερού να κατεβαίνει κατάλληλη του φράγματος. Όταν αυτό γίνει και πρέπει να γίνει, άσχετα αν εγκρίθηκε το πρώτο σχέδιο ή το δεύτερο και αν ήταν σύνομο ή όχι με την αρχική νομοθεσία, άσχετα από αυτό, πρέπει να γίνει οικολογική παροχή. Όταν θα γίνει οικολογική παροχή, θα πρέπει να αδειοδοτηθεί, όπω είπε και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για όλο το έργο. Είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε αυτό. Όσο θα υπάρχουν αυτέ οι αρνητικέ συνέπειες θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασία για την τοπική κοινωνία. Είναι πολυδιάστατο το πρόβλημα. Και επειδή όταν πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση με οποιοδήποτε τρόπο και έχει ε, ε, ενοχληθεί και στο παρελθόν από αιρετή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τη δεκαετία του 90 προς το τέλος της δεκαετίας του 90 υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις ότι θα δούμε το ένα έργο, το δεύτερο έργο, κάτι άλλο και δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό καταλήγουμε και λέμε ότι αν υπήρχε ένα αντιστάθμισμα, ένα, το ένα χιλιοστό τη αξία του νερού, γιατί πωλείται το νερό αυτό εκεί που πωλείται και όπω πωλείται, δεν παίρνουμε σε αυτή τη διάσταση αυτή τη στιγμή όμω. Το ένα χιλιοστό, αν είχε θεσμοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία, όπω υπάρχουν αντίστοιχα θεσμοθετημένα αντισταθμιστικά τέλη για ανεμογεννήτριε, για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για μεταλλεύματα κλπ. Θα μπορούσε να υπάρχει γι' αυτόν τον φυσικό πόρο που φεύγει από μία περιοχή και πάει σε μία άλλη τέτοιο που θα μας είχε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα η αυτοδιοίκηση από μόνη της γιατί είναι αρμόδια για αυτά τα προβλήματα να είχε τη δυνατότητα να τα έχει λύσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή την παρέμβαση συζητάμε και τώρα. Μπορεί να υπάρξει αυτός ο διάλογος στην Ελλάδα. Θέλουμε την βοήθειά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για, όσον αφορά το, το ερώτημα που είπε ο κ. Γιάρης είναι ακριβώς αυτό που είπα και πριν. Είναι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις. Έχει. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, δεν είναι μόνο νομικά. Έχει μια σειρά προβλημάτων που ξαναλέω μας έχει καταστήσει την πιο ταλαιπωρημένη περιοχή όχι της χώρας μου, της Ευρώπης. Και γι' αυτό είμαστε εδώ ζητώντας τη βοήθειά σας, την παρέμβασή σας στην ολική πολιτεία και ελπίζουμε να συμβάλλετε στο να αρχίσει αυτός ο διάλογος και να αρχίσουμε σιγά σιγά να επιλύουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Yes, we understand. Ναι, απόλυτα πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση και το αναγνωρίζουμε φυσικά. Με μεγάλη απογοήτευση φυσικά. Το 1969, το 1971, όταν ολοκληρώθηκε το φράγμα, η Ελλάδα δεν ήταν μέλος. Ε, εκτίμηση αντικτύπου για το περιβάλλον δεν έγινε. Ήταν ένα μακρινό όνειρο ακόμα. Σήμερα όμως ε, έχει γίνει πραγματικότητα και η καταστροφή είναι πολύ σημαντική και για τους κατοίκους και για το περιβάλλον οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε πιστεύω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι φυσικά να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ξεκινήσουμε μια στενή συνεργασία με την Κομισιόν επί των όσων μόλις ακούσαμε να μας εξηγείτε να ασκήσουμε πίεση στις εθνικές αρχές Το σχέδιο διαχείρισης για την κεντρική και δυτική Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογηθεί. Το σχέδιο του 2014 όπου η Κομισιόν αποφάσισε ότι τα κριτήρια δεν τηρούνταν. Ε, το έχουμε το, αυτό του 2017 θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ θα παρατρύνω την Κομισιόν να έρθει σε επαφή και με εμά να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές απόλυτα γραπτός μόλις θα έχει τις απαραίτητες προφορές στα χέρια της. Μια πλήρης απάντηση, δηλαδή γραπτή. Αυτό θα θέλαμε από την Κομισιόν. Επίσης πιστεύω ότι θα έπρεπε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να καθίσουμε κάτω και να υπογραμμίσουμε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα σε μια επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ελλάδος. Αυτή την οδό προτείνω να ακολουθήσουμε αν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Ναι. Ωραία ούτως και θα πράξουμε. Ευχαριστήσω γιατί ήρθατε σήμερα ε, και σας εύχομαι καλός ο δρόμος πίσω στην, στην όμορφη Ελλάδα. So we move on to the next petition. We... Περνάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά. Πρόκειται για την αναφορά 900 του 2016 για την ανάληψη δράση κατά μια πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου λόγω τη αμφισβήτηση τη κλιματική αλλαγή. Φρίντα Κίνιγκερ, η αναφέρουσα, είναι εδώ. Πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ που θεωρήσατε παραδεκτή τη σημαντική αυτή αναφορά, την οποία υποστηρίζουν πάνω από 700 και πολίτες. Είναι απλά τα γεγονότα. Η ExxonMobil, μία από τι μεγαλύτερε πολυεθνικέ για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ήξερε ήδη από το δεκαετία του για την κλιματική αλλαγή. Αντί να ενημερώσει την κοινή γνώμη και του επενδυτέ, η εταιρεία δαπάνησε εκατομμύρια σε μία εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ήξερε ExxonMobil ότι με τι δραστηριότητέ της επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή, αλλά παραπλανούσε και αποπροσανατόλιζε την κοινή γνώμη για πολλά χρόνια. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν πολλοί γενικοί ε, εισαγγελεί που ερεύνησαν την εκστρατεία, αλλά και επιχείρηση και βέβαια και με την ε, κυβέρνηση Τραμπ ε, ουσιαστικά ε, ανεστάλησαν αυτές οι έρευνες. Είναι γνωστό ότι έχει στενούς δεσμούς με την ExxonMobil η κυβέρνηση Τραμπ και η απόσυρση από την Συμφωνία των Παρισίων που αποφάσισε ο Τραμπ αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο κακό κάνει η σχέση μεταξύ της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και των πέφτουν λήψεις αποφάσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώ για αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιοποιήσει τι ε, ε, ευθύνε του και την αρμοδιότητα που έχει να ζητήσει από την ExxonMobil να λογοδοτήσει για τη δράση τη και να ενημερώσει την κοινή γνώμη για του κινδύνου. Έχει υπογράψει η Ένωση τη Συμφωνία Παρισίων. Θέλει να είναι ηγέτη τη ανώσιμε πηγέ ενέργεια, να προστατεύει του πολίτε. Από την άλλη πλευρά η ExxonMobil έχει καταστροφικό ιστορικό σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική καταστροφή ε, και τον αντίκτυπο στη δημόσια ε, υγεία. Επίση, ε, με τι δραστηριότητε στον τομέα των ορεικτών καυσίμων ε, επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Είναι πέμπτη στον κατάλογο των εκπαιμπόντων ε, αερία του θερμοκηπίου μεταξύ των ιδιωτικών παραγωγών ορεικτών καυσίμων για την περίοδο 88-2015. Είναι σημαντικό λόμπι, μια σημαντική δύναμη λόμπι στην Ευρώπη. Το 2016 θα πάνε σε σχεδόν 5 δι ευρώ για δραστηριότητε άσκηση πίεση και δραστηριοποιείται σε διάφορα κράτη-μέλη στον τομέα των πετροχημών χημικών και φυσικού αερίου πετρελαίου. Πρόκειται για μια σημαντική αναφορά. Ε, η παρουσία μας ε, και η αναφορά μας προστίθεται σε μια μακρά σειρά άλλων αναφορών για την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι αποτέλεσμα ενός κινήματος ισχυρού μεταξύ των Ευρωπαίων που θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον, την υγεία, αλλά και το κλίμα εν γέννη. Οι αιρετοί εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη πρέπει να φροντίσουν δραστηριότητες Exxon Mobil να μην υπονομεύουν ε, τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ε, έχουμε ήδη σχετικέ προσπάθειε με διάφορα νομοθετήματα. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ και αγαπητοί Πρόεδρε τη Επιτροπή Μεταφορών, ε, σα παρακαλούμε να γνωρίσετε τη σημασία τη αναφορά αυτή ε, και να αναλάβετε δράση. Έχουμε δύο προτάσει για πιθανά μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η Επιτροπή. Πρώτον, θα ζητούσαμε να παρακαλέσετε να συμμετάσχει η ExxonMobil σε ακρόαση που θα οργανωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτό για την ακρόαση να ερωτηθεί η ExxonMobil πώ θέλει να τηρήσει τη Σύμφωνα του ε, και να εξηγήσει ε, τις ε, τον αντίκτυπο που προκαλούν οι δράσεις της και πώς μπορεί αυτός να αντιμετωπιστεί. Επίσης, καλό θα ήταν και οι αρμόδιες επιτροπές να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Επομένως, θα ήθελα να διαβιβαστεί αναφορά στις επιτροπές ΕΝΒΙ και ΙΤΡΕ, δηλαδή Επιτροπή Ριβάλλους και Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η Επιτροπή παρακαλώ, κύριο Σούστερ. Σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τη δυνατότητα να αναφερθεί στο σημαντικό αυτό θέμα και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Κίνιγκερ για την εισαγωγική της παρέμβαση. Σίγουρα ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα παραπληροφόρηση ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και αυτό είναι όλο και πιο λυπηρό όταν ε, έχουμε πολύ αρνητικέ δράσεις για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί σίγουρα να αντιμετωπίσει τη τις αιτίες ε, της κλιματικής αλλαγής για να μετριάσει τις επιπτώσεις της. Ε, η παραπληροφόρηση υπάρχει και νομίζω ότι είναι δεδομένο ε, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στην Σύνθηκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης για όλους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, την μείωση, τον περιορισμό των θερμοκηπιακών αερίων, έχουμε ε, ευθύνη εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο καθένα βέβαια μπορεί να εκφράσει τι απόψει ε, του. Έχουμε επίση τα συμβαλόμενα μέρη που υπέγραψαν τη Συμφωνία των Παρισίων και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντες, επενδύτες, επιχειρήσεις, ε, αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις πολιτικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το πλανήτη μας, ότι χρειάζεται μια βιώσιμη διαχείριση ε, των πηγών ενέργειας ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνές επίπεδο και σε διάφορους φορείς και στο πλαίσιο των Εθνών αλλά και σε άλλους διεθνείς φορείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για το μετριασμό ε, των επιπτώσεων ε, της αλλαγής ε, του κλίματος. Η κυρία Κίνιγκερ, αναφέρουσα, μίλησε για τις έρευνες που ξεκίνησαν και διακόπησαν στις ίπα Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε γνώση και παρακολουθεί, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση, αλλά δεν υπάρχει αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, την δυνατότητα οποιοδήποτε να εκφράσει τις απόψεις του, ε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και της εν λόγω επιχείρησης. Και δεν μπορούμε επομένω ε, να προχωρήσουμε σε σχέση με το αίτημα της αναφέρουσας. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ, Μάντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που θίγεται το σημαντικότατο αυτό ζήτημα. Συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν απαγορεύεται από καμία νομοθεσία να αρνείται κανείς το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Σαφώς είναι λάθος, σαφώς αυτό είναι γελίο και σαφώς είναι και τραγικό να αρνείται κανείς την κλιματική αλλαγή, ιδίως αν αυτό συμβαίνει από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εφόσον όμως όλοι μας καλούμεθα να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση στα πλαίσια συζητήσεων, ε, στα πλαίσια χάραξης πολιτικής, ε, είτε στα πλαίσια των επιχειρήσεων, είτε στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. Ε, μπορούμε αυτό να το κάνουμε και κατά της άρνησης της κλιματικής αλλαγής, ενημερώνοντας σωστά τους πολίτες. Πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να επιλήφθει του ζητήματος Επιτροπή Αναφορών, διότι δεν παραβιάζεται κάποια νομοθεσία από το όλο ζήτημα. Επομένως, η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η δική μου προσωπική θέση είναι να κλείσουμε αυτή την αναφορά, λέγοντας πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε ορθά τους πολίτες για την κλιματική αλλαγή και κυρίως να λαμβάνουμε δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστούμε. κυρία Σκοτ, Σκάτο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω τα όσα μας είπε η κυρία Κένιγκερ και η συναδελφή της. Ε, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρουμε ότι ασκείται συστηματικό λόμπινγκ κατά της δράσης ε, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε ότι γίνονται εδώ πέρα προσπάθειες παρεμποδισμού της δράσης αυτής για την κλιματική αλλαγή. Τα ζητήματα αυτά αφορούν όλο τον πλανήτη, όλους τους πολίτες το γεγονό ότι υπάρχουν εταιρείε οι οποίε ασκούν λόμπινγκ, αρνούμενες τελικά φαινόμενα όπω κλιματική αλλαγή μόνο και μόνο για να κερδοφορήσουν περισσότερο, αυτό είναι απαράδεκτο. Εταιρείε σαν την ExxonMobil θα πρέπει να αποτελέσουν μέρο τη λύση και όχι του προβλήματο. Εταιρείε σαν και την ExxonMobil, οι οποίε ειδικεύονται στα ρηπτά καύσιμα, δεν έχουν άλλωστε κάποιο μέλλον πλέον. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουν και αυτέ να συνεργαστούν για έναν μετασχηματισμό όσον αφορά τις ε, πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των χρημάτων για να κινήσουμε την οικονομία προς ε, μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρακα και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει πλέον να εγκαταλειφθούν και να κινηθούμε προς άλλες πηγές ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι οι εταιρείε την ExxonMobil προασπίζονται τα κέρδη του και τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά από την άλλη υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Αυτήν πρέπει να προασπιστούμε και εμεί ω πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουμε να τηρήσουμε τι δεσμεύσει μα στα πλαίσια τη συμφωνία των Παρισίων. Η Συμφωνία πλέον αυτή θέτει συγκεκριμένε δεσμεύσει τι οποίε θα πρέπει να τηρήσουμε. Ξέρετε ότι ω ομάδα των Πρασίνων αναφερθήκαμε αυτή την εβδομάδα σε μια έκθεση που έχουμε συντάξει όσον αφορά το φαινόμενο των revolving doors, τη μεταπίδηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ ε, ιδιωτικέ εταιρείε. και αναφερθήκαμε επίση σε όλα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που προκύπτουν από τι καταστάσει αυτέ. Ε, επίση, θα ήθελα να αναφερθώ στο Ίδρυμα εκείνο, επικεφαλής του οποίου είναι ο κύριο Νάιτζελ Λόσον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίο ε, προασπίζεται βέβαια το Brexit και δεν δεσμεύεται τόσο πολύ για την ε, κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό να μπορούμε να εκφραζόμαστε όλοι ελεύθερα. Αυτό δεν το θέτουμε να αμφιβόλω. Θα πρέπει αυτό όμως να γίνεται με τρόπο διαφανή. Να μην έχουμε δηλαδή μυστικές διαπραγματεύσεις, να μην έχουμε εκστρατείες παραπληροφόρησης και να υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτά τα οποία κάνουν εταιρείε σαν την ExxonMobil. Υποστηρίζω λοιπόν ε, την ε, αναφέρουσα και θεωρώ ότι θα πρέπει, όπως είπε, να έχουμε μια δημόσια ακρόαση προκειμένου να δούμε τι δράση θα μπορούσε να ληφθεί κατά, να ληφθεί κατά αυτής της παραπληροφόρησης. Ευχαριστούμε, κυρία Εύη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω και εγώ το λόγο για να πω ότι υποστηρίζω αυτή την αναφορά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μία μέρα σαν τη σημερινή που για πρώτη φορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αναφερθήκαμε στη νέα οδηγία για την προώθηση των καθαρών αυτοκινήτων και για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ευτυχή αυτή η συγκυρία να μπορούμε τώρα και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών να συζητούμε σήμερα αυτή την αναφορά. Δεν θα πρέπει με τίποτα να μειώνουμε την επαγρύπνησή μα για το ζήτημα αυτό. Το αντίθετο μάλιστα θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά πω κάποιε ιδιωτικέ εταιρείε προσπαθούν να παρεμποδίσουν την όλη εργασία που γίνεται κατά των ορεικτών καυσίμων. Νομίζω ότι η στάση τους είναι εντελώ παροχημένη και αναχρονιστική. Δεν ε, μπορούμε πλέον να θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές που βασίζονται στα ορεικτά καύσιμα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο από 39 έως 200 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται ως ε, υποστήριξη σε επιχειρήσεις οι οποίες μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται και στον τομέα των ορεικτών καυσίμων. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια χρηματοδότηση, μια τέτοια χρηματοοικονομική υποστήριξη θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι προκειμένου να προωθήσουν άλλες πολιτικές. Θεωρώ ότι χάνουμε αυτή τη στιγμή σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Δείτε τι κάνει η Κίνα η οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ στην ηλεκτρική ενέργεια και πολύ σύντομα θα δούμε τα δικά τους ηλεκτρικά προϊόντα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι η αναφορά αυτή είναι πολύ σημαντική, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και προσβλέπω και εγώ στη διοργάνωση μιας δημόσιας ακρόασης, προκειμένου πραγματικά να δούμε ποια ήταν ε, η στάση τη εταιρεία αυτή και άλλων ε, παρόμοιων εταιρεών, οι οποίε προωθούν καμπάνιες παραπληροφόρηση ε, για την κλιματική αλλαγή και νομίζω ότι θα πρέπει η αναφορά αυτή να αποσταλεί προς ενημέρωση και στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βάιτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά μια επιχείρηση που κερδίζει με ε, τα ορυκτά καύσιμα ε, προσπαθεί τα αρνητικά στοιχεία ε, να τα κρύψει, αλλά το θέμα είναι ότι το 95% της επιστήμης, ε, των επιστημόνων μάλλον, ε, λέει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και υπάρχει ένα 5% που δεν το κάνει και αυτοί ανήκουν σε αυτούς που χρηματοδοτεί η ExxonMobil και άλλες τέτοιες εταιρείες. Θα ήθελα επίσης πολύ ξεκάθαρα τους συναδέλφους και κυρίως τον κύριο Μάντιλ που εκπροσώπησε την ε, ε, άποψη ε, της Αυστρίας και ιδίως και την αυστριακή κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε βέβαια σίγουρα και να τιμωρήσουμε την ε, ελευθερία έκφρασης, το λέω και για την Κομισιόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως ε, είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εκεί να στρίψουμε την προσοχή μας, ε, γιατί πρέπει να τους δείξουμε ότι η Mobil ενεργεί σε βάρος της υγεία τους για το συμφερόντων τους όταν αμφισβητεί την αλλαγή του κλίματος και αν δούμε και πώς προχωρούν τα λαϊκιστικά κόμματα στην Ευρώπη, ακριβώς αυτό κάνουν ε, βασίζονται στους 2, 3, 5 επιστήμονες στους οποίους επικαλούνται που μιλάνε ε, για ε, το κλίμα έχοντας χρηματοδοτηθεί από αυτές τις εταιρείες για, και μιλάνε για το ρηκτά τα κτλ. Δεν υπάρχουν όμως αμφιβολίες ότι αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να βοηθούν τη βιομηχανία και να δυσκολεύουν εμάς και την πολύ μεγάλη πλειονότητα στις χώρες μας που θέλουμε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Θέλω λοιπόν ξεκάθαρα να υποστηρίξω την πρόταση οργάνωσης μιας ακρόασης, να προσκληθεί και η ExxonMobil και δημοσία μπροστά ε, στους Ευρωπαίους ε, να μας πούν κατά πόσον έμαθαν το μάθημά τους, αν έχουν δεχτεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να μας πούν αν είναι διατεθειμένα να συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος ή θα διαψεύουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή ε, και επομένως να μας ξεκαθαρίσουν τι παιχνίδι παίζουν και αυτές τις επιχειρήσεις όπως η Nexon Mobile πλέον, αν έτσι κάνουν, πρέπει να τις τιμωρούμε και να μην τις αφήνουμε αλεξέλιτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις σας, ε, όλους σας. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα αυτό. Όλοι αισθάνονται ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. αλλά για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε άλλο σε αυτό το θέμα επίσημα, διότι είναι θέμα κρατών μελών, έχουμε την ελευθερία έκφρασης, αλλά οι διάφορε ομάδε μπορούν να λάβουν διάφορες δράσεις για να προχωρήσουμε. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να κάνω τίποτα παρά να σας προτείνω να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Εσείς θα πρέπει να με καθοδηγήσετε. Δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε οδός. Πιστεύω ότι αν κλείσουμε αυτή τη στιγμή την αναφορά κανείς δεν θα το ειστηρίξει. Το να οργανωθούν κάποια πράγματα δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτή εδώ η Επιτροπή. Πρέπει να το λάβει ως απόφαση να το λάβουν οι συντονιστές. Τι μπορώ να κάνω εγώ, θα το συμπεριλάβω στην ημερησία των συντονιστών, να δούμε αν θέλουν να το επιδιώξουν, τι να γίνει στο μέλλον. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να προτείνουμε η Επιτροπή σας να υποστηρίξει την ιδέα μιας ακρόασης παρότι δεν μπορεί να λάβει την απόφαση. Να το δώσετε, πείτε αυτό στους συντονιστές. Όχι, αλλά μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην ατζέντα των συντονιστών και ευχαρίστω εγώ να το πράξω αφού έχουν έτσι τα πράγματα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σας προσφέρω. Ωραία, ούτως και θα πράξουμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ. Καλή επιστροφή. Και τώρα ας κάνουμε μισό λεπτό διάλειμμα πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα. Ξανά καλησπέρα σας και ζητώ συγγνώμη για το διαλυματάκι αυτό. Χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να προετοιμάσουμε κάποια σημεία για την υπόλοιπη συνεδρίαση. Όλοι πιστεύω εδώ που βρίσκονται στην αίθουσα θα πρέπει είτε να καθίσουν κάτω είτε να αποχωρήσουν. People are leaving the room, which... Βλέπω κόσμο να φεύγει. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έξοχα. Πάμε στο σημείο 19, αναφορά 1024, σχετικά με την έλλειψη αντικειμενικότητας της ισπανικής τηλεόρασης. Έχουμε τους αναφέροντες μαζί μας. Σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτρόπη Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και ξεκινάμε δίνοντάς σας το λόγο. Νομίζω ότι η κυρία Μαρία Γκόμες Μπένιο θα είναι η πρώτη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που αφιερώνετε χρόνο για να μας ακούσετε. Λέγομαι Αθούν Γκόμες Μπένιο και είμαι εδώ ε, εκ μέρους του Συμβουλίου ε, Ειδήσεων TV που δημιουργήθηκε δυνάμει του νόμου 17-2006 της RTV. Τα 13 μέλη του ε, εκλέγονται από επαγγελματίες ε, της ενημέρωσης κάθε δύο χρόνια με καθήκον να διασφαλίζουν την εκδοτική ε, ανεξαρτησία του ομίλου. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ βλέπετε τι εξέπεμπαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ισπανία το πρωί της 26 Ιουλίου του 2017. Όπως βλέπετε όλα τα κανάλια πλην του TVE1 είχαν τον Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχώη, ως μάρτυρα σε δίκη για την κατηγορία ε, διαφθοράς του κόμματός του, του Λαϊκού Κόμματος. Ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ισπανικής που, ε, κυβέρνησης ε, εν ενεργεία εκλήθη ως μάρτυρας. Πιστεύουμε ότι αυτό δείχνει σαφώς τι συμβαίνει στην TV. Αυτό που βλέπετε συνέβη το πρωί. Την ίδια μέρα η εσωτερική προπαγάνδα που είχε αναπτύξει το κυβερνόν κόμμα για να καθαρίσει την δημοσία εικόνα του Πρωθυπουργού μεταδόθηκε σε ξεχωριστή είδηση στο δελτίο. Επρόκειτο για ένα εσωτερικό έγγραφο του κόμματο και στα δεξιά βλέπετε το έγγραφο της ανώτατη διοίκησης του TV, όπω ε, όπως το έδωσαν στου δημοσιογράφου για να γράψουν το είδηση. Είναι ακριβώ το ίδιο, αλλά δεν το είπαν αυτό στου δημοσιογράφου. Το παράδειγμα που βλέπετε εδώ δείχνει ότι η ανώτατη διοίκηση ε, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες υπέρ της κυβέρνησης. Επιπλέον έχουν απομακρύνει έμπειρους επαγγελματίες και τους έχουν αντικαταστήσει σε θέσεις ευθύνη με υπάκους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν ε, πληρούν τα επαγγελματικά ανεξάρτητα κριτήρια, τα επαγγελματικά κριτήρια ανεξαρτησίας αυτών που έδιωξαν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου του 2016 14 ε, ήταν η ημερομηνία μιας ε, αποφασιστικής αντίστασης. Εκείνο το απόγευμα ε, συνεδρίασαν στα γραφεία της Ανώτατης Διοίκησης για να διαμαρτυρηθούν βαθιά και σιωπηλά. Αυτή ήταν η πρώτη από τις αξιοπρεπέστατες διαμαρτυρίες του προσωπικού της RTV. Για παράδειγμα, τέσσερις μέρες πριν από τις γενικές εκλογές του Ιουνίου του 2016, ένα βίντεο μέλους της κυβέρνησης κυκλοφόρησε και σε αυτά που σε αυτά τα βίντεο που τα έδειξαν όλα οι σταθμοί, τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδε, ο τότε Υπουργό Εσωτερικών Χόρχε Φερνάντε Δία μιλούσε με τον επικεφαλή του Γραφείου Καταπολέμηση τη Απάτη τη Καταλωνία, ε, επιδόκοντα να βρει έναν τρόπο να ε, κατηγορήσει αυτονομιστές ηγέτες. Ε, αναφέρθηκε μεν η συνεδρίαση, αλλά λογοκρίθηκαν από όλη την RTV. Ή μάλλον να σας πω την αλήθεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο χρόνος ε, μετάδοσης μετατέθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Εδώ βλέπετε εικόνες των, ε, της διαμαρτυρίας εκείνης της ημέρας και άλλο ένα παράδειγμα πριν τελειώσω τα talk show της εβδομάδας πριν από την 1η Οκτωβρίου την ημερομηνία του δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας της Καταλωνίας αυτονομιστές ομιλητές ε, σπάνια καλούνταν να συμμετέχουν στα προγράμματα της RTV αληθεύει ότι το δημοψήφισμα δεν ήταν νόμιμο, ότι εμείς ως δημόσια τηλεόραση έχουμε την υποχρέωση να δείχνουμε τον πλουραλισμό της κοινωνίας μας, τα επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά του δημοψηφίσματος. Αυτός ο πλουραλισμός δεν φάνηκε, ήταν κρυφός. Απαγορεύτηκε την ημέρα του δημοψηφίσματος, δεν επιτράπηκε να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα στην TV1. Ήδη τα περισσότερα chat shows στην έδειχναν μια θέση της κυβέρνησης ε, έδειχναν τη θέση της κυβέρνησης και όχι τη θέση των ε, κόμματων της αντιπολίτευσης. Εδώ βλέπετε την παρουσία των πολιτικών κομμάτων στην ΤΒΕΝ στο κύριο δεσογραφικό δελτίο στις 8 Μαρτίου που ήταν μια σημαντική ημέρα. Η πρώτη φεμινιστική απεργία στην ιστορία της Ισπανίας με τεράστια προσέλευση. Γι' αυτό το λόγο καταγγέλουμε την ανώτατη διοίκηση τη ΑΡΤΕΒΕ, επειδή δεν συμμορφώνεται με την Ισπανική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων θεσπίζει ότι τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρούν τι αρχέ αντικειμενικότητα, πλουραλισμού και αμεροληψία. Το ίδιο προβλέπει και η Ισπανική νομοθεσία. Το RTV παραβιάζει μία από τις ε, θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών τη και την ελευθερία τύπου θεμελιώδεις αρχές για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Χωρίς την ελεύθερη δημοσιογραφία δεν υπάρχει δημοκρατία. Όλοι το γνωρίζουμε. Γιατί όμως πρέπει να ερχόμαστε εδώ και να το επαναλαμβάνουμε. Είναι θλιβερό. Όπως βλέπετε έχω ντυθεί στα μαύρα. Το ίδιο και οι συνάδελφοί μου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και πάλι να διαμαρτυρηθούμε για την RTV. Το κάνουμε κάθε Παρασκευή. Όχι όλοι, οι περισσότεροι από εμάς όσοι βρισκόμαστε πίσω από τις κάμερες σε κλειστές πόρτες. Τέλος, τι σας ζητάμε να κάνουμε. Παρακαλώ, ενώστε τις δυνάμεις σας, κυρίες και κύριοι, με τις δικές μας, στην καθημερινή μας μάχη. Ζητήστε την Ισπανική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όσοι είναι αρμόδιοι για την RTV να συμμορφωθούν με την Ισπανική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Α δώσουμε την RTV πίσω στους πολίτες, στους πραγματικούς ιδιοκτήτες της Ισπανική Δημόσια Τηλεόραση για τους οποίους πρέπει και θέλουμε να δουλεύουμε. Να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω με αυτή την ιδέα η οποία εκφράζεται σε αυτό το φίλμα. Before I finish, Πριν τελειώσω θα ήθελα να ευχαριστήσω τα θεσμικά όργανα και τις ομάδες που υποστήριξαν το αίτημα του Ιδιοσιογραφικού Συμβουλίου, την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογραφών, Δημοσιογράφων, τους Reporters Without Borders, διάφορες ενώσει δημοσιογράφων και το κίνημα γυναικών της RTV. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεπεράστε λίγο τον χρόνο που προβλεπόταν. Πέντε λεπτά σας είχα δώσει και μιλήσατε για επτά λεπτά. Αυτό όμω δεν σημαίνει, και το ξεκαθαρίζω, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δικαιούστε να περάσετε το χρόνο αγόρευση. Έδωσα λίγο περισσότερο λόγο στην αναφέρουσα, ήμουν λίγο πιο επίκη μαζί τη. Η επίκη αυτή όμω δεν ισχύει για όλου του υπόλοιπου. εντάξει. Τίθεται ότι θα είχαμε και τον εκπρόσωπο της RTV σήμερα μαζί μας, αλλά αποφάσισε τελικά να μην έρθουν. Μας στείλανε ένα πολύ εκτενές έγγραφο ηλεκτρονικά. Στη γραμματεία έφτασε το έγγραφο αυτό. Είναι πολυσέλιδο πραγματικά και νομίζω θα ήταν ε, δύσκολο τώρα να σας το δώσουμε, το διανύμουμε σε όλους. Πάντως στην ηλεκτρονική σελίδα μας ή πέτη μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο αυτό. Μπορείτε να το ανοίξετε με τον υπολογιστή σας και μπορεί να σας βοηθήσει και η γραμματεία αν χρειάζεστε βοήθεια. Απουσία πάντως ε, των εκπροσώπων του RTVE δίνω το λόγο στον κύριο Φίλιμπεκ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσουμε αυτή την αναφορά. Σας έχουμε δώσει, θεωρώ, και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη. Θα ήθελα να θίξω λίγο το νομικό πλαίσιο για την αφορά αυτή. Τα βασικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ότι προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια δημοκρατική κοινωνία να υπάρχει ένας αμερόληπτος φορέας ραδιοτηλεόρασης που να λειτουργεί ανεξάρτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να πω ότι οι αρμοδιότητες ανάληψης δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό είναι πολύ περιορισμένες. Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη αναφορά, το πρωτόκολλο για τις βασικές συνθήκες, το πρωτόκολλο υπαριθμών 29, αναγνωρίζει τη σημασία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά αναθέτει αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη προκειμένου να αποφασίσουν την εντολή χρηματοδότηση και τις περαιτέρω αρμοδιότητες Τη δημόσια ραδιοτηλεόρηση. Ο Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στο άρθρο 11 αναφέρεται στον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως βασική θεμελιώδη ελευθερία μαζί με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Επίσης, ο χάρτης ισχύει για τα κράτη-μέλη που εφαρμόσουν το νοσιακό δίκαιο. Αυτό πολύ κρίσιμη σημασία. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επέμβει στα πλαίσια μια διαδικασία σε παραβάση όταν παραβιάζεται κοινοτική νομοθεσία. Εμεί μπορούμε να λάβουμε δράση μόνο στα πλαίσια του χάρτη όταν υπάρχει διασύνδεση και μόνο τότε με την κοινοτική νομοθεσία. Όσον αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη αναφορά, δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική νομική βάση προκειμένου να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ το λέω αυτό. Μολονότι μα μίλησε πολύ συναισθηματικά φορτισμένη σήμερα η αναφέρουσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει δράση. Για να κλείσω όμω και την παρέμβαση μου αυτή με μια πιο αισιόδοξη ξέρετε ότι ε, αυτή τη στιγμή η οδηγία όσον αφορά την δημόσια ραδιοτηλεόραση βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης. Έχουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από το Μάιο του 2016 και προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την ε, ραδιοτηλεόραση και άλλους κρίσιμους δημόσιους φορείς. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και χέγγια ανεξαρτησία τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Τι τελευταίε εβδομάδε, πολύ πρόσφατα μάλιστα, τα θεσμικά όργανα κατέληξαν σε μια ευρεία συμφωνία όσον αφορά τα περισσότερα στοιχεία αυτή τη αναθεωρημένη οδηγία συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων εκείνων που έχουν να κάνουν με την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση. Η αναθεωρημένη λοιπόν αυτή οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα θα προωθήσει περισσότερο, θεωρούμε, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση και αυτή τη στιγμή εγκριθεί και τεθεί σε ισχύ από τα κράτη-μέλη. Οι διατάξει αυτέ πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικέ επιπτώσει για, τις, ε, για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση και ειδικότερα για τι υπηρεσίε ραδιοτηλεόραση. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει επίσημη δράση, δεν μπορούμε εμείς να ασκήσουμε πίεση αυτή τη στιγμή στην Ισπανική κυβέρνηση. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ρεοτηλεόραση να ακολουθεί τις βασικές αρχές της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι ευρωβουλευτές τώρα έχουν το λόγο και ως εκθαύματος βλέπουμε εδώ πέρα την ισπανική κυρίως αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Όλος τυχαίως, όλος τυχαίως με μία-δύο εξαιρέσεις βλέπουμε σχεδόν όλους τους Ισπανούς ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή με το χρόνο όμως. Δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ Σίλια. Νομίζω ότι τελευταία είχα στήσει το λόγο, αλλά τέλος πάντων. Ε, σε ευχαριστώ. Ε, θέλω να πω ότι... Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τους προσώπους ε, της ε, Ισπανικής Ραδιοτηλεόρασης. Ε, πολύ γενναία στάση τους και δύσκολη μετά από τόσα χρόνια. Είναι κάτι που δεν έχει ξεκινήσει, αλλά ξεκίνησε με ένα από τους σημαντικότερους νόμους. Είχαμε πρόοδο για τη δημοσιογραφία και γενικά την ελευθερία Είχαμε την προλαριστική τηλεόραση με την ομοθεσία Θαπατέρο. Ε, και σήμερα ουσιαστικά αυτό ζητούν ε, οι δημοσιογράφοι σίγουρα ε, με την αντιπολίτευση από το Λαϊκό Κόμμα. Η Ισπανία είναι αυτή που θέλει τώρα το Λαϊκό Κόμμα. Εμείς όμως έχουμε σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι η Ισπανία τη δημοκρατική. Κάποια δημοκρατικά στοιχεία ναι υπάρχουν και έχουμε και τον νόμο που φημώνει την ελευθεροτυπία ή έχουμε την ε, ποσοστώσει στη δικαιοσύνη που δυσκόλευαν την πρόσβαση. Είχαμε μείωση επίσης ε, των ε, πολιτικών ελευθεριών. Όλα αυτά μέσω του Λαϊκού Κόμματος. Υπάρχει μια υποχώρηση και υπαναχώρηση Ίσως ο στόχος είναι η επιθυμία ελέγχου των μέσων ενημέρωσης ανώπιση των προσεχών γενικών εκλογών. Αυτό που θέλω να στήσω εγώ είναι να προασπιστεί η ελευθεροτυπία. Η δημοκρατία βασίζεται μεταξύ άλλων στην ελευθεροτυπία. Ε, και είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά και θα πρέπει εμείς να στείλουμε ως Επιτροπή Αναφορών ε, στο Κοινοβούλιο και στη Γερουσία και στην Ισπανική Κυβέρνηση για να ε, ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Μία επιστολή λοιπόν την οποία θα υπογράφουν όλοι οι Ευρωβουλευτές. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς ε, θα μπορούσε να αιτιολογήσει τον έλεγχο της δημόσιας τηλεόρασης και την κατάργηση ουσιαστικά της ελευθεροτυπίας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Άγγελα Βαλίνα. Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέρους καταρχάς για το στένος τους, για την ε, γενναιότητα το θάρρος να φτάσουν εδώ και να καταγγείλουν ε, την χειραγώγηση και τη φήμωση ε, του τύπου, αλλά και γιατί προασπίζονται ένα δημόσιο μοντέλο για την Ισπανική ραδιοτηλεόραση που θα γιάται σε όλους τους Ισπανούς και τις Ισπανίδες που το πληρώνουμε το δικαίωμα στην πραγματική πληροφόρηση, στην αντικειμενική και πλουραλιστική πληροφόρηση, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε ούτε κατά διάνοια. Νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ ξεκάθαρες οι καταγγελίες, ε, είδαμε ε, κάποιες και μεταφέρουν αυτή την κατάσταση καταχρήσεων και μη επαρκούς πράσπισης των εργαζομένων. Πρόκειται για μια κατάσταση που φαίνεται ότι προέκυψε όταν έφτασε στην εξουσία το Λαϊκό Κόμμα το 2011 και επιδεινώθηκε σίγουρα Κάποια χειραγώγηση στην πληροφόρηση πάντα υπήρχε. Και οι ειδήσει ε, μας δείχνουν ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση μετά το 2011 σε βαθμό που σήμερα είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητούμε το θέμα αυτό, να, που συζητούμε αν η Ισπανία εφαρμόζει σωστά το χάρτη θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων και το δίκαιο της Ένωσης. Ε, νομίζω ότι η δομή ε, της Διεύθυνσης των Ενημερωτικών Δισογραφικών ε, ε, Υπηρεσιών δεν σέβεται τον νόμο του 2006 για την ραδιοτηλεόραση. Δεν τηρεί τις αρχές αντικειμενικής πληροφόρησης, της αληθούς και πλουραλιστικής πληροφόρησης, ούτε την ελευθερία έκφρασης, ούτε προωθεί την εδαφική συλλογή και την, το πλουραλισμό. Είμαστε σε ένα σενάριο σίγουρα παραπληροφόρησης ή μερικής πληροφόρησης. Ε, δεν υπάρχει δημοσιογραφική ε, ακρίβεια. Και γι' αυτό ζητώ να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, να ζητηθούν περισσότερε πληροφορίε από την Κομισιόν για να δούμε κατά πόσο παραβιάζεται ο χάρτη των μελετών δικαιωμάτων και να ζητήσουμε και από τι Ισπανικέ αρχέ πληροφορίες. Και εγώ συμφωνώ με την αποστολή αυτή τη επιστολή, αλλά θα πήγαινα και πιο μακριά. Θα έλεγα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ουσιαστικά είναι το σύμπτωμα του προβλήματο. το πρόβλημα είναι το μοντέλο το ίδιο, το μοντέλο τηλεόραση που έχουμε είναι μια δημόσια τηλεόραση, αλλά κατά την άποψή μου είναι κρατική. Αλλά όχι με την έννοια του κρατικού εθνικού, αλλά την έννοια του κρατικού κυβερνητικού. Είναι κυβερνητική η τηλεόραση. Εμείς θα θέλαμε να είναι αντίστοιχο, αντίστοιχη η ισπανική ραδιοτηλεόραση με το BBC, με το γερμανικό μοντέλο. Έτσι θα ήταν εγκυμένα όλα τα δικαιώματα των Ισπανών, που πληρώνουμε για να έχουμε πληροφόρηση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιράντα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Λαϊκό Κόμμα που είναι στην κυβέρνηση σήμερα, όπως είπατε και εσείς, ε, ε, χειραγωγεί, φημώνει, λογοκρίνει, χωρίς να ερυθριά. Ε, και βλέπουμε τι κάνουν ε, και οι δημοσιογράφοι. Ντύνονται στα μαύρα και διαδηλώνουν κάθε Παρασκευή. Το μαύρο είναι το χρώμα του πένθους, το χρώμα της θλίψης αλλά και της χειραγώγησης, ε, της αδιαφάνειας των ζωφερών καιρών της λογοκρισίας του τύπου. Η ελευθεροτυπία είναι το κεντρικό στοιχείο της δημοκρατίας, το κεντρικό στοιχείο της ελευθερίας έκφρασης. Το Ισπανικό κράτος αυτή τη στιγμή απειλεί με την έλλειψη ελευθερίας έκφρασης, με καταστολή και των μέσων ενημέρωσης, όπως το είδαμε και στις εικόνες, που είναι λίγες, υπάρχουν πολύ περισσότερες. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για το θάρρος ε, τους αναφέροντες, ε, για το κουράγιο που έδειξαν, για τη γενναιότητα που σίγουρα συνεπάγεται αντίπεινα, μετατάξεις, αλλαγή πόστου κτλ. Ακόμα και σε δαφικές αντιπροσωπείε στη Γαλλική, στη Μαδρίτη. Τα ελεύθερα πλωραλιστικά μέσα ενημέρωση όμω είναι σπονδυλική στήλη τη Δημοκρατία. Πώ μπορεί να λέει η Κομισιόν, όπω μα είπε πριν, ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει, ε, ότι θα εγγυάται η τηλεόραση σέβεται την πολυμορφία όταν εγκρίναμε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πλουραλισμό και μέσα επικοινωνίας που ζητά ακριβώς ε, να είναι δημόσια αυτά τα μέσα σε ό,τι αφορά την ισπανική τηλεόραση μιλάμε για χειραγώγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και θα πρέπει να εμπλακεί, θα πρέπει να δώσει την άποψή της, μα γι' αυτό είμαστε εδώ, αλλιώς τι κάνουμε εδώ αν δεν εγγυόμεθα δικαιώματα και ελευθερίες. Η έλλειψη αυτή ανεξαρτησίας είναι δημόσια υπηρεσία, από την πληρώνουμε με φόρους, με τέλη που σίγουρα περικόπτουν, ε, ε, ε, έχουν περικόψει και τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορεί αυτή η δημόσια υπηρεσία να φημώνεται, να λογοκρίνεται. Και η πράσινη και η άλλη ζητεί να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να πάμε και πιο μακριά. Να στείλουμε μια τχόκα αντιπροσωπεία πριν το τέλος της θητείας. Να πάμε να δούμε το ΔΣ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τι κρίμα που είναι ε, στην υπηρεσία ε, του κοινού ε, που χρησιμοποιούμε την Επιτροπή με αναφορών για την προεκλογική εκστρατεία στην Ισπανία. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Ακούστε. Και το λέω στην κυρία ε, ότι είχαν οκτώ λεπτά οι αναφέροντες και δύο λεπτά έχουμε εμείς οι βουλευτές, ε, κυρία Μιράντα. Ε, εσείς μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αυτά που λέτε Καλό είναι πάντως να ακούμε και τις δύο πλευρές. Έχω άκουσα και τις δύο πλευρές και τους αναφέροντες, έχω συναντήσει, τους καλωσορίζω και την Κάρμεν Σάστρε όμως είδα και τη διεύθυνση ε, της ε, ραδιοτηλεόρασης. Η Κάρμεν Σάστρε 40 χρόνια είναι στο τιμόνι ε, της ε, αρχισυνταξίας από σοσιαλιστική ομάδα. Ήταν ε, και συνήγορος για πολλά χρόνια. Η η Ισπανική τηλεόραση έχει του περισσότερου ελέγχου από την Ισπανία. Υπάρχει επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου και τη ε, Γερουσία ε, που ελέγχει και μηνιαίως ο πρόεδρος της εταιρείας Ισπανική Ραδιοτηλεόραση παρέσταται στην Επιτροπή, λογοδοτεί στην εκτελεστική εξουσία και στον έλεγχο ε, της ε, Εθνικής Επιτροπής που ελέγχει ε, τις αγορές είναι υπόλογη η Ισπανική Ραδιοτηλεόραση. τα δελτία ειδήσεων σέβονται τον πλουραλισμό στην Ισπανία και μάλιστα πάρα πολύ Το λένε σε εκθέσεις του 2015 και 2016 οι ρυθμιστικές αρχές, η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού και αγορών και τα δελτία τα βλέπουν οι περισσότεροι πολίτες τους τελευταίους 18 μήνες. 16% είναι το ποσοστό τηλεθέασης και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα δελτία ειδήσεων πήραν και βραβείο ούτε λίγο ούτε πολύ από την Ακαδημία της Ισπανικής Τηλεόρασης που περιλαμβάνει πάνω από χίλιους επαγγελματίες. Το 2017 το δελτίο ειδήσεων πήρε αυτό το βραβείο για το καλύτερο δελτίο ειδήσεων. Πήρε το βραβείο από την Ακαδημία και το έχει Ανκόν βραβείο. Δέσμευση για την ε, υπέρ της πολυμορφίας και του πλουραλισμού. Υπήρχαν 108 προσφυγές ε, οι 98 ε, δεν κρίθηκαν παραδεκτές, μόνο 10 κρίθηκαν παραδεκτές προσφυγές ε, και ε, όχι όλες για έλλειψη πλουραλισμού. Το RTVE έχει πολλούς αναλυτές, έχει πολλούς δημοσιογράφους από 40 μέσα έχετε όλα τα στοιχεία και από ό,τι ξέρω και τα λέει και η διεύθυνση είναι ότι ο Ραχόη πράγματι, να και ολοκληρώνω, όταν ε, ήταν μάρτυρας ε, στις 26 Ιουλίου και στο TV1 και στο TV2 ε, προβλήθηκε η, η ακρόαση που έδωσε. Και ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι και μια ξένη συμβουλευτική εταιρεία είπε ότι είναι πληρέστετα τα δελτία ειδήσεων. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που μας λέτε εδώ και γι' αυτό θα ζητήσω ότι δεν, δεν θα υποστηρίξω την επιστολή. Μακάρι να είχε κληθεί η Ισπανική κυβέρνηση, όπως προβλέπει το άρθρο 11 των κατευθυντηρίων γραμμών και μιλούν ταυτόχρονα ο πρόεδρος και η κυρία Εσταράς. Τουλάχιστον η δική μου φωνή προασπίζεται την Ισπανία και όλους τους Ισπανούς πολίτες. Εγώ έβγαλα τα ακουστικά μου, λέει ο πρόεδρος. Γιατί δεν μπορούσα ε, να κλείσω το μικρόφωνο όπως μπορούν να το κάνουν οι πρόεδρες στην Ολομέλεια. Θα το είχα κάνει, θα είχα κλείσει το μικρόφωνο εμένα μπορείτε να με επηρεάσετε όταν σας ακούω. Αν δεν σας ακούω δεν μπορείτε να με επηρεάσετε. Πήρατε το λόγο για πάνω από δύο λεπτά, δύο παραπάνω μάλιστα από αυτά που είχατε στη διάθεσή σας. Και αυτό δεν είναι ok σε καμία περίπτωση. Μπεατρίθ Μπεθέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προσπαθήσω να περιοριστώ ε, στους κανόνες μας. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους αναφέροντες και θα ήθελα εδώ να επενθυμίσω ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει δημόσια τηλεόραση που έχει ένα δημόσιο λειτουργήμα λάβει και όλες ε, οι ραδιοτηλεόρασει στην Ευρώπη το ίδιο, την ίδια πρόκληση αντιμετωπίζουν παρά τους εσωτερικούς κανονισμούς, τους κανόνες που ισχύουν ε, και στην οργάνωση και στη χρηματοδότηση. Ε, υπάρχουν διαφορέ στην Ισπανία σε σχέση με τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε για την τηλεόραση, αλλά η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμό είναι κλειδί για τη δημοκρατία σε κάθε χώρα, για του πολίτε και ιδίω για εμά του νομοθέτε. Είναι κάτι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία αυτή η έννοια, αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται και στα κανάλια των αυτόνομων περιφερειών που σε περισσότερες περιπτώσεις ε, μεταφέρουν ε, τα απόψει ε, των κυβερνήσεων των περιφερειακών. Ουσιαστικά βλέπουμε τις γενικές αρχές σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Το θέμα είναι να υπάρχει αντικειμενικότητα, αλήθεια, βασμό στην πολυμορφία αντικειμενικότητα. Δεν είναι σωστό να γίνεται κομματική προπαγάνδα το λιγότερο που μπορώ να πω, ε, διότι έτσι ο τύπος γίνεται ένα εργαλείο για την καταστροφή ε, της ε, συνταγματικότητας, όπως συμβαίνει με το TV3 στην Καταλωνία ή με τις καταγγελίες που ακούσαμε σήμερα από τους αναφέροντες. Πρέπει να προασπιστούμε την ελεύθερη και αντικειμενική ε, τηλεόραση. Δεν μπορούμε ε, να αποφύγουμε την προσπάθεια των κυβερνήσεων να έχουν την εξουσία, όμως ε, και οι δημοσιογράφοι ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία και πρέπει και αυτοί να μπορούν να μιλούν ελεύθερα. Η Κομισιόν μιλά για γρήγορες κινήσεις ό,τι αφορά την αναθέτηση οδηγίας. Ελπίζουμε να υπάρξουν νέε απαιτήσει για να επιτύχουμε την ανεξαρτησία. Γιατί πρέπει να το λέει αυτό το Ευρωπαϊκό και Το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο παγόμαστε θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Για να ζητηθεί ακριβώς η εφαρμογή τη οδηγία με αυτέ τι νέε απαιτήσει και από του νέου αυτού όρους. Thank Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί η στα Σταράση συντρόφισα τα έπε όλα, τα έδωσε όλα τα στοιχεία που ε, νομίζω ότι ξεκαθαρίζουν πολύ το θέμα. Ουσιαστικά είναι μια εκστρατεία δυσφήμισης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Εγώ νόμιζα ότι οι αναφέροντες μιλούσαν για το TV3 και την Καστίγια Λαμάντσα, ε, όπου εκεί είναι πράγματι υπάρχει πολιτικός έλεγχος και υπάρχει έλλειψη πλουραλισμού. Τέλος πάντων, εγώ σας παρακαλώ να διαβάσετε το έγγραφο το οποίο έστειλε η Ισπανική Ραδιοτηλεόραση, Τελευσιόν Εσπανιόλ. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε τέσσερις εικόνες εκτός ε, context. Μπορεί να μην είναι ακριβώς να στο ίδιο. Αυτό που είναι σημαντικό ε, γίνεται λόγος εδώ για έλλειψη πληροφόρηση, για χειραγώγηση. Για μένα έλλειψη πληροφόρηση πλουραλισμού είναι από την πλευρά της εκπροσώπου Σοσιαλιστικού Κόμματος που, έφερε τους αναφέροντες αλλά και τους αναφέροντες που πήρε μικρόφωνο στην ε, ε ραδιοτηλεφόρηση. Εγώ δεν είχα ποτέ μικρόφωνο της Ισπανικής τηλεόρασης ε, όσα χρόνια είμαι βουλευτής. Τώρα έχω βέβαια μικρόφωνο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην δοθεί η εντύπωση ότι η συζήτηση είναι καθαρά ισπανική, θα ήθελα να πω κι εγώ ότι ούτε η Σλοβενία αποτελεί υπόδεγμα δημοκρατικής συμπεριφοράς όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο έχουμε μια δημόσια τηλεόραση. Το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι είναι πολύ αυστηρή και επικριτική προς την κυβέρνηση ελέγχουν δηλαδή την, την κυβέρνηση. Αυτό κάνει η δημόσια τηλεόραση και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα παντού. Συγχαίρω τους αναφέροντες ε, που ήρθαν εδώ. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται λίγο ενθάρρυνση. Έχετε μεγάλο θάρρος που ήρθατε εδώ και ανοίξατε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο για τα ε, στάνταρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί βασικό λειτουργήμα, βασικό καθήκον όλων μας το να μεριμνούμε ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι ισορροπημένα, να είναι δίκαια και ανοιχτά. Με απεριόριστη πολυφωνία. Έχω την αίσθηση ότι η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας ε, έχει πρόβλημα. Από τα όσα ακούω βέβαια στη συζήτηση σήμερα αντιλαμβάνομαι το ταμπεραμέντο, έχω Ισπανούς συναδέλφους με τους οποίους ενίοτε διαφωνώ και εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι και έτσι θα παραμείνουν τα πράγματα. Είχαμε την υπόθεση των ειδήσεων για την Καταλωνία και για το σχετικό θέμα που αναφέρθηκε. Εγώ το παρακολουθώ στενά και περισσότεροι γνωρίζετε γιατί και πραγματικά σας μιλάω, η δημόσια τηλεόραση δεν μπορεί να μεταχειρίζεται έτσι ένα τόσο περίπλοκο ε, και δύσκολο ζήτημα. Δεν μπορεί δηλαδή να βάζει μια ετικέτα στη μία πλευρά και να λέει ότι είναι σχεδόν εγκληματική, ούτε να υποστηρίζει την καταστολή και τα μέτρα ξέρω, φυλάκισης ολόκληρης της ε, κυβέρνησης και του αιρετού εκπροσώπου στην Ισπανία. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ που φέρατε αυτό το πρόβλημα στην Επιτροπή μας. Πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Είναι τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, ε, τι μπορεί να κάνει η κοινή γνώμη σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα στην ίδια την Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχω ένα τεράστιο κατάλογο μιλητών. Θα δώσω το λόγο πρώτα στα μέλη της Επιτροπής και μετά σε όσους δεν είναι μέλη της Επιτροπής αλλά είναι ευρωβουλευτές. Θα πάρετε το λόγο όλοι, αλλά προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε σε κάποιο είδους... Θα πρέπει να ορίσουμε κάποια προτεραιότητα, οπότε τα μέλη θα λάβουν πρώτα το λόγο και μετά τα μη μέλη. Οπότε τώρα έχουμε την κυρία Τερικάβρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι καλό που η φίλη Ρώσα Εσταράσα με πολύ συμφιλιωτικό τόνο υπερασπίστε την Ισπανία. Τι κρίμα, αυτό είναι κρίμα. Και άλλοι εποφελούνται και μιλάνε για άλλους σταθμούς τηλεόρασης που δεν είναι το θέμα μας. Αυτό είναι κρίμα. Είπατε για, την, ε, για το τι διακυβεύεται εσείς από την Κομισιόνα. Όλα τα ακούσαμε. Τα γεγονότα είναι αυτά που είναι, τα είπαν οι εκπρόσωποι της επιχείρησης αυτής και είναι γεγονότα, διαφυσβήτητα. Τώρα το θέμα είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτήν θέλω να κριτικάρω. Πραγματικά λυπούμε και θλίβομαι που δεν προστατεύεται τους πολίτες και τους δημοσιογράφους. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε, τουλάχιστον εμείς στην Επιτροπή Αναφορών και να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι η τηλεόραση όλων και όχι της κυβέρνησης στην Ισπανία, σε όλη την Ισπανία. Η δημόσια τηλεόραση είναι ιδιωτική τηλεόραση τη κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση όπου και αν είναι αυτή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το θέμα λέγεται ισπανική τηλεόραση. Όμω ε, θα έπρεπε να λέμε είναι ε, το πρόβλημα της κάθε δημόσιας ε, τηλεόρασης στην Ισπανία. Εγώ καταλαβαίνω τη μεγάλη ευαισθησία κάποιων αυτονομιστών. Θα ήθελα να είναι το ίδιο ε, ευαίσθητο. Θα μιλήσουμε για, την, ε, για το σταθμό τ.ε. 3 είναι ο διευθυντή υπέρ τη απόσχεση και αυτό είναι το δικαίωμά του, αλλά πρέπει και αυτό να τηρεί τα περί πλουρανισμού κτλ. Υπάρχει αυτή η επαγγελματική δίκτυα, την οποία εγώ υποστηρίζω και γιατί οραματίζομαι διαφορετικά την ισπανική τηλεόραση, αλλά και γιατί είμαι δημοσιογράφος ε, εδώ και 40 χρόνια. Όμως αυτό που λέει ε, το ε, Συμβούλιο Σύνταξη είναι σωστό, αλλά ισχύει για όλε τι δημόσιε τηλεοράσει. Δεν είναι πρόβλημα ούτε του ΠΕΣΟΕ ούτε του Λαϊκού Κόμματο. Ε, αυτό ε, που ξεχνάμε εδώ είναι ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα, να υπάρχει πραγματική αληθινή δημόσια τηλεόραση. Η τηλεόραση όμω χρησιμοποιείται, χειραγωγείται για τα συμφέροντα των διαφόρων κυβερνήσεων. Το ίδιο συμβαίνει και με το TV και με το tv 3 Εγώ στηρίζω να ανοίξει ε, η αναφορά. Ε, η να παραμείνει ανοιχτή. Αλλά ελπίζω την ίδια ηθική να την εφαρμόσουν και για το τεράστιο σκάνδαλο του TV3, TV3. Ευχαριστώ, Μητροφάνος. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ μια, ένα κόμμα μηνωτικό τη και πρέπει να σας πω ότι ε, μας απασχολεί και μας η υπόθεση αυτή. Ξέρετε ότι εμείς ως μειονότητα δεν είχαμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στην επίσημη γλώσσα της χώρας μου, εκπροσωπώντας τη μειονότητα αυτή, δεν μας δόθηκε καμία διάβλος μέσω των μέσων ενημέρωσης. Επομένω θεωρώ ότι η αναφορά αυτή συνδέεται και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη δική μου τη χώρα, με την, δημοκρατι... κατάσταση δημοκρατίας στην χώρα μου. Προσπαθούμε εμεί τώρα να παρακάμψουμε την κατάσταση αυτή χρησιμοποιώντα το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Το πρόβλημα όμω τώρα, το οποίο βλέπουμε στην Ισπανία, ενδεχομένω να είναι πιο σοβαρό τελικά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινότητα η οποία δεν μπορεί να απευθυνθεί καν στους πολίτες, στους ψηφοφόρους. Τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και ενδεχομένως θα έπρεπε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εδώ στο Κοινοβούλιο να ζητήσουμε να κάνει μια ευρύτερη διερεύνηση της κατάστασης που ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δυνατότητα χρήσης της δημόσιας τηλεόρασης. Έχετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με τη συζήτηση στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Συζητούμε όμως συγκεκριμένη αναφορά, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν κάνουμε μια ευρεία συζήτηση ακρόαση για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Ας το έχετε αυτό κατά νου. Λόπες Έχω δύο λεπτά στη διάθεσή μου. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ελευθερία έκφραση. Και ο πληρολισμό τη δημοσιογραφία, ιδίω για τα δημόσια μέσα, φυσικά και είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα στην Ισπανία. Άρθρο 20. Και είναι πολύ σοβαρό εδώ να έχουμε σαφή επιχειρηματολογία και παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αυτή η παραβίαση του πλουραλισμού. Αλλά κυρίως ε, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη το άρθρο 7, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου. Έχουμε ασχοληθεί με τον δημοσιογραφικό ε, πλουραλισμό. Εγώ λοιπόν θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου ε, στο να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και θέλω να γίνει γνωστό το θέμα ε, και θα προβάλλω και τις απόψεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Οι εκπρόσωποι που έφεραν το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών δεν είναι μισθοφόροι, δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Είναι μέλη του Συμβουλίου ε, των ε, Συντακτών των Δελτίων Ειδήσεων είναι επαγγελματίε έξω και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επαγγελματίε που δεν ε, πρόσκειται σε κανένα κόμμα έρχονται εδώ και καταδεικνύουν ότι υπάρχει συνεχή χειραγώγηση των δικτύων ειδήσεων. Αυτό που θέλω να τονίσω όμω είναι ότι δεν είναι αλήθεια ότι είναι ένα ε, πρόβλημα που αφορά όλου του σταθμού και όλα τα κανάλια ε, στην Ισπανική τηλεόραση, σε όλε τι αυτόνομε περιφέρειε. Σίγουρα υπάρχουν βαθμοί, βαθμίδε ο πλουραλισμός ε, πολλές φορές ε, ε, ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε το 2006 τον νόμο που ακύρωσε όταν ήρθε το ΑΕΛΚ στην εξουσία αμέσω. Και αυτός ο νόμος το 2006 εγγύει άτο την πλουραλισμό. Και ήταν υποδειγματικό αυτό για την Ισπανία. Και τότε θέλαμε να πλησιάσουμε και πλησιάζαμε το BBC. Το πρόβλημα είναι τι κάνει τώρα το ΤΕΒΕ. Είναι πολύ θεμητή η καταγγελία και εμείς θα τη στηρίξουμε από την ομάδα μας. Κύριε Ραφ Γκαρθία, ευχαριστώ πολύ η ποιότητα και το μεγαλείο, αν θέλετε, του έργου ενός σταθμού, μιας τηλεόρασης στους επαγγελματίες. Ε, κυρία Καμπεθόν, έχει μπροστά της ένα μικρόφωνο. Δεν έπρεπε να το έχει και η κυρία Σταράς Είναι και οι δύο μέλη της Επιτροπής. Τι κάναν αυτοί οι επαγγελματίες εδώ, αρνήθηκαν να το κάνουν. Και αυτό είναι άδικο και δείχνει, δείχνει την ποιότητα αυτής της αναφοράς. Τι γίνεται εδώ ουσιαστικά. Είναι ότι βρισκόμαστε ε, απέναντι σε μια καμπάνια τη πολιτικές σκοπιμότητες ε, ε, σε ό,τι αφορά την αλλαγή και του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ε, το είπε και η κυρία Καμπεθόν ότι υπάρχουν κοντά εκλογέ. Είναι τελείως αντιδημοκρατικό αυτό. Ποιο είναι όμως αντιδημοκρατικό να έχουμε μια δημόσια ε, τηλεόραση ε, που ξεχνάει να αναφέρει ένα θέμα όπως είναι οι προμήθειες, οι πιστηριασμοί για τα φάρμακα. Αυτό δεν εμφανίζεται στο δικό του σε αυτόνομο κανάλι ή ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, το μεγαλύτερο που έζησε στην ε, Ισπανία, το ΣΕΡΕ, δεν αναφέρεται και αυτό στο ΤΕΒΕΤΡΙ. Αυτό δεν είναι αντιδημοκρατικό όπως και δεν, ε, όπως δεν, είναι, δεν είναι δημοκρατικό να μην βάζετε το μικρόφωνο μπροστά στην κυρία Εσταράς για να ακουστεί και αυτή. Επίσης, μιλάμε για το Κοινοβούλιο και για την Γερουσία. Εκεί έγινε ακρόαση, απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα με τεκμηρίωση και δεν υπήρξε καμία δευτερολογία, ήταν τόσο ικανοποιητικά τα στοιχεία. Αν υπάρχουν έγγραφα, αν υπάρχουν στοιχεία που έχουν κατατεθεί. Τα ίδια ή παρόμοια με αυτά που πήρατε. Χίλια ε, σελίδες λέτε αυτό το έγγραφο. Ναι, υπάρχουν σίγουρα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και έπρεπε να καταρριφθούν όλα τα επιχείρηματα ένα προς ένα. Γι' αυτό και ήταν τόσο ογκώδες αυτό το αρχείο. Πρέπει να τα διαβάσουμε όλα αυτά τα έγγραφα. Τα διαβάζουμε όμως αυτά τα έγγραφα δεν τα διαβάζουμε γιατί ουσιαστικά ε, πρόκειται για πολιτική κριτική, πολιτικό διαχωρισμό ε, και αυτό κάνει πάντα η αριστερά εδώ στο Κοινοβούλιο. Thank you very much. Thank you very much. Una cuestión de orden. Διαδικαστικό, Σεσίλια, λέει η κυρία Βαλή. Διαδικαστικό. Εγώ νομίζω ότι στην Επιτροπή αυτή δεν συνέβη ποτέ να έχουμε έλλειψη σεβασμού για τους αναφέροντες. Και εδώ έχουμε ακούσει ε, δύο και τρεις φορές αυτό για το μικρόφωνο. Ούτε εγώ είχα μικρόφωνο μπροστά μου, αλλά με μαγνητοσκοπούν, όπως και όλους και όλου τους άλλους. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι σωστό να λέτε κάτι το οποίο είναι λάθος, το οποίο είναι ψέμα και δεν είναι αλήθεια. Μας παίρνουν οι κάμερες και εμένα και εσάς και την Εσταράς και όλους. Επομένως, παρακαλώ, ε, μην ε, είστε άδικοι απέναντι ούτε στους αναφέροντες, ούτε απέναντι στην αλήθεια. Micro a Televisión Española la cámara para mí y el cámara ha dicho que a mí no me lo ponía. Y tenemos allí la chica que lo ha pedido. Εγώ ζήτησα, ε, δεν μου δώσανε το μικρόφωνο, αλλά στην κυρία με τα κόκκινα τη το δώσανε. Δεν σου έδωσα ε, τον λόγο Ρώσα, λέει πρόεδρο. Ε, να έχουμε λίγη τάξη εδώ πέρα, παρακαλώ. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερο. Άρα τι κάνουμε, ζητάμε το λόγο, μας δίνεται ο λόγος και μετά μιλάμε. Όχι έτσι, ξαφνικά και χωρίς να μας έχει δοθεί ο λόγος. Αυτή είναι η διαδικασία που ισχύει σε όλες τις επιτροπές και σε αυτήν και στις άλλες. Ο κύριος Μαρινίου Ελπίντο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ δεν υπάρχει πορτογαλική διερμηνία. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στην ε, γλώσσα που είναι αναγνωρισμένη ως πορτουνιόλ, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν κάπως να μεταφραστούν τα ισπανοπορτογαλικά που θα μιλήσω. Εδώ είμαι εδώ ως Πορτογάλος για τους ίδιους λόγους ε, που η Πορτογαλία στηρίζει τις ε, καταγγελίες, ε, τα αιτήματα των Πορτογάλων δημοσιογράφων και τις αναφορές σχετικές που ασκούν κριτική στα δημόσια μέσα ενημέρωσης για έλλειψη πλουραλισμού. Ήρθα εδώ γιατί όταν δημοσιογράφοι, επαγγελματίε λένε ότι δεν είναι εγγυημένος ο πλουραλισμός, αυτό δεν είναι πρόβλημα της δημοσιογραφίας, αλλά της δημοκρατίας. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρόβλημα. Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Γι' αυτό αγωνίζομαι για την ελευθερία τύπου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον η ε, Επιτροπή Αναφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το ερευνήσει το θέμα. Γιατί η ελευθεροτυπία είναι ουσιώδης προϋπόθεση της δημοκρατίας. Δημοκρατία χωρίς ελευθερία τύπου, χωρίς πλουραλισμό, χωρίς σεβασμό για την ε, ε, πολυμορφία της γνώμης δεν γίνεται στην κοινωνία. Εγώ ήρθα εδώ για να στηρίσω τα δικαιώματα των δημοσιογράφων όχι συνδικαλιστικά, γιατί εδώ μιλάμε για τη δημοκρατία. Ε, δημοκρατία αυτά είναι εχέγγυα για την κοινωνία. Πρέπει να σέβεται ε, τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης. Γι' αυτό ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί στη σχετική έρευνα για να ε, δει κατά πόσο αναλυθεύουν ή όχι αυτά τα όσα καταγγέλουν οι αναφέροντες. Αν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νύπτει τα οσα καταγγελουν η αναφερονται αν τωρα η ευρωπαικη επιτροπη νυπτει τα σχηρα της και λέει ότι δεν θέλει, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη σχετική αρμοδιότητα και μπορεί να το προχωρήσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπενίτο Ζιλουάγκα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και γιατί ε, μας δίνετε το λόγο στην Επιτροπή Αναφορών. Αν και δεν είμαστε λίγο, θέλω να στηρίξω το, από πλευρά του Ποδέμος τους αναφέροντες και την αναφορά τους. Αυτό ε, που με διαφοροποιεί τη φωτό από τη θέση της Κομισιόν. Η Κομισιόν που φαίνεται ότι τις αρμοδιότητές της ε, αντιλαμβάνεται ανάλογα με το θέμα. Το θέμα εδώ είναι η εγγύηση της ε, ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού των μέσων ε, δημόσιας ε, ενημέρωσης. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Είναι θεματοφύλακας των θεμελιωδών δικαιωμάτων η Κομισιόν, άρα έπρεπε να μπορεί αυτά τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, να τα προστατεύσει και θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον να τα προστατεύσει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και αυτό θέλω να στήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εκπονηθεί μια έκθεση με τα στοιχεία που έδωσαν οι αναφέροντες και τα οποία μας έπρεπε Και θέλω να ζητηθούν άμεσα εξηγήσεις στην Ισπανική κυβέρνηση. Βέβαια σας προειδοποιώ ότι ο Υπουργός μάλλον θα σας πει αλλάξτε κανάλι. Το έχει πει κάποιος ε, σε ένα κοινοβουλευτικό έδρανο που υποτίθεται ότι ήταν και υπουργός το Λαϊκό Κόμμα αυτό κάνει. Δεν του αρέσει ο πλουραλισμός, δεν του αρέσει να ακούει κριτικές, του αρέσει μόνο στα χαρτιά ο πλουραλισμός. Είναι λυπηρό που έχουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, αυτά τα θέματα εδώ στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ξεχνάτε ε, σε όλες αυτές τις πληροφορίες ε, πόσες ε, παρετήσεις επαγγελματιών έγιναν που δεν ήθελαν να ποσιοποιήσουν ειδήσει για σκάνδαλα, για τις υποκλοπές της κυβέρνησης και σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση, μάλλον την ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής κυβέρνησης δεν συμμετέχουν στη λογοκρισία επαγγελματίε και τι κάνουν, ε, τους μεταφέρουν σε άλλη θέση οι προϊστάμενοι τους. Ε, τελικά γιατί γίνεται λόγος εδώ, για τη δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια, ε, τηλεόραση πρέπει να είναι δημόσια και όταν έχουμε ένα δημόσιο κανάλι περιμένουμε αντικειμενική πληροφόρηση και όχι πολιτική επιχειρηματολογία του κόμματο, τη κυβέρνηση στην περίπτωση. Ευχαριστώ. Έχουμε σχεδόν τελειώσει τον κατάλογο. Απομένει ένα ομιλητή μόνο και επειδή είναι Σουηδέζα ξέρω ότι θα είναι απολύτω ακριβής. Κυρία Βαλέρο. Θα μιλήσω όμως στα Ισπανικά και δεν είμαι Ισπανίδα. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Ε, φαίνεται όμως ότι γίνεται μια ισπανο-ισπανική συζήτηση εδώ, μια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Ισπανίας. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία έκφρασης και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την περίπτωση της Ισπανίας βέβαια. Και ακριβώς για αυτό το λόγο θεωρώ περίεργο αυτό που λέει Κομισιόν. Ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε εδώ να το συζητήσουμε, δεν μπορεί να μας απασχολήσει, αλλά μιλάμε για τις θεμελιώδεις μας αξίες Μιλάμε για αυτό που υπόθηκε ήδη εδώ, ότι δηλαδή η ελευθεροτυπία είναι θεμελιώδες, αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας, μιας δημοκρατία που λειτουργεί. Και εμείς ως βουλευτές ε, είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τον πλουραλισμό αυτόν. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτή την εσωτερική σπανισπανική συζήτηση μόνο. Άκουσα τους αναφέροντες δεν νομίζω ότι για το τίποτα ντύνονται στα μαύρα ε, στην οθόνη τη τηλεόραση κάθε Παρασκευή. Αν το κάνουν αυτό, αν διαδηλώνουν κατά αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι είναι σοβαρή η κατάσταση. Εμείς λοιπόν πρέπει να τους ακούσουμε και να διερωτηθούμε γιατί, γιατί το κάνουν αυτό οι δημοσιογράφοι, γιατί διαδηλώνουν, γιατί διαμαρτύρονται. Διότι δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω ε, για το θέμα αυτό, γιατί δεν είμαι μέλος ε, τώρα τη επιτροπή Αναφορών, όμως, όπως και πολλοί άλλοι, εδώ θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, γιατί ναι, πράγματι πρέπει να ακούμε τους αναφερόντε αλλά να μην περιοριζόμαστε και σε αυτή την ισπανισπανική συζήτηση. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτονόητο ότι διαδικαστικό, κυρία Μιράντα. Ναι, διαδικαστικό. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας θέλω να αναφερθώ για τις συμπεριφορισμένων μιλών ε, του ΕΛΚΑ. Πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμό απέναντι στου αναφέροντε. Ε, ξέρω τι θα πει, κάνω προεκλογική εκστρατεία. Αυτό σημαίνει δεν σέβομαι του αναφέροντε. Γιατί αυτό ο κύριο ε, που ε, έχει την κάμερα εδώ δεν ήρθε με του αναφέροντε, αλλά γιατί οι αναφέροντε ενημέρωσαν τον τύπο καθώ και του βουλευτέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε ότι είχαμε αυτή τη συνάντηση εδώ. Παρακαλώ, λιγάκι σεβασμό. Όχι μόνο για του αναφέροντε, αλλά και για κάποιου από εμά που έχουμε ψηφιστεί ε, και ε, όχι ε, σαν, και, ψηφίζουμε αυτά που θέλουμε και όχι αυτά που σας πασάρουν εσάς και ψηφίζετε ό,τι σας έχουν πει. Ακόμη περισσότερα διακυβεύονται. Ξέρετε, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανά σε όλη την Ευρώπη και να βλέπουν ξαφνικά ανθρώπους να φωνασκούν, να ορλιάζουν ένα στον άλλο σαν απολύτιστοι. Είναι το χειρότερο πρόσωπο που θα μπορούσε να δείξει το κοινοβούλιο. Αυτό ισχύει για όλους. για όσους φώναξαν, για όσους ύψουσαν τη φωνή, για αυτούς τα λέω. Να σας πω ότι έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεστε ούτε να διακόπτετε την πρόεδρο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, θα ήθελα να στραφώ στους αναφέροντες και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους όλων όσοι ένα διαδικαστικό πρόεδρε Διαδικαστικό πρόεδρε, Θα σας δώσω το λόγο όταν θέλω. Θα σας δώσω το λόγο σε ένα λεπτό εφόσον είναι διαδικαστικό. Και ζητώ συγγνώμη για όσους ε, δεν ε, έδρασαν ως πολιτισμένα μέλη αυτού του κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Για το σεβασμό για την κυρία Μιράντα χρησιμοποιεί λέξεις όπως λογοκρισία, χειραγώγηση απέναντι ε, στην πολιτική ομάδα που εκπροσωπώ. Και ζητώ σεβασμό. Σεβασμό και εγώ, γιατί αυτό απαιτεί και η συμμετοχή μας σε αυτή την Επιτροπή. Αυτό που λέω είναι ότι η Επιτροπή της οποίας την χάνω πρόεδρος δεν είναι παιδική χαρά για ενήλικες που έχουν εκλεγεί εδώ στο Κοινοβούλιο να να φωνάζουν, να τον λόγο χωρίς να τους τον δίνει κανένας. Αυτό ισχύει σε άλλα κοινοβουλία, όχι σε αυτό εδώ. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά στρέφομαι ξανά προ του αναφέροντε και έχετε τον λόγο για επιπλέον δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αλεχάνδρο Καμπαγέρο δε λέγομαι. Είμαι ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Συντακτών Ειδήσεων. Εξελέγει ε, σε δημοκρατικέ εκλογέ από του συναδέλφου μου. Δεν εκπροσωπώ κανένα κόμμα, αλλά μόνο του επαγγελματίου συναδέλφου μου από την Ισπανική τηλεόραση, όπου υπάρχουν και αριστεροί και δεξιοί και κεντρώοι όπως είναι προφανές, επομένως ε, θέλω να πω ότι ε, ως φορέας ε, δεν έχουμε κανένα κομματικό χαρακτήρα. Καταρχάς θα ήθελα να επενθυμίσω κάτι που έγινε το Δεκέμβριο του 2015. Είχαμε μια αποστολή της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη που εξέδωσε την τελική έκθεση αξιολόγηση των εκλογών στην Ισπανία και μεταξύ των συστάσεων τους πριν δυόμιση χρόνια λέγανε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η μέθοδος για την επιλογή των ανώτατων στελεχών της Ισπανικής Ραδιοτηλεόρασης το λέγανε αυτό, γιατί έλεγαν ότι πρέπει να προστατευτεί η, από πολιτικές παρεμβάσεις ε, η δημόσια ραδιοτηλεόραση και για να διατηρηθούν τα πρότυπα και τα υψηλά στάνταρ. Και δυόμιση χρόνια μετά ο πρόεδρος ε, της εταιρείας, ε, ε, παραμένουν στη θέση τους, δεν έχουν αλλάξει. Τώρα, άκουσε η Επιτροπή σας την συντρόφισσα μίλησε για πέντε λεπτά περίπου φυσικά και δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως το θέμα. Έχουμε όμως πλήρη τεκμηρίωση. Έγγραφα τα οποία επισυνάπτουμε στην αναφορά μας και με τα έγγραφα αυτά νομίζω ε, ότι μπορείτε να το δείτε. Τα στείλαμε αυτά τα έγγραφα και στη διοίκηση τη Ισπανική Ραδιοτηλεόραση και εκεί τεκμηριώνουμε ότι πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή υπάρχει έλλειψη ανεξαρτησίας, έλλειψη πλουραλισμού και δεν υπάρχει ουδετερότητα στη δημόσια Ισπανική Ραδιοτηλεόραση. Τελευταία απόδειξη αυτό με το μικρόφωνο. Αν θέλετε πρώτα καταγγείλετε το Συμβούλιο, ε, όπως ε, εμείς ασχολούμαστε οποιαδήποτε άλλη καταγγελία, έτσι θα ασχοληθούμε και με αυτή την καταγγελία κατά πόσον ε, δηλαδή υπήρξε κακοδιαχείριση, εμείς θα το παραδεχθούμε. Αν βέβαια δεν υπήρξε, δεν υπήρξε. Και ολοκληρώνω. Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελμών στον ε, κλάδο της πληροφόρησης, που επαναλαμβάνει το αριστερό το δεξί, όλοι είναι, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε από το Συμβούλιο των Συντακτών ε, Δελτίου Ειδήσεων, θέλουμε να είμαστε ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα πλουραλισμού αντικειμενικότητας ε, στην Ισπανία για όλους. Ε, θέλουμε όλοι οι πολίτες να μας αντιμετωπίσουν όπως και αν σκέπτονται, αλλά να νιώθουν και υπερήφανοι για τη δημοσία ραδιοτηλεόραση. Και αυτό, συγγνώμη, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε εργαζόμαστε για να τους υπηρετήσουμε. Για να υπηρετήσουμε τους. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στην απόφαση που θα λάβετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι πάντα τόσο ταραγμένη αυτή η Επιτροπή όπως σήμερα. Ήταν πολύ συναισθηματική η συζήτηση από όλες τις πλευρές και από αριστερά και από δεξιά και από παντού. Ζητώ συγγνώμη για την κακή συμπεριφορά που είδαμε σήμερα. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι Αυτά που είδατε εδώ απλά αποδεικνύουν ότι η ελευθερία έκφρασης είναι σημαντικό ζήτημα. Αφορά τους πάντες αναξαρτήτως ε, ιδεολογίας ε, και πολιτικής τοποθέτηση. Θα προσπαθήσουμε τώρα να συνοψίσουμε αυτή την ε, αναφορά. Πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή. Ακούσαμε ευρία υποστήριξη γι' αυτό. Επίσης θα πρέπει να ε, στραφούμε στον εκπρόσωπο της Κομισιόν που μας έκανε ε, μια προφορική παρουσίαση ως απάντηση σήμερα. τι χρειαζόμαστε γραπτός. Αν μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε την απάντησή σας γραπτός, θα μας βοηθούσατε ιδιαίτερα. Ήδη έχουμε διαβιβάσει την αναφορά αυτή στην Επιτροπή ε, πολιτισμού και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών προς ενημέρωση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να εκφράσουμε σε μια επιστολή προς την Ισπανική κυβέρνηση την ανησυχία μας και να δούμε τι θα μας απαντήσουν, τι εξηγήσει θα δώσουν. Να μας εξηγήσουν πώς βλέπουν αυτή την κατάσταση, την τρέχουσα κατάσταση και τι προβλέπουν ότι θα γίνει βάσει της αναφοράς που έχουμε λάβει. Ναι, ωραία. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Καλή επιστροφή στην Ισπανία. Και όσοι σκοπεύετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα, παρακαλώ φύγετε πολύ γρήγορα γιατί απομένει μία αναφορά. Και θα... δεν θα ήταν πολύ ευγενικό να αφήσουμε τον αναφέροντα να περιμένει πολύ ώρα. Πρόκειται για την αναφορά 1074, 1074 για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε υποστηρικτέ ναζιστικών εκδηλώσεων και φασιστικών ιδεοδών. Κάνουμε ένα διάλειμμα 30 δευτερολέπτων. Μπορούμε να συνεχίσουμε νομίζω όσο το δυνατόν ταχύτερα με την επόμενη αναφορά. Σημείο 20. Ο αναφέρον είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κούζινς. Σας δίνω το λόγο και να παρακαλέσω τους συναδέλφους και τους λοιπούς να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο ήσυχα. Please go ahead. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, Γιάννης Κούζινς ονομάζομαι. Είμαι επικεφαλής της Ένωσης κατά του Ναζισμού της Λετωνίας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω εδώ σήμερα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις σε υποστηρικτές ναζιστικών εκδηλώσεων και φασιστικών ιδεοδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει έναν κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων επί των οποίων θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσει, διότι υποστηρίζουν ναζιστικές εκδηλώσεις και πρεσβεύουν φασιστικά ιδεώδη. και νομίζω ότι θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοοικονομική υποστήριξη που δίδεται σε αρχές οι οποίες υποδαβλίζουν τέτοια φαινόμενα. Γνωρίζουμε τον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε άλλες χώρες, βλέπουμε τη Βόρειο Κορέα, βλέπουμε το Ιράν, βλέπουμε την τρομοκρατική οργάνωση ISIS στον κατάλογο αυτό συμπεριλαμβάνονται φορείς της ε, Κρυμαίας, ε, βλέπουμε άλλους οι οποίοι δρούν στο Αφγανιστάν και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το ιδεώδες της δημοκρατίας. Προωθεί τα όσα είπε ο Σούμαν για μια ενωμένη Ευρώπη. Ποιος είναι λοιπόν ο εχθρός εδώ. Στον κατάλογο αυτό των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πάντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον θεωρεί πάντα ότι ο εχθρός βρίσκεται εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν εχθροί της Ένωσης στο εσωτερικό της Ένωσης. Για παράδειγμα στις βαλτικές χώρες βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν υπουργοί ή ακόμα και μέλη της κυβέρνησης που ε, τρέφουν ε, εξτρεμιστικές νοοτροπίες και ιδεώδη. Βλέπουμε σε άλλες χώρες όπως η Ουγγαρία πως προωθούνται τάσεις οι οποίες είναι λαϊκιστικές ή πολλές φορές ακόμα και ναζιστικές Νομίζω λοιπόν ότι ε, ο κατάλογος αυτός των χρηματοπιστωτικών κυρώσεων δεν θα πρέπει να αφορά μόνο χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπως η Βόρειος Κορέα για παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανθρώπους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν εξτρεμισμό και τρομοκρατία και αναφέρομαι εδώ πέρα βέβαια και σε χώρες γειτονικέ της Ευρώπης, γειτονικέ Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ουκρανία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αναφοράς σας καλώ να ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δείτε τι μπορεί να γίνει. Βλέπετε πως έχει σήμερα η κατάσταση. Αντί να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη, έχουμε φαινόμενα όπως το Brexit, έχουμε αναδυόμενες εθνικιστικές στάσεις ε, στην Ήπειρό μας και έχουμε αρχίσει να καταστρέφουμε τελικά την ενωμένη ενιαία Ευρώπη. Ενώ αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τελικά είναι μια ενιαία Ευρώπη με μια κοινή προσέγγιση επιδημοκρατίας και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι μπορούμε να κινηθούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο που να περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εκπροσωπείτε εδώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερσάτ Πικιουέρας παρακαλώ. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είχαμε το χρόνο να σας αποστείλουμε γραπτή απάντηση. Θα προσπαθήσω πάντως να εξηγήσω εν συντομία Ποια είναι η απάντηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ευχαριστήσω καταρχά τον Αφέροντα και να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βαθιά προσιλωμένη στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού, του εθνικισμού, της μυσαλλοδοξίας, γενικότερα των τάσεων αυτών που στρέφονται κατά των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντείνει την αντίδρασή της στα φαινόμενα αυτά. Έχουμε την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου να καταπολεμήσουμε εκφράσεις εξτρεμιστικές, ρητορική, ξενοφοβική και είμαστε σε θέση επίσης μέσω της κοινοτικής νομοθεσίας να καταπολεμήσουμε τη ρητορική μίσους που βασίζεται στο φύλλο, στην διαφορετική φιλετική καταγωγή, την ε, διαφορετικές θρησκευτικέ ε, πεπιθήσεις ε, και το καθεξής. Και ξέρετε ότι πέρα από το κοινοτικό δίκαιο έχουμε και το εθνικό ποινικό δίκαιο που ποινικοποιεί τις πράξεις αυτές. Έχουμε επίσης νομοθεσία και σε εθνικό επίπεδο που στρέφονται κατά της άρνησης της γενοκτονίας του ολοκαυτώματος και εθνικές νομοθεσίες οι οποίες στρέφονται και οι ίδιες κατά της ρητορικής μίσους. Και επίσης καταδικάζουμε και ποινικοποιούμε την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλου έντυπου υλικού προκειμένου να προωθηθούν εξτρεμιστικές, ξενοφοβικές, ακραίες τάσεις. Εναπόκειται πάντως στο εθνικό δίκαιο και στις εθνικές αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν και να διώξουν τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο νοσιακό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο έχει διμερείς επαφές με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει ότι έχουμε τη μεταφορά της ε, σχετικής κοινοτική ε, νομοθεσίας. Παρακολουθούμε όμως και την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και έχουμε και ομάδες εργασίας προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και γι' αυτό το λόγο έχουμε και την ομάδα υψηλού επίπεδου κατά της ξενοφοβίας όπου πέρα από τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ο αλλά και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Στα πλαίσια της εφαρμογής νομοθεσίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί δράσεις κατά της ρητορικής μίσους και κατά των ακραίων αυτών τάσεων που καταγγέλει ο αναφέρον. Προσπαθούμε μέσω της χρηματοδότησης εθνικών προγραμμάτων να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά και αυτό ισχύει επίσης και για κάποια προγράμματα μέσω διαδικτύου. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα συμπεριλαμβανομένου και του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Το 2016 Έχουμε επίσης και την δημοσίευση ενό κώδικα δεοντολογίας όπου ουσιαστικά προσπαθούμε μέσω του διαδικτύου και για τις διαδικτυακές πλατφόρμες για μέση κοινωνική δικτύωση όπως ε, το Facebook, το Twitter κτλ. να υπάρχει μια κοινή συμφωνία για την καταπολέμηση τη ρητορική μίσου. Και επίσης έχουμε την 23η Αυγούστου όπου κάθε χρόνο έχουμε την ημέρα αυτή μνήμης και έχουμε και προγράμματα υπέρ των πολιτών με 3,5 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καταπολεμήσουμε εγκληματικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα λοιπόν από τις οικονομικές κυρώσεις έχουμε και ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους. Δεν μπορούμε να δώσουμε όμως συνέχεια στην αφορά αυτή γιατί όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα ουσιαστικά υπερβαίνουν τις ε, οικονομικές κυρώσεις. Σας ευχαριστώ. Very much. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητροφάνοφ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Κούζενς, ο αναφέρον, δεν είναι μέλος του κομματός μου παρότι συμπατριώτης μου, οπότε δεν έχω καμία υποχρέωση να τον στηρίξω. συζητήσαμε όμως πριν δύο χρόνια. Αν είχαμε συζητήσει συγγνώμη, πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσα να είχα υποστηρίξει αυτή την αναφορά, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η κατάσταση στη χώρα μου, στη Λετωνία, άλλαξε. Επιδεινώθηκε. Και έτσι έχω αλλάξει άποψη. Και θέλω να υποστηρίξω στεναρά αυτή την αναφορά γιατί διότι η σχετική ιδεολογία έχει ενισχυθεί, η νεοναζιστική ιδεολογία έχει φύγει από το πολιτικό σύστημα, από τα περιθώρια του πολιτικού συστήματος και έχει γίνει, έχει γίνει mainstream. Για πολλές δεκαετίες ε, οι ακροδεξιοί οργάνωναν πορείες στο κέντρο της Ρήγας, της πρωτεύουσα της Λετωνίας, για να γιορτάσουν τους πρώην στρατιώτες ΕΣΕΣ της Λετωνίας. Φέτος οι ακροδεξιοί ε, βουλευτές ε, στο Κοινοβούλιο πρότειναν να, να γίνει ε, να υπάρξει μια μέρα εορτασμού αυτών των στρατιωτών. Ονομάζονται Εθνική Συμμαχία και είναι κομμάτι του κυβερνοντός κόμματος. Δεν υιοθετήθηκε το σχέδιο αυτό. Και έτσι δεν έγινε αυτή η μέρα γιορτή αργία, αλλά μόνο λόγω της πίσης των εξωτερικών συμμάχων και της διεθνούς κοινότητας. Δεν βλέπω όμως εσωτερικά να υπάρχουν εμπόδια για τέτοιες αλλαγές ε, της πολιτικής. Ε, αφορά κάποια ζητήματα... Ε, έχουμε μία στροφή προς τα δεξιά στην Λετωνία. Υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο ένα ψήφισμα ώστε να προωθηθεί το αίτημα ε, να υπερασπιστούμε τους ε, ρωσόφωνους, ε, να καταλήψουν οι ρωσόφωνοι που δεν αναγνωρίζουν τη Λετωνία. Νομίζω ότι εδώ έχουμε εθνικιστική συμπεριφορά. προσπαθούν να οθήσουν ε, τη ρωσική μειονότητα να εγκαταλείψει τη χώρα, καταστρέφοντας το σύστημα εκπαίδευσης σε μειονοτικές γλώσσες. Μετά από 200 χρόνια ανάπτυξη των ρωσικών σχολείων στη χώρα μας, τα σχολεία αυτά θα πρέπει να καταστραφούν αντικαθιστώντας τη γλώσσα σε μόνο λετονικά. Το επόμενο βήμα θα είναι το σχέδιο απαγόρευσης χρήσης της ρωσικής γλώσσας και άλλων μειονοτικών γλωσσών ε, στην προεκλογική εκστρατεία Κάτι άλλο που συζητείται επίση στο, στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι η απαγόρευση των τηλεοπτικών σταθμών ε, ρωσική γλώσσα. Το επόμενο βήμα θα είναι, ήταν η σύλληψη δύο ακτιβιστών εκπροσώπων τη ρωσική κοινότητα. Για ασαφεί λόγου. Τώρα το κόμμα μου διώκεται ποινικά για την οργάνωση ειρηνικών διαδηλώσεων κατά της διαγραφής της μειονοτικής εκπαίδευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε συνάδελφο που κάθε μέρα φοβάται ότι θα τη συλλάβει η αστυνομία λόγω μια συνάντηση που έκανε το κόμμα μα πριν από μερικέ εβδομάδε. Δεν είναι υπερβολικό να πει κανεί ότι στη Λετωνία οι ριζοσπαστικοί νεοναζί έχουν έρθει στην εξουσία. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να υποστηρίξει την αναφορά να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις σε υποστηρικτές ναζιστικών ιδεοδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευτυχώς είναι μικρή ο κατάλογο των ομιλητών. Σας δίνω δηλαδή περισσότερο χρόνο από όσο θα είχατε κανονικά και μπορείτε να υπερβείτε και λίγο το πεδίο εφαρμογή, το, πεδίο, το αντικείμενο αυτής τη αναφοράς. Κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Σεσίλια. Θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα πρώτα απ' όλα, διότι πράγματι αυτό είναι ανησυχητικό. Η ιδεολογία, η νεοναζιστική ιδεολογία είναι κάτι που το βλέπουμε στις διάφορες χώρες της Ένωσης και στις εκλογές ε, που προκύρουν στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε να αυξάνει η δύναμη της άκρας δεξιάς και να συγκεντρώνει ψήφους. Εδώ χαιρόμαστε για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιορτάζουμε ε, τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα βλέπουμε να ανεβαίνει η ακροδεξιά και τελικά οι αντιευρωπαϊκές ε, τάσεις αρχίζουν να παίρνουν το πάνω χέρι. Μπορεί δηλαδή να αρχίσει να επικρατεί εκ νέου ε, αυτή η ιδεολογία. Υπάρχει κίνδυνος, είναι εδώ η απειλή. Αν δεν το βλέπουμε σημαίνει ότι είμαστε κοντόθωροι, δεν μας αρέσει να διαβάζουμε ιστορία. Δεν ξέρω, πολύ χαλαρά τα αντιμετωπίζουμε με αυτό το θέμα και πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτρέπει σε ομάδες όπως είναι οι Έλληνες Ναζί της Χρυσής Αυγής ή την ομάδα της Λεπέν να είναι εδώ. Διότι κάποιες φορές ακούσουν ολομέλεια πράγματα που πραγματικά ε, είναι να τους βάλεις είτε ζουρλομανδία είτε χειροπέδες. Και αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε και να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, ε, να μην επαναλάβουμε σφάλματα του παρελθόντος. Ακούστε, υπάρχουν πράγματα που κάνουν οι κυβερνήσεις και είναι κρίμα που έφυγαν όλοι οι Ισπανοί που ήταν εδώ πριν. Στην Ισπανία έχουμε αυτό το νόμο για τη φήμος του τι, το έχουμε καταδικάσει, μπαίνουν ε, μέχρι και τραγουδιστές στη φυλακή, τέλος πάντων επιβάλλονται πρόστιμα και άλλοι καλλιτέχνες. Και η κυβέρνηση επιδοτεί την Ένωση Φρανθίσκο Φράνκο. Παίρνει συμβάσεις αυτή η Ένωση. Και πέραν των ετήσιων επιδοτήσεων ε, επιδοτούνται ε, και κάποιες ενώσεις στρατιωτικών υπέρ του Φράγκου. Άρα μπαίνουμε σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και είναι κρίμα. Όλοι αυτοί και όλες αυτές που τόσο υπερασπίζονταν ε, την ε, έκφραση, την ελευθερία της έκφρασης, ε, να έχουν φύγει τώρα και να μην καταφέρονται εναντίον αυτού του νόμου στην Ισπανία. Ε, ενώ κάποιοι άνθρωποι ε, για ε, μία μπλούζα, για μία ζωγραφιά πάνε φυλακή και εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα. Επίσης περιχαρακώνονται όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί μέχρι και επιδοτήσεις παίρνουν και δεν κουνάνε ρούπι. Ευχαριστώ. πετεριά. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας ουσιαστικά από αυτή την αναφορά. Η άποψή μου είναι σαφής ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα κράτα, κράτη-μέλη. Και κατά τη δική μου άποψη θα ήταν λάθος δρόμος να υπάρξει απαγόρευση από τις Βρυξέλλες γιατί τότε θα αυξηθούν αυτά τα ρεύματα τα λαϊκίστα και τα ακροδεξιά. Σίγουρα υπάρχουν τελείως διαφορετικές αιτίε για το τι γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα. Ε, ουσιαστικά είναι παιδιά προβληματικά ή ε, άλλοι ε, λόγοι. Σίγουρα είναι και η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του συναθρίζεστε που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, και δεν ξέρω ε, τι επιπτώσεις θα είχε η απαγόρευση. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει προς λάθος κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Νομίζω επαρκώς μας τα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ περιορίζομαι στην αναφορά εδώ, γιατί μπορούμε να κάνουμε ολόκληρο σεμινάριο. Ε, για τους ε, εθνικιστές και τους ακροδεξιούς κτλ. Για την αναφορά συγκεκριμένα λοιπόν, νομίζω ότι αυτά που είπε η Κομισιόν είναι επαρκή. Αν υπάρχει πρόβλημα εφαρμογή στα κράτη-μέλη, πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, ε, αν θα κλείσουμε την αναφορά, αν θα απαντήσουμε γραπτός ή αν θα το συζητήσουμε τα των Δεν ξέρω. Απλά το είδαμε το θέμα και το πιάσαμε πάρα πολύ έτσι ε, ευρέως και το συζητήσαμε πολύ πιο ανοιχτά σε σχέση με το πεδίο, το περιορισμένο της, της ε, αναφοράς. Ευχαριστώ κύριο Στερή Κάμπρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να αποτίσω φόρο τιμής στην συμμαχία αυτή μεταξύ, των Μύρος, μεταξύ του Μύροσλαφ και των αναφερόντων, ότι ανήκουν σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα, ουσιαστικά ενώνονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των αναφορών και όλων αυτών των ανησυχιών που εκφράζονται. Εντελώ διαφορετική εικόνα που μας δώσανε από εμά τους Ισπανούς, οι οποίοι διαιρεθήκαμε μεταξύ μόνο και μόνο επειδή ανήκουμε σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα και ξαφνικά όλοι οι Ισπανοί συνάδελφοι εξαφανίστηκαν γιατί από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρονται μόνο για τα ισπανικά ζητήματα και όχι για άλλα ζητήματα και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Ξέρετε ότι εγώ είμαι Ισπανός, μάλλον είμαι από την ε, Ισπανία αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου Ισπανό τελικά. Λοιπόν, Θεωρώ ότι οι φασιστές και οι νεοναζιστές είναι πραγματικά στοιχεία πολύ επικίνδυνα, αυτό το γνωρίζουμε. Βλέπουμε επίσης ότι αυξάνονται οι ακροδεξιές τάσεις στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο συνάδελφός μου αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του με τους αναφέροντες στα πλαίσια αυτής αναφοράς. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. και θα έπρεπε μάλιστα να στείλουμε και μια επιστολή στις αρχές της χώρας, της Λετωνίας, ζητώντας δύο πράγματα. Πρώτον, μία περιγραφή και έπειτα μία εξήγηση των όσων αναφέρει ο Μύροσλαφ και οι αναφέροντες. Δηλαδή ποια είναι η αντίδρασή τους, πώς βλέπουν αυτή τα πράγματα βλέπουν και αυτοί τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία, έχουν την ίδια άποψη, ενδεχομένω να πρεσβεύουν ε, διαφορετικά πράγματα. Θα ήταν πάντω πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τελικά ποια είναι η άποψη των λειτουργικών αρχών και αν υπάρχει διάσταση απόψεων. Λοιπόν, πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα ξεκαθαρίζαμε και κάπως την κατάσταση. Σε μια εποχή λοιπόν αναδυόμενου φασισμού και ναζισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν εξηγήσει και να δίδονται σαφηνήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλύψαμε κάθε πιθανή πτυχή του ζητήματος αυτού. Νομίζω ότι όλα τα είπαμε, όλα τα καλύψαμε. Κύριε Κούζενς, λοιπόν, έχετε πάλι το λόγο εφόσον θέλετε να μιλήσετε για ακόμα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη πιστεύω δεν κάνουν αρκετά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι γνωρίζετε τις ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ευρώπη και οργανισμούς όπως η UEFA, όπου εγώ είμαι παρατηρητής. Που όταν βλέπουμε κάποιες σημαίες στα στάδια, στα γήπεδα, γράφουν πάνω SS ε, ή κάτι τέτοιο, τέτοιου είδους ε, σημαίες, θα έπρεπε να επιβάλλουμε οικονομικές κυρώσεις στην ομάδα, όχι στους οπαδούς, στην ομάδα. Οι υπουργοί μας λοιπόν έτσι κάνουμε στα γήπεδα. Ε, το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και στη χώρα μας όταν έχουμε υπουργού βουλευτές ε, που πηγαίνουν σε ναζιστικές πορείες. Ε, και στην Πολωνία καταστρέφουν μνημεία και σε άλλες χώρες. Στην Ουγγαρία το βλέπουμε στη Δρέζη, στη Γερμανία. Ένα σωρό πράγματα. Αν κάνουμε λοιπόν αυτό που κάνει η UEFA, επιβάλλουμε οικονομικές κυρώσεις, όταν βλέπουμε τώρα σημαίες με SS, στέλνουμε μια επιστολή, άμα το δούμε λοιπόν να την κρατάει κάποιος υπουργό, να πάμε να στείλουμε μια επιστολή. Γιατί κρατάει τέτοιο πράγμα, κατά τέτοια σημαία ένας υπουργός και λέτε εγκληματίες, αλλά αυτοί είναι κυβερνήσεις. Ε, δεν είναι ε, υπόκειται σε νόμους όπως οι πολίτες. Στο κοινοβούλιο δεν ισχύουν τέτοια. Είναι διαφορετικό, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μέχρι τις Βρυξέλλες σήμερα. Ελπίζω να έχετε καλή επιστροφή. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα να το κλείνουμε. Λοιπόν, λέω να την κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, συμφωνείτε, και να ζητήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει μια γραπτή ενημέρωση, απάντηση, ώστε να ξέρουμε κι εμείς ε, ποιο θα είναι το επόμενο μας βήμα. Θα ήθελα επίσης να στείλουμε μια επιστολή στη λετονική κυβέρνηση για να τους ενημερώσουμε για την ύπαρξη της αναφοράς και να τους ε, ζητήσουμε να μας πούν τις απόψεις τους επί του θέματος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Πηγαίνετε στα γραφεία σας. Να είστε ευγενικοί με όλους. Τελειώνουμε 10 λεπτά νωρίτερα. Καλό σας βράδυ. Παρά τη δύσκολη μέρα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.